So, dear colleague, so, and ladies Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, έχει πάει δυόμιση. We have now, um, Ξεκινάμε λοιπόν. Έχουμε την πρώτη δημόσια ακρόαση για το Brexit και τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις. Όπως πάντα, η ακρόαση αυτή είναι ιδιαίτερος επίκαιρη, διότι πριν από δύο ημέρες είχαμε μια καταρχήν συμφωνία για τη μεταβατική περίοδο μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό βεβαίως μας προσφέρει μια σαφή προοπτική για να ξεκινήσει όλος προβληματισμός για το τι θα πρέπει να συμβεί ε, και τι θα συμβεί στη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου και τι θα γίνει και μετά το 2020, πώς ε, θα διαμορφωθούν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Χαίρομαι λοιπόν που μοιράζομαι αυτή την πολύ σημαντική ακρόαση εδώ μαζί σας. Θα έχουμε αρκετό χρόνο σε σχέση με άλλες ακροάσεις και άλλα εργαστήρια σχετικά μέχρι τις 5. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι μπορούν να μιλήσουν όση ώρα θέλουν. Μας περιορίζει και κάπως ο χρόνος. Έχουμε δύο πάνελ και δύο σημεία το ένα είναι ο αντίκτυπος ε, της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Ηνωμένου Βασιλείου, να δούμε λίγο πώς έχει κατάσταση και πού βρίσκονται τα προβλήματα. Και δεύτερον, πώς ε, θα πρέπει να δράσουμε κατά τη μεταβατική περίοδο. Και το δεύτερο πάνελ αφορά τις μελλοντικές σχέσεις ε, και περιλαμβάνει ιδίως ε, το ε, τελωνιακό καθεστώς. Έχουμε πολλούς γνωσμένους κύρους εμπειρογνώμονες και θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω με το πρώτο τμήμα του πρώτου πάνελ, το θέμα του αντίκτυπου για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα δώσω καταρχάς το λόγο στη Μπάρμπαρα Μπάρσμα, που είναι καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Και θα μας ε, πει κάποια πράγματα για τον αντίκτυπο του Brexit. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στη δημοκρατική καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σας μιλήσω για τον αντίκτυπο του Brexit. Δεν είμαι απλώς ε, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, είμαι και διευθύντρια ε, διαχείρισης γνώσεων και στη Rabobank. Βλέπετε και το λογότυπο της Rabobank και θα αναφερθώ και σε μελέτες ε, τις οποίες έκανα στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ αλλά και στη Rabobank. Βάσει ε, μιας ε, πολύ διεξοδικής ανάλυσης που κάναμε, πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ απεσιόδοξη για τον αντίκτυπο του Brexit στην οικονομική ανάπτυξη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις κατοχώρες, αλλά κυρίως για το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Από οικονομική σκοπιά, όσο πιο ήπιο είναι το Brexit, τόσο καλύτερα. Και θα ξεκινήσω με μια παρατήρηση η ψηφοφορία για το Brexit και οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη ε, ε, ζημιώσει την ε, Βρετανική οικονομία. Η ετήσια ανάπτυξη επιβραδύνθηκε κατά 1,7% πέρσι, που είναι ο χαμηλότερος ρυθμός από το 2012 και περιμένουμε να μειωθεί η ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά μείον 1,4% και 1,1% το 2019. Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι Ποιε θα είναι οι μόνιμε αρνητικέ ε, συνέπειε για τη Βρετανική αλλά και για την ευρωπαϊκή οικονομία αυτή τη στιγμή υλοποιηθεί το Brexit. Υπάρχουν ε, αρκετοί διάβλοι μέσω του οποίου θα μπορούσε να πλήξει την Βρετανική και την Ευρωπαϊκή οικονομία το Brexit και ο πρώτος σημαντικός διάβλος από το οποίο θα μπορούσε να συμβεί είναι το εμπόριο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικός εταίρος ε, του Ηνωμένου Βασίλειου σε θέματα εμπορίου και για ε, Δασμού και αγαθά και μη δασμολογικά αγαθά, όπω για παράδειγμα τελωνιακή έλεγχη. Όλα αυτά αυξάνουν το κόστο του εμπορίου για τι ε, βρετανικέ εξαγωγέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιστρόφως. Και φυσικά οι υψηλότερες ε, πληθωρισμό εισαγωγών λόγω του αυξημένου κόστου του εμπορίου θα σημαίνει ότι θα υπάρχει και χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα για τα νοικοκυριά που θα χάσουν την αγοραστική του δύναμη. Επιπλέον, οι αγορές, το Ηνωμένο Βασίλειο αγοράζει ε, τα μισά από τα ενδιάμεσα προϊόντα του ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η αγορά των ενδιάμεσων προϊόντων θα γίνει πιο δαπανηρή λόγω των φραγμών στο εμπόριο, που σημαίνει ότι οι βρετανικέ επιχειρήσει θα αντιμετωπίσουν υψηλότερες τιμές εξαγωγών, επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας τους και μικρότερο μερίδιο της αγοράς. Επίσης, ελοχεύει ο κίνδυνο, το Ηνωμένο Βασίλειο να χάσει τη θέση του ως ε, είσοδος ε, προς την Ευρώπη και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Και αυτό είναι ο δεύτερος διάβλος μέσω του οποίου το Brexit θα μπορούσε να πλήξει τη Βρετανική οικονομία και είναι ε, η επιρροή στην παραγωγικότητα. Οι χαμηλότερε επενδύσεις θα έχουν αρνητικές συνέπειες για το κεφάλαιο που θα σταματήσει και την ε, ανάπτυξη της παραγωγικότητας και η παραγωγικότητα θα πληγεί με διάφορους τρόπους. Καταρχάς θα γίνονται χαμηλότερες επενδύσεις σε κεφάλαια. Ε, θα υπάρχει λικλότερη ε, ε, μεταλαμπάδευση γνώση από το εξωτερικό, θα υπάρχουν χαμηλότερες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη από ξένες επιχειρήσεις και το γεγονός ότι η οικονομία μετά το Brexit θα είναι λιγότερο ανοιχτή βαρύνει όχι μόνο τη δυνατότητα να μάθουν ε, από ξένες γνώσεις, αλλά μειώνει και τον ανταγωνισμό, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν και λιγότερα κίνητρα για καινοτομία και θα μειώσει και ε, τις ε, ε, διάφορες αποτελεσματικότητες. Θα οδηγήσει σε έλλειψη αποτελεσματικότητας. Οπότε έχουμε έξι πράγματα. Υψηλότερους φραγμούς, χαμηλότερες εξαγωγές, υψηλότερο πληθωρισμό, υψηλότερη ανεργία, χαμηλότερες ξένες άμεσες επενδύσεις και μικρότερη παραγωγικότητα. Θα περάσω τώρα κάποιες διαφάνειες. Δεν δουλεύει όμως. Να πάμε στην τρίτη διαφάνεια παρακαλώ. Αυτή θέλω. Λοιπόν, η χαμηλότερη παραγωγικότητα είναι αυτή που δημιουργεί προβλήματα ε, στα σενάρια που έχουμε. Έχουμε πολύ περισσότερες αρνητικές συνόπιες από τα περισσότερα ε, στοιχεία που έχουμε σε άλλες μελέτες που λαμβάνουν υπόψη και μοντέλα μακροοικονομικού επίπεδου, όπως ε, για παράδειγμα το μοντέλο Nigem που σας παρουσιάζω εδώ. Και γιατί συμβαίνει αυτό. Θα σας δώσω δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι εκτιμούμε όπως δεν γίνεται στις άλλες ε, ε μακροοικονομικές μελέτες, ένα μοναδικό παραγωγικό μοντέλο για το Ηνωμένο Βασίλειο που μας επιτρέψει να ε, εκτιμήσουμε καταλήλως τις αρνητικές συγκεκριμένε συνέπειες που θα προκαλέσει το Brexit για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο δεύτερος λόγος που έχουμε τόσο πολύ περισσότερα αρνητικά στοιχεία και προβλέψεις για τις συνέπειες του Brexit είναι ότι χρησιμοποιούμε μια βελτιωμένη δασμολογική εκδοχή του μακροοικονομετρικού μοντέλου που μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε καλύτερα τις αρνητικές συνέπειες ε, της, ε, του πληθωρισμού που θα προκύψει από το εμπόριο και θα θέσει φραγμού στο εμπόριο. Ευχαριστώ που με βοηθάτε με τις διαφάνειες. Τι κάναμε λοιπόν, εξετάσαμε τέσσερι εναλλακτικέ εκδοχές και τα συγκρίνουμε αυτό με την εναλλακτική λύση του παραμονή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε σκληρό Brexit που σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου θα διακοπούν και το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί εμπορική συμφωνία. Οι συμφωνίε του ΠΟΕ θα αποτελέσουν και τη βάση αυτού του ε, σκληρού Brexit και ε, υποθέτουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορέσει να αντιγράψει τα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του δασμού και τι ποσοστώσει το δεύτερο είναι ένα πιο ήπιο Brexit, έτσι θα συμμετέχει στην ενή αγορά του Ηνωμένου αλλά θα φύγει από την Τελωνιακή Ένωση και το κόστος του εμπορίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προκύπτει από τους μη δασμολογικούς φραγμούς. Και αυτό είναι το μοντέλο της Νορβηγίας. Ενδιαμέρω έχουμε συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που θα μπορέσουν να συμφωνήσουν ίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο για μια διμερή συμφωνία, αντίστοιχη με αυτή που έχουμε με την Ελβετία και ίσω και με τον Καναδά τώρα οι δασμοί αναμένεται να παραμείνουν μηδενικοί στα προϊόντα, αλλά θα αυξηθούν οι μη δασμολογικοί φραγμοί περισσότερο από το σενάριο του ήπιου Brexit. Οι υπηρεσίε πλέον δεν θα επιτρέπεται να παρέχονται ελεύθερα ε, για τους Βρετανούς. Και χρησιμοποιώντα ω βασικό σενέρια το Bremain, την παραμονή δηλαδή, ε, ε, υπολογίζουμε το κόστο τη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν είναι το βασικό μας σενάριο και το τονίζω αυτό και θα επανέλθω σε αυτό. Το χρησιμοποιούμε απλώς για να είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο αντίκτυπος του Brexit. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω ότι αυτή η μελέτη έγινε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και στη συνέχεια δεν συμπεριλάβαμε τη μεταβατική περίοδο γιατί τότε ήταν πολύ αβέβαιο κατά πόσον θα υπάρξει μεταβατική περίοδος. και θα τύχει και διαπραγμάτευσης. Στην επόμενη διαφάνεια ε, βλέπετε ότι κάθε φορά που πρέπει να κάνουμε ε, μια μελέτη με διάφορες εναλλακτικέ εκδοχές ε, πρέπει να έχουμε διάφορες υποθέσεις. Και εδώ έχουμε κάποιες από τις υποθέσεις που χρησιμοποίησαμε για να εξετάσουμε τα διάφορα ενδεχόμενα. Ας δούμε το σκληρό Brexit. Υποθέτουμε ότι το κόστος του εμπορίου θα αυξηθεί κατά 11% ε, ο λογαριασμός του Brexit θα είναι 11 δις ευρώ, θα, αυξηθούν, θα μειωθούν οι άμεσες ξένες επενδύσεις κατά 12% και η μετανάστευση θα μειωθεί κατά... 500.000 ε, ε, και ανθρώπους και θα μειωθούν κατά 1,3% οι θέσεις εργασίας των μεταναστών. Να σας πω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Αν πατήσει το κουμπί πάει πίσω αντί να πάει στην επόμενη διαφάνεια. Αυτή τη διαφάνεια δεν θα σα τη συζητήσω γιατί αναφέρθηκα στις συνέπειες του Brexit και πάμε στα ε, συνέπειε για την ε, οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Και πάλι σας υπενθυμίζω αυτό που είπα, η μελέτη έγινε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, δεν υπήρχε μεταβατική περίοδο τότε. Το αποτέλεσμα θα είναι δύο ετών ύφεση και στις τρεις εκδοχές, και σε σκληρό και σε ήπιο Brexit και σε συμφωνία ελευθέρου εμπορίου όταν το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα πληγεί πολύ περισσότερο και για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ε, στο, ε, στην εκδοχή του σκληρού Brexit σε σχέση με το ήπιο Brexit. Και τώρα εδώ στην επόμενη διαφάνεια Νομίζω ότι ε, αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι πλήττεται η μακροπρόθεσμη δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, περνάμε από το 1% ε, παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 1,3% συγγνώμη, από το 2,1% παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 1,3% αν φύγει με ε, σκληρό Brexit. Και η βασική μοχλή της μείωσης είναι χαμηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα και χαμηλότερος παράγοντας παραγωγικότητας. Το σωρευτικό αποτέλεσμα στην οικονομία της Ένωσης είναι γύρω στο 2% το ΕΠ το 2024 σε όλα τα σενάρια και αυτό το βλέπουμε με βάση το σενάριο ανάπτυξη του Οκτωβρίου 2018 που έχει αλλάξει, αλλά αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι πως υπάρχει μια μικρή διαφορά με το βασικό σενάριο, κατά το οποίο δείχνει ότι υπάρχει περιορισμένο αποτέλεσμα του Brexit στην οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης. Βλέπετε ότι ο αντίκτυπος των τριών σενάριων ε, βλέπετε ότι έχει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά ουσιαστικά τα ίδια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε οικονομικά μιλώντας ε, το είδος του σενάριου έχει πολύ λιγότερη σημασία ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Γιατί, γιατί ε, όπως είπαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερος εταίρος ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά έχει το αντίστροφο. Αλλά συμβαίνει αυτό για την Ολλανδία, οπότε είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μου. Επόμενη διαφάνεια. Το πιθανότερο σενάριο αυτή την στιγμή, αυτό το οποίο υποθέτουμε ότι θα γίνει, είναι μια διετής μεταβατική περίοδος που μάλλον ε, φαίνεται ότι συμφωνήθηκε πριν από δύο μέρες και μετά μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, μια νέα συνθήκη και το τι μορφή θα μπορούσε να έχει είναι ακόμα κάτι το πολύ αβεβαίο και η αβεβαιότητα ήδη είναι κάτι το οποίο προκαλεί ζημία στις βρετανικές ε, εταιρείε, όμως υπάρχουν συγκρίσεις με τις υφιστάμενες συνθήκες ε, που έχουν γίνει παραδείγματο χάρη με τον Καναδά, όπου βλέπουμε ότι όλα τα προϊόντα ουσιαστικά έχουν δεσμού κοντά στο 0%. Οπότε, εάν υπάρχει συνθήκη, οι δασμοί θα είναι 0% ή πολύ χαμηλή. Κάτι σαν ένα καθεστώς Καναδά συν. Στο πιθανότερο σενάριό μας, όπως είπα. Προβλέπουμε λοιπόν και βλέπετε σε αυτήν την διαφάνεια πως ε, θα πέσει η Βρετανική ανάπτυξη στο 4% στο 2020 και θα ανακάμψει σιγά σιγά μετά και μετά τις επόμενες διαφάνειες μπορούμε να τις προσφεράσουμε, δεν υπάρχει και χρόνος. Ε, καλό είναι λοιπόν πάντα να ξέρουμε τα γεγονότα και κάποια από αυτά τα γεγονότα είναι δυσάρεστα, το έχω δει και σε προηγούμενες συζητήσεις και ακροάσεις αλλά νομίζω ότι τα γεγονότα θα σας ε, δώσουν μια πιο ενήμερη θέση στις ε, διαπραγματεύσεις και ελπίζω και οι Ευρωπαίοι και οι Βρετανοί να δουν καλά τα σενάρια μας και να γνωρίζω ότι είναι πολύ απεσιόδοξα και αρνητικά. Ελπίζω λοιπόν να ε, το ξανασκεφτούν πριν προχωρήσουν σε ένα σκληρό Brexit. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμά σας. Και τώρα θα δώσω τον λόγο στην Κίρστη Χιούζ, Διευθύντρια του Σκοτσέζικου Κέντρου για τις ε, Ευρωπαϊκές Σχέσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση να σας απευθυνθώ σήμερα. Δεν είμαι βέβαιη ότι θα προσφέρω περισσότερη αισιοδοξία. Ξέρουμε τι λένε τα κόμματα που είναι υπέρ της παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου και ξέρουμε ότι φτάσαμε στο 66-68% υποστήριξη υπέρ της παραμονής της Σκοτίας της πρόσφατας δημοσκοπήσεις. Σε κάποιο βαθμό λοιπόν ακόμη παραμένει ένα ενδεχόμενο και μια ελπίδα. Ίσως αυτό είναι η μόνη νότα αισιοδοξία ότι το Brexit μπορεί να μην συμβεί. Αυτό που θέλω να κάνω είναι πρώτα απ' όλα να κάνω κάποια σχόλια για την πολιτική κατάσταση, διότι νομίζω ότι το Brexit το υποκινούν οι πολιτικές δυνάμεις και βεβαίως οι οικονομικές συνέπειες υπό τα περισσότερα σενάρια θα είναι αρνητικά. Η χώρα πηγαίνει προς μια οικονομική υποβάθμιση, αλλά οι πολιτικές δυνάμεις που το αποκοινούν αυτό ε, είναι σαφείς. Υπάρχει σταθερότητα στην πολιτική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και υπάρχει και κάποιο είδους ε, θεσμική συνταγματική κρίση, η οποία θα επηρεάσει και την έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων και το τι είδους σχέση θα διαμορφωθεί στο μέλλον. Μερικά σύντομα σχόλια λοιπόν για την πολιτική κατάσταση και μετά μερικά σχόλια για, την οικονομική για τον οικονομικό αντίκτυπο όπως τον αντιλαμβάνομαι και μετά θα ολοκληρώσω. Ξέρουμε ότι από την Τερέζα Μέη η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θέλει την ευρύτερη και βαθύτερη δυνατή σχέση που μπορεί να ε, φανταστεί κανεί ε, από οποιαδήποτε σχέση ελεύθερων συναλλαγών που γνωρίζουμε από τον κόσμο. Αλλά όπω είπα, η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ε, βασίζεται και καθορίζεται από πολιτικέ επιταγέ. Και αυτό ε, προξενεί και την αβεβαιότητα που περιέγραφα πρέπει να λυθεί το θέμα του πώς θα μείνει ανοιχτό το σύνορο με τη Βόρεια Ιρλανδία και η πρόκληση για το Ηνωμένο Βασίλειο, στην οποία χρειάζεται απάντηση, είναι αν το backstop θα είναι μέρος ε, του τελωνιακού χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι και πώς θα αποφύγει το Ηνωμένο Βασίλειο ένα σύνορο στην θάλασσα της Ιρλανδίας. Αυτό απαιτεί και από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο να είναι μέρο μια τέτοια ε, διευθέτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και εμπορευμάτων, αλλά εξαρτάται και από τι κοκκίνε γραμμέ, τι κατευθυντήριε γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να μην είναι αποδεκτή μια τέτοια λύση για του Ευρωπαίου. Στη θάλασσα τη Ιρλανδία, όπω ξέρουμε, αυτή τη στιγμή ε, η ε, Βρετανική κυβέρνηση επηρεάζεται από τον DUP και θα συνεχίσει. Εάν η κυβέρνηση σκεφτόταν την ε, πιθανότητα του συνόρου στη θάλασσα της Ιρλανδία, μπορεί και να βρισκόταν κάποια είδου συνένεση στο κόμμα των συντηρητικών. Όμως και εκεί υπάρχει πολύ πολιτική αβεβαιότητα. Επίσης, ω προς τα πολιτικά πράγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία του Brexit ω προ το νόμο για το εμπόριο, του νόμους θα περάσουν για το εμπόριο και την τελωνιακή ένωση το Westminster δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει πλειοψηφία. Μπορεί, εάν οι αντιρρησίες των Τόρις, των συντριπτικών ε, ή ψηφίσουν ε, κάποιοι που είναι υπέρ του Brexit ε, μαζί με την κυβέρνηση, μπορεί να έρθουν και να πούν ότι τελικά θέλουμε τελωνιακή σχέση στο μέλλον. Αλλά μου φαίνεται αρκετά απίθανο δεν πιστεύω η Τερέζα Μέη να μπορέσει να συνασπίσει όλους την κυβέρνησή της και στο κόμμα της και μπορεί να χρειαστούν και γενικέ εκλογέ των οποίων θα είναι άγνωστο το αποτέλεσμα. Μια πιθανότητα είναι να έχουμε πρόορε ε, εκλογές και να υπάρξει κυβέρνηση ψηφία. Και εκεί είναι τρίτο κόμμα στο Westminster το Εθνικό Κόμμα της Σκοτίας που έχει και αυτό πολύ σοβαρή ε, επίδραση στα πράγματα. Μπορεί να καλέσουν τον επόμενο Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου να οργανώσει πάλι δημοψήφισμα για, το για την ε, αποχώρηση παραμονή. Άγνωστο λοιπόν και αυτό. Επίση, για να επανέλθω στην Τερέζα Μέη και την κυβέρνηση τη Βρετανία, είναι πραγματικά η εκεχηρία αυτή τη στιγμή πολύ, ε, βασίζεται σε πολλέ εντάσει και αβεβαιότητα, διότι δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον της σχέση. Θα χρειαστεί ευθυγράμμιση νομοθετική καθώς και διατήρηση της πολιτικής, ε, της πολιτικής κυριαρχίας και της δυνατότητας να υπάρχει ρυθμιστική αυτονομία. Αυτό όμως εξαρτάται και από το τι γραμμές θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμπορική ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Δηλαδή, είτε η Βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να πάει περισσότερο προς το soft Brexit, ή σε μια άλλη πιο ε, ενδιάμεση θέση. Όμω δεν ξέρω αν μπορούν οι πολιτικοί και οι πρόσωποι τη κυβέρνηση να κινηθούν προ αυτή την κατεύθυνση. Για την ώρα αυτή η κατάσταση μεταξύ του ε, δεν φαίνεται να συνάδει με του στόχου τη ευρωπαϊκή πολιτική. Και προφανώ υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πόσο θα είναι ίσοι οι κανόνε του παιχνιδιού εμπορικά και τι εγγυήσει μπορεί να δώσει η ευρωπαϊκή πλευρά θα εξαρτηθεί αν θα κερδιθεί η εμπιστοσύνη ε, από το Ενωμένο Βασίλειο. Δύο ακόμη σύντομες παρατηρήσεις για τα πολιτικά πράγματα ως την θεσμική κρίση, την αναδυόμενη θεσμική κρίση και δεν μιλάω για την Βορειλανδία, μιλάω για το γεγονό για ότι και το Κοινοβούλιο στη Σκωτία και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση διαφωνούν με την Βρετανική κυβέρνηση για την επιστροφή των εξουσιών στις αποκεντρωμένες περιοχές. Αυτή τη στιγμή θα περάσει ένα νόμος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο για να περάσουν νόμοι που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σκοτσέζικη νομοθεσία για το εμπόριο, την γεωργία και άλλα. Αυτό θα δυσκολέψει ενδεχομένω το εμπόριο στο μέλλον και επίσης εξίσου σημαντικό, ακόμη και αν δεν ξέρει κανεί τι θα γίνει στο τέλο με την ε, συμφωνία συνολικά, πώ θα κυρωθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και τι θα γίνει αν δεν κυρωθεί από όλου. Πολιτική αβεβαιότητα και αστάθεια λοιπόν και όλα αυτά ε, γύρουν πολλά ερωτηματικά. Είναι ένα ε, απρόβλεπτο διαπραγματευτικό εταίρο του ΕΒ Βασίλειου συνολικά. Επίση, ε, λίγα σχόλια για τον οικονομικό αντίκτυπο τη μελλοντική συμφωνία και κάποιε λεπτομέρειε. Ο πιο άμεσο αντίκτυπο και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει το Brexit έχουν να κάνουν με νέους τρεγμούς, νέου φραγμού και στα σύνορα και μακρύτερα από αυτά βεβαίω. Έχω ένα κατάλογο από παρόμοια σχόλια με τη Μπάρμπαρα για, την, ε, για το εμπόριο, του, τις ροές, το τι θα γίνει στα σύνορα, για την παραγωγή, για την, ε, το τι θα έρχεται προς τα μέσα και τι θα φεύγει προς τα έξω, εξαγωγές και εισαγωγές, την ελεύθερη κυκλοφορία, για το εργατικό δυναμικό, την ε, μετανάστευση και την κίνηση του εργατικού δυναμικού των εργαζομένων σε πολλούς κλάδους. Νομίζω ότι η μελλοντική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για τις ε, ρυθμίσεις που θα πρέπει να αναλάβουν ή την απόκλησή τους από τις ρυθμιστικές διευθετήσεις μέχρι τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε ακόμα και μπορεί να επηρεάσουν. Θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες λόγω των ε, φραγμών ε, δασμολογικών και όχι και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Κάποια κρατημέλη, ιδίω η Ιρλανδία, θα πληγούν ιδιαίτερως και βεβαίω θα υπάρξει και περαιτέρω αντίκτυπο, ε, θα υπάρξουν συνέπειε σίγουρα σαν ντόμινο στου ε, φόρου, του δασμού, ε, το, τα έσοδα τη κυβέρνηση, τη δυνατότητα επενδύσεων και ούτω καθεξής. Η εκστρατεία του δημοψηφισματο. Ξέρουμε ότι χρησιμοποιεί το επιχείρημα του, του Εθνικού Συστήματο Υγεία, Το εκμεταλλεύτηκαν ω ήταν υπέρ του Brexit, αλλά τελικά είδαμε στην πράξη να συμβαίνει το αντίστροφο. Τώρα ε, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επικεντρώνεται σε μια πιθανή συμφωνία σαν του Καναδά, αλλά τρει φορέ πιο ισχυρή, ή ένα είδο διαθέτηση μέσω του ΠΟΕ. Ή ε, η Τελωνιακή Ένωση και η Ενιαία Αγορά είναι μια άλλη επιλογή. Κάτι όμως που δεν φαίνεται να προκύπτει, ε, αν τα συνδυάσουμε όλα μαζί, δεν δίνει το αποτέλεσμα που θέλουν. Και αυτοί που είναι υπέρ της παραμονής αλλά δέχονται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην ουσία ε, προστηρίζουν αυτό το ιδιαίτερα ήπιο Brexit. Αυτό είναι προβληματικό εάν σκεφτούμε τι γίνεται με την ε, Νορβηγία λόγου χάρη που είναι διαφορετική ως προς το καθεστώς της. Είναι δύσκολο να σκεφτούμε πώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι μέρος της Τελωνιακής ε, Ένωσης και της ενιαίας αγοράς. Δεν μου μένει πολλής χρόνος για να πω για τα στατιστικά δεδομένα, αλλά ήδη ακούσαμε, υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι ακόμη και με την επιλογή της ενίας αγοράς πέφτουν ε, τα έσοδα, 1,6% μείωση τουλάχιστον στην ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από 15 χρόνια και 7,7% μείωση με την επιλογή του ΠΟΕ. Η Ιρλανδική κυβέρνηση και αριθμοί ε, της Επιτροπής δείχνουν μετά από 10 χρόνια 7% μείωση για την Ιρλανδία βάσει του σενάριου του ΠΟΕ ε, και με την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ενιαία αγορά. Είναι λοιπόν πολύ διαφορετικές ε, συνέπειες αναπεριοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και το, τη ζημιά που θα υποστούν, ιδίως στα, στα βορειοανατολικά της ε, Αγγλίας, αλλά και το τι θα γίνει με τη Σκωτία και την Ιρλανδία, εκεί θα υπάρξουν ακόμα αρνητικότερε συνέπειε από το μέσο όρο τη υπόλοιπη χώρα. Να ολοκληρώσω και να πω κάτι γιατί σε σχέση με αυτά που είδαμε στα νέα για την Αλία ε, και που είναι αρκετά συγκινησιακά, είναι ειδήσει που ε, προκαλούν εντύπωση. Παρόλα αυτά ε, φαίνεται η πολιτική να επιδιώκουν μια συμφωνία ελεύθερου μπορίου με την ελεύθερων συναλλαγών με, τον, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η αίσθηση που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν βρισκόμαστε σε μια απλή σταθερή κατάσταση ήρεμων διαπραγματεύσεων για το επόμενο εξάμεινο για να μεταφέρουμε το πλαίσιο των μελλοντικών μα σχέσεων. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχουμε την πλήρη εικόνα οικονομική και πολιτική για τον αντίκτυπο του Brexit και στις δύο πλευρές ε, και όχθε της μάχης. Τώρα, ε, είναι σαφές ότι θα έχουμε μεταβατική περίοδο μέχρι το τέλος του 2020 για να δούμε τι θα κάνουμε. Για να δούμε λοιπόν το τι θα γίνει σε αυτήν την μεταβατική περίοδο θα ακούσουμε τον κύριο Λόου από το Κέντρο για την Ευρωπαϊκή Μεταρρυθμίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από αυτήν την συζήτηση εγώ θα εστιάσω σε κάτι πιο ε, στενό συγκεκριμένα το τι σημαίνει η υποσημείωση 77 της ε, συμφωνίας της ε, Δευτέρας. Δεν θα εστίαζα συγκεκριμένα στις πτυχές των συμφωνιών με τρίτες χώρες. Ευχαριστώ να δεχτώ ερωτήσεις μετά. Αλλά είναι κάτι από αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει πλήρως αντιληπτά την ημέρα που θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ένωση, ακόμα και αν περάσουμε σε μεταβατική περίοδο που εσείς ε, έχετε ε, μεγάλη σιγουριά ότι θα γίνει, ελπίζω εγώ, εν πάση περιπτώσει, τη στιγμή που θα φύγουμε, δεν θα είμαστε συμβαλόμενο μέρος, το Ηνωμένο Βασίλειο εννοώ, στις ε, συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες που αφορούν εμπόριο αλλά και άλλα πράγματα που αφορούν ισοδυναμία, αναγνώριση συμφωνιών, συμμόρφωσης και μέχρι προσφάτως δεν ε, ξέραμε το τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Και οι συμφωνίες αυτές, οι εμπορικές, ε, είναι με χώρες που εισάγουν ε, περίπου, το 100, περίπου 12% των Βρετανικών εξαγωγών. Είναι μεγάλο ζήτημα, δηλαδή αφορά χώρες όπως η Ελβετία, η Τουρκία, η Κορέα, χώρες ΕΟΧ ε, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και μέχρι τον Ιανουάριο φέτος η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν ότι θα αντικαταστήσουμε όλες αυτές τις συμφωνίες μέχρι τον Μάρτιο του 2019. Το είπε ο Λίαμ Φόξ στο Κοινοβουλίο. Αυτό δεν ήταν ποτέ δυνατόν. Δεν ξέρω γιατί είπαν κάτι τέτοιο. Ίσως γιατί ε, μοιάζει τόσο σίγουρο ότι θα υπάρξει μεταβατική περίοδος. Αλλά ευτυχώς άλλαξε η προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν κάτι το οποίο είχαμε ε, συστήσει και εγώ και το κέντρο μου. Ε, δεν νομίζω να τους επηρέασα, αλλά καλό είναι να σκέφτεται κανείς έτσι. Και τον Ιανουάριο φέτος άλλαξε θέση το Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα σκοπεύει να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πείσει τις ε, τρίτες χώρες να συνεχίσουν να μεταχειρίζονται το Ηνωμένο Βασίλειο ως κράτος μέλος ε, στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών κατά τη διάρκεια της μεταβατικής ε, περίοδου, παρά το ότι δεν θα είναι πια. Και ερχόμαστε τώρα στην υποσημείωση 77 που λέει η Ένωση θα κοινοποιήσει στα άλλα μέλη των, μέλη των συμφωνιών αυτών πώς ε, για τη μεταβατική περίοδο το Ηνωμένο Βασίλειο θα την χάνει αυτή τη μεταχείριση. Μέχρι εδώ όλα καλά. Το θέμα έχουμε είναι ότι αυτή ήταν ε, η μόνη δυνατή προσέγγιση ε, και έξυπνο είναι ότι λέει ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ειδοποιήσει αυτές τις χώρες, δεν θα τους ρωτήσει δηλαδή. Αλλά δεν μπορούμε όμως να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο μέσω μιας διμερούς συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου σε τρίτες χώρες και βεβαίω έτσι όμως μετατοπίζεται το βάρος ε, στις τρίτες χώρες που θα πρέπει να πούν όχι εμείς δεν θέμε να θεωρούμε το Ηνωμένο Βασίλειο συμβαλόμενο μέρος των συμφωνιών. Κατ' οποίο εντάξει είναι δύσκολο να γίνει πολιτικά αλλά θεωρώ ότι κάποιες χώρες θα το κάνουν. Και ο λόγος είναι πως υπάρχει μια κάποια συμμετρία σε αυτό το ζήτημα. Εννοώ δηλαδή ότι Μπορεί να μην έχουν πλέον προτιμησιακή μεταχείριση οι βρετανικέ εξαγωγέ από την Κορέα. Οι κορεατικέ εξαγωγέ προ το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπαίνουν υπό προτιμησιακού όρου γιατί θα δεσμεύεται ακόμα από το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο του Ηνωμένου Βασίλειο και τους άλλους συνοριακούς ελέγχους. Οπότε πλησιάζουμε σε ένα σημείο όπου θα υπάρχει μία ασυμμετρία και δίνει στις τρίτες χώρες ένα μοχλό πίεση του Ηνωμένου Βασίλειου. Και αυτό το οποίο θεωρώ ότι θα δούμε είναι οι τρίτε χώρε να ζητάνε παραχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο όταν θα αντικατασταθούν αυτέ οι συμφωνίε, κάτι το οποίο θα ε, πρέπει να γίνει, απλά εδώ πέρα κερδίζει χρόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα ζητήσουν τις παραχωρήσει τώρα για να ε, συμφωνήσουν με τον συμβιβασμό αυτό Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Ξέρουμε ότι αυτό συμβαίνει ως ένα βαθμό. Υπάρχουν συζητήσεις με την Κορέα για την μελλοντική συμφωνία όπου το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ζητήσει ε, την ε, βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προϊόντα του να θεωρούνται ενωσιακής προέλευσης. Οι Κορεάτες είπαν θα το σκεφτούμε αλλά δεν θέλουμε τότε θα πρέπει να δούμε το τι θα γίνει και με τις ε, κινέζικες εισαγωγές που εξάγουμε προς τον Βασίλειο. Οπότε και αυτό θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Και τελικά νομίζω, αυτό είναι γνώμη βεβαίω. ότι πολλέ χώρες θα πάρουν παραχωρήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για να δεχτούν την μεταβατική αυτή συμφωνία και νομίζω ότι τελικά οι περισσότερες θα το επιτρέψουν. Δύσκολες, λίγες θα δυσκολέψουν τα πράγματα και θα αρνηθούν με επιθετικό τρόπο την προτιμησιακή μεταχείριση στα προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ τα δικά τους θα συνεχίσουν να την λαμβάνουν. Ίσως κάποιες ε, το κάνουν αυτό και θα δούμε. Ε, το ερώτημα τώρα είναι γιατί ε, θα πρέπει να ενδιαφέρει αυτό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει ότι θα ειδοποιήσει αυτές τις τρίτες χώρες ότι θα πρέπει ε, για τους σκοπούς αυτούς να θεωρούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέλος της Ένωσης, αλλά ε, προσωπικά έχω ένα ερώτημα για το πόσο πολιτικό κεφάλαιο είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να σπαταλήσει για κάτι τέτοιο αν μια χώρα πει δεν θέλει να το κάνει. Και αυτό είναι ένα ερώτημα για το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν, το Συμβούλιο. Εάν δηλαδή θα ρίξουν όλο τους το διπλωματικό βάρος, εάν πει όχι η Νότια Αφρική ας πούμε. Αλλά γιατί θα έπρεπε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πως υπάρχει ένα προηγούμενο όσον αφορά την ε, συνεργασία στο διεθνές εμπόριο μετά το Brexit, δηλαδή συνεργάζονται οι δύο πλευρές στον ΠΟΕ όσον αφορά τις ε, ποσοστώσεις, ε, τις δασμολογικές και βεβαίως και οι διαπραγματευτικές οδηγίες λένε πως αναμένεται από το Ηνωμένο Βασίλειο να τηρήσει το κομμάτι που το αναλογεί στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Ε, δηλαδή, καλό θα ήταν να είναι όλοι ευγενικοί. Όμως, αυτό σημαίνει πως υπάρχουν κάποιες συνέπειες για τις χώρες που θα βασίζονται στις 27 χώρες. Παραδείγματο χάρη, αν η Κορέα δεν επέτρεπε την ε, βρετανική συνεισφορά στα κοινοτικά προϊόντα, αυτό σημαίνει ότι κάποιες εταιρείες που εξάγουν στην ε, Κορέα πλέον δεν θα είχαν προτιμησιακή μεταχείριση. Πρέπει να αναφέρω ότι αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα για τους εξαγωγείς του Ηνωμένου Βασιλείου παρά για τους εξαγωγείς της Ένωση, αλλά υπάρχει. Ο άλλος λόγος για τον οποίο θα μπορούσε να ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και να κάνει κάτι παραπάνω από το να αποστείλει μια επιστολή είναι ότι θα επέτρεπε περισσότερο χρόνο ε, να διαπραγματευτεί τριμερός με τις ε, τρίτες χώρες ε, για το ποιες συμφωνίες θα αντικαταστήσουμε αυτές τις υφιστάμενες συμφωνίες και ο λόγος για τον οποίο θα ήθελε να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι θα ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης να διαπραγματευτεί τις διατάξεις για την σώρευση της προέλευσης όπως είπα όσον αφορά δηλαδή το εάν τα βρετανικά προϊόντα θα χαρακτηρίζονται ως ε, κοινοτικά για την ε, μεταβατική αυτή περίοδο. Υπάρχει και η Ευρωμεσογειακή Συμφωνία. Ίσως είναι λιγότερο πρόβλημα για τις ε, συμφωνίες με την Ιαπωνία, γιατί υπάρχουν εκεί πέρα κάποιοι μηχανισμοί που προέβλεπαν ακριβώς το θέμα της ε, σώρευση ε, της ε, προέλευση αν υπάρξει κάποια συμφωνία με τρίτο μέρος και από πλευρά Ιαπωνία και ΕΕ αλλά έχουμε συμφωνίες με την Κορέα, το Μεξικό και τον Καναδά που επιτρέπεται πιθανώ με τις ΥΠΑ, αλλά όχι αλλού. Οι συνέπειε ε, του να μην βοηθηθεί το Ηνωμένο αν οδηγούσε στο ότι το βρετανικό μέρος των εξαγωγών να μην θεωρείται πλέον κοινοτικό θα οδηγούσε βέβαια σε κάποια διαταραχή και μετά θα μετατοπίζονταν η ε, αλυσίδα παραγωγής είτε στην Ένωση είτε στον Ηνωμένο Βασίλειο, πιθανότερα στην Ένωση. Και μετά οι συνέπειες του να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ότι θα πάμε σε μια τριμερή διαπραγμάτευση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο καθώς ε, σημαίνει ότι θα υπάρξουν ε, και απαιτήσει μετά από την Ένωση. Και εδώ πέρα τελειώνω. Η μετάβαση λοιπόν είναι και αυτή πρόκληση. Και τώρα για την πολιτική πλευρά έχουμε τώρα τον ε, Νικολάη Βουνοντάρτσα από το Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών ε, ε, ε, Υποθέσεων και Υποθέσεων Ασφαλείας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θα προσπαθήσω να προσθέσω την πολιτική και την νομική σκοπιά στο θέμα της μετάβασης στην εμπορική πολιτική του, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σχέση με αυτά που ακούστηκαν αλλά περισσότερο κοιτάμε τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι θα βασίσω το μεγαλύτερο τμήμα της παρουσίασής μας ε, στο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις συμφωνίες ε, ευτυχώς ε, η Επιτροπή και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν διαπραγματευτεί τα περισσότερα πράγματα της μεταβατικής περίοδου αυτή την εβδομάδα επομένως αυτά είναι συμφωνημένα σε πολιτικό επίπεδο βασική ε, πρόκληση, όπως ανέφερε και ο ΣΑΜ, είναι ότι η μετάβαση στην πραγματικότητα είναι ε, μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 27 και θα επηρεάσει και την ε, συμφωνία τρίτων και την κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου ενώπιον τρίτων χωρών. Την ημέρα που θα αποχωρήσει επισήμω ε, το Ηνωμένο Βασίλειο στις 29 Μαρτίου του 2019 γίνεται τρίτη χώρα και δεν καλύπτεται πλέον από αυτέ τι συμφωνίε. Και το τρίτο πολιτικό και όχι τόσο νομικό θέμα είναι τι ακριβώ θα γίνει με αυτό. Και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά κυρίω θα επικεντρωθώ στο τι σημαίνει για την Ευρώπη των 27 και τι θα μπορούσε και θα έπρεπε να κάνει γι' αυτό. Καταρχάς, τι ακριβώς σημαίνει η μετάβαση για το Ηνωμένο Βασίλειο ε, όσον αφορά την εμπορική του πολιτική ενώπιον της ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουμε κάτι το οποίο ε, θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε υπερήπιο ε, Brexit, να παραμένει στην ενή αγορά και στην Τελωνιακή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο να δεσμεύεται να εφαρμόσει το τελωνιακό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την τελική του αποχώρηση. Δηλαδή η ημερομηνία λήξης είναι το τέλος της μεταβατικής περίοδου βάσει της οποίας θα δεσμεύεται από όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Και για να δείξουμε την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωσης ως ε, διεθνής παράγων, η Επιτροπή και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν ότι από όλο το κεκτημένο που δεσμένει το Ηνωμένο Βασίλειο, οι διεθνείς συμφωνίες περιλαμβάνονται πλήρως και το Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεούται πλήρως ε, από όλα όσα απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι, και αυτό το σημαντικό το ανέφερε και ο ΣΑΜ, από τα ωφέλη δεν καρπώνεται τα ωφέλη. Τώρα, όσον αφορά την όλη μετάβαση, όπου το Ενωμένο Βασίλειο ε, εμπίπτει σε ένα καθεστώς ε, ε, του λεγόμενου ε, αυτού που θα αποδέχεται τους κανόνες, δεν συμμετέχει στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν σημαίνει απλώς τα συνήθι θεσμικά όργανα που αποφασίζουν για το εμπόριο, αλλά και τους συγκεκριμένου φορείς που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες για την εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών, με δύο εξαιρέσεις θα έλεγα, εκτός από την περίπτωση περίπτωση στην οποία συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο αυτοδικαίως, όπως για παράδειγμα στον ΠΟΕ, ή όταν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι προς το συμφέρον της να εμπλέξει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει λοιπόν πάντα ένα παραθυράκι. Κάτι άλλο το οποίο είναι επέκταση των συνήθων κανόνων ε, της μετάβασης είναι ότι οι νέες συμφωνίες του Ηνωμένου Βασιλείου που θα αποφασιστούν και θα κυρωθούν στη διάρκεια της μετάβασης, παραδείγματος χάρη η Εταιρική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας ή Ευρωπαϊκή Ένωση Μερκοσούρ, αν τεθούν σε εφαρμογή στη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου θα ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να έχει λόγο το Ηνωμένο Βασίλειο γι' αυτό. Ακόμα λοιπόν και στο εμπόριο μπορεί να ε, από υποχρεώσεις που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια τη μετάβαση χωρί να συμμετέχουν. Απ' την άλλη πλευρά του νομίσματο όμω, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί μόνο να διαπραγματευτεί αλλά και να υπογράψει και να εφαρμόσει νέε συμφωνίε εμπορίου, αλλά ε, δεν μπορεί να τι θέσει σε ισχύ. Δηλαδή, μπορούν να τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία μετά τη μετάβαση, αλλά δεν μπορούν χωρί την έγκριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθούν σε ισχύ πριν τελειώσει τελειώσει η μεταβατική περίοδος. Ορισμένες φορές λειτουργεί. Αυτό το μηχαναματάκι με τις υπέρυθρες δεν είναι πολύ καλό αυτό που ενδιαφέρει του περισσότερου από εμά είναι τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη των 27. Τι τη νοιάζει την Ευρώπη των 27, εάν υπάρχουν ακόμα υποχρεώσει για το Ηνωμένο Βασίλειο ε, και αν δεν υπάρχουν τριβέ ε, στο εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Να σα αναφέρω τρει λόγου για του οποίου θα έπρεπε να ενδιαφερόμαστε. Ο πρώτο είναι αυτό που ανέφερε ήδη ο, ο ΣΑΜ, ε, οι κανόνε ε, προέλευση και τα προϊόντα τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω αυτοκινητοβιομηχανία βιομηχανίας που ε, υπάρχουν ε, ε, εξαρτήματα των οχημάτων που παράγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν λοιπόν είναι κάτω από το όριο που καθορίζονται σε κάποιες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα και αν παράγονται στην ενιαία αγορά όπως θα ισχύει για τη μετάβαση, δεν είναι αδασμολόγητα για εξαγωγές στην Κορέα, που σημαίνει ότι θα επηρεάσει και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ε, δεύτερον, νομίζω δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω στα περισσότερα μέλη της Επιτροπής ε, ότι υπάρχει λόγος για τον οποίο η εμπορική πολιτική είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απορρέει από την ε, ενιαία αγορά και όταν υπάρχει κοινή τελωνιακή πολιτική πρέπει υποχρεωτικά να έχει και κοινή εμπορική πολιτική. Εάν ε, ισχύσουν τα θέματα συμφωνών ελευθέρων εναλλαγών για το Ηνωμένο Βασίλειο σημαίνει ότι υπάρχουν οι ίδιοι δασμοί και κατά την εξαγωγή στην εσωτερική αγορά και είναι διαφορετική η δασμή των κρατών μελών της ε, ε, ε, ενιαίας αγοράς όταν εξάγουν σε τρίτες χώρες. Και αυτό φυσικά δημιουργεί στρεβλώσεις εντός της ενιαίας αγοράς και προϊόντα τα οποία παράγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο τιμολογούνται διαφορετικά από όταν παράγονται οπουδήποτε άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάποιοι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αποκαλούν ετοιμότητα για τον Brexit. Η εκτίμηση της αλυσίδας αξίας θα πρέπει να γίνει όχι μόνο στο τέλος της αλυσίδας, αλλά και στην αρχή των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Ένα άλλο που επηρεάζει τις επιχειρήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 είναι η αβεβαιότητα. Οι επιχειρήσεις πάντα ε, ε, τονίζουν ότι πρέπει η μετάβαση να παρέχει ασφάλεια. Η αβεβαιότητα όμως για το τι θα συμβεί με τις εμπορικές συμφωνίες υπάρχουν δημιουργεί και αβεβαιότητα για τι μελλοντικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου, εάν δεν λάβουμε απαντήσει από τρίτε χώρε για το πώ θα συμπεριφερθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο στη διάρκεια τη μεταβατική περίοδου. Αντί λοιπόν να υπάρχει ασφάλεια και ελπίζοντα να έχουμε και νομική συμφωνία για τη μετάβαση, ε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ασφάλεια που επιθυμούμε. Και εδώ φτάνω και στο τελευταίο και ίσω και το πιο κρίσιμο σημείο. Τι επιλογέ έχουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το πρώτο είναι ότι από νομική σκοπιά είναι πολύ πιο εύκολο και από πολιτική σκοπιά είναι πολύ δύσκολο. Επέκταση των ε, σκηνοποίηση του άρθρου 50 για το κατά πόσον ε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μείνει κράτος μέλος μέχρι το 2020 και να μην υπάρχει μεταβατική περίοδος, απλώς παράταση της περίοδου πριν την αποχώρηση. Αυτό δεν το επιθυμεί κανείς όμως, ούτε το ΕΒ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ακόμα λιγότερο πιθανό, δεδομένου ότι τώρα φαίνεται να υπάρχει πολιτική συμφωνία για τη μετάβαση. Ουσιαστικά λοιπόν το αποκλείουμε αυτό το ενδεχόμενο ή θα έλεγα ότι τουλάχιστον ρεαλιστικά για τις ε, διαπραγματεύσεις όπως έχουν αυτή τη στιγμή αποκλείεται αυτό. Η δεύτερη επιλογή είναι να μην κάνουμε τίποτα. Δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο να πει ότι αυτό αφορά κυρίω το Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, οι επιχειρήσει μα ε, θα επηρεαστούν, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποια ωφέλη, διότι μπορεί να υποχρεωθούν να μετεγκαταστήσουν κάποιε από τι αλυσίδε αξιών του ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κλπ. Όπως σας είπα ότι αυτό θα γίνει ανάλογα με το τι θα προκύψει κυρίως για τις αρνητικές και ανεπιθύμητες συνέπειες για ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να ε, βρει μια λύση στο πρόβλημα με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις τρίτες χώρες. Η τρίτη επιλογή είναι λίγο στο ενδιάμεσο. Τι ακριβώς ήθελε να πετύχει αρχικό στο Ηνωμένο Βασίλειο να ε, ξαναδημιουργήσει τις ε, Συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες. Ουσιαστικά τι μετακυλήσει στο μέρο τους. Και νομίζω ότι αυτό δεν προβλέπεται ακόμα, αλλά τουλάχιστον και από πλευρά ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανεπιθύμητο. Διότι αφενό δεν θα επιλύσει το πρόβλημα των κανόνων ε, προέλευση, διότι αν υπάρχουν ξεχωριστέ συμφωνίε ελευθέρου συναλλαγών για το Ηνωμένο Βασίλειο και τι άλλε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κανόνε για την προέλευση θα ισχύουν, επομένως δεν θα λύνει το πρόβλημα και ε, δεύτερον δεν συνάδει και με αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετάβαση, δηλαδή να μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Τελωνιακή Ένωση και στην νέα αγορά και να μην υπογράψει νέε συμφωνίε δικέ του. Επομένω, αντιβαίνει στην ίδια αρχή που μόλι συμφωνήθηκε για τη μεταβατική περίοδο. Ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να θέσει σε ισχύ δικέ του συμφωνίε ελευθερωπορίου στη διάρκεια τη μεταβατική περίοδου. Έχω και ένα λεπτό ακόμα και την τελευταία επιλογή που βρισκόμαστε τώρα, συμφωνία με τρίτε χώρε να συμπεριφερθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο ω μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια τη μεταβατική περίοδου. Και έχει αυτό και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε τη δυνατότητα να διατηρήσει το status quo και για τις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά κατά την άποψή μου υπάρχουν ε, σοβαρά προβλήματα με αυτό το ενδεχόμενο. Καταρχά, η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώ κοινοποιεί σε τρίτες χώρες. Ε, τίποτα δεν είναι διατεθειμένη να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιέσει το ζήτημα προ το παρόν. Και το θέμα είναι πότε του το κοινοποιεί και τι θα πούν οι τρίτε χώρε. Πότε μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση επισήμω να κοινοποιήσει σε τρίτε χώρε, μόνο όταν η συμφωνία αποχώρηση ε, θα υπογραφεί. Και αυτό θα γίνει τον Οκτώβριο ή και αργότερα στη διάρκεια του 2018, που σημαίνει ότι έχουν ελάχιστο χρόνο επιχειρήσει για να έχουν μια κάποια εξασφάλιση. Και επίση, όπω είπε και ο Σαμ, υπάρχουν κίνητρα να πούνε ότι το επιθυμείτε αυτό, α ξανακάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διάρκεια τη μεταβατική περίοδου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύεται από τι υποχρεώσει των τρίτων χωρών και επομένω μπορεί να προσφέρει ελάχιστα κίνητρα ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να χαίρει ειδικού καθεστώτο στη διάρκεια αυτή τη περίοδου. Επομένω, η εντύπωσή μου και η αξιολόγησή μου διαφέρει λίγο από του ΣΑΜ στο ότι οι τρίτε χώρε θα δούνε τι μπορούμε να αποκομίσουμε εμεί από αυτή τη συμφωνία και τουλάχιστον στην αρχή θα διστάσουν να δώσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο καθεστώ ε, κράτου μέλου Ευρωπαϊκή Ένωση απευθεία στη διάρκεια τη μεταβατική η αξιολόγησή μου είναι ότι αυτό που μάλλον βλέπουμε είναι μια παραταταμένη περίοδος αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις που δεν θα επιλουθεί σύντομα και ε, Φαντάζομαι ότι θα έχουμε και εμβαλωματικά λύσεις από τρίτες χώρες ε, και δεν θα έχουμε μια συνολική απόφαση που θα ληφθεί από όλες τις χώρες και θα είναι κοινή για όλους. Και γι' αυτό ακριβώ νομίζω, και αυτό είναι και το τελευταίο που θα πω, οι επιχειρήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν να προετοιμαστούν για το Brexit ε, στη διάρκεια τη μετάβαση και δεν θα μπορούν να περιμένουν μέχρι το τέλο τη μετάβαση. Τουλάχιστον αυτέ που κάνουν εξαγωγέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα, αυτό σημαίνει ότι το Μίνι Κούπερ από τη Βρετανία θα το μεταχειριστεί η Νότια Κορέα ως ένα μη ευρωπαϊκό αυτοκίνητο βάση του τελωνιακού καθεστώτος που θα ισχύει. Να και κάτι το καινούριο, μια νέα ιδέα για μένα για να τη σκεφτώ. So. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Δύο λεπτά ο καθένας θα έλεγα και ως μόνιμος εισηγητής η κυρία Γκοτλίβε Ρόδους. Ευχαριστώ. Σε ένα λεπτό δεν μπορώ να θέσω όλα τα ερωτήματα που έχω. Έχω όμως ένα ερώτημα αρχής. Ακούστηκαν ε, διαφορετικά σενάρια. Ακούστηκε ότι το χ το είναι πιθανότερο, αλλά έχω την εντύπωση ότι Κάθε μέρα προκύπτει κάτι νέο. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να εγώ να ακούσω από τους ειδικού είναι ο καθένας από τη δική του την ειδικότητα και τη σκοπιά. Τι θα ήταν το λογικότερο σενάριο ή το πιθανότερο κατά την αποψή σας το επιθυμητό αν θέλετε, για την Ευρώπη των 27. Σας ευχαριστώ για τους σοσιαλδημοκράτες, ο Ντέιβιτ Μάρτιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα για τους κανόνες προέλευσης. Φανταστείτε. Αν υποθέσουμε ότι θα συνεχίσουν να σωρεύουν τους κανόνες προέλευσης ε, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην έχει αντίρρηση κάποια τρίτη χώρα, αλλά δεδομένων των κανόνων του ΠΟΕ, κάποιος ανταγωνιστής μια εταιρεία σε μια τρίτη χώρα να πει ότι δεν το δεχόμαστε. Ε, και θα είχε πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Οπότε, ακόμα και αν συμφωνήσουν οι τρεις χώρες, υπάρχει, οι τρεις πλευρές, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Και κάτι άλλο που ίσως αφορά κάποιον άλλον ομιλητή ένα από τα παραδείγματα που άκουσα είναι ότι τα αυτοκίνητα, τα μίνι, αυτήν την στιγμή δεν θα μπορούσαν να θεωρούνται ούτε βρετανικό ούτε ευρωπαϊκό προϊόν. Ε, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Πιθανώς ε, θα ισχύσει αυτό το οποίο λέτε, θα μετατοπιστεί κάπου αλλού η παραγωγή για να θεωρείται ή το ένα ή το άλλο. Για τους δύο πρώτους ομιλητές, ειδικά τις δύο πρώτες ομιλήτριες, για το θέμα της ε, μείωσης κατά 2% του ΑΕΠ ε, της Ένωσης. Ε, δεν έχω κοιτάξει τα μοντέλα, αλλά με εκπλήσει δεδομένου του ότι πρώτον βλέπουμε ήδη κάποια μετατόπιση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα έλλειμμα υπηρεσιών απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι σαφές πως η ανταγωνιστικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου στις υπηρεσίες θα μειωθεί όχι μόνο οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αλλά και άλλες. Οπότε οι υπηρεσίες ε, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μεταφερθούν στην υπηρετική Ευρώπη. Οπότε δεν ξέρω πώς θα ε, έχει πτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μην έχει άνοδο, αλλά και το 2% έστω ναι, και σε βάθος 15 ε, ετών είναι μεγάλο κομμάτι. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν πώς φτάσατε σε αυτόν τον αριθμό. Σας ευχαριστώ για το ECR, κυρία Μακλάφη. Πριν ξεκινήσω με τα δυο μου λεπτά, νομίζω ότι ε, ίσως κάποιοι θεωρούν ότι βρισκόμαστε σε λάθος συνεδρίαση, γιατί ακούμε για το παρελθόν και όχι για το μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω κάποια πράγματα ε, για την ζημία που θα προξενήσει το Brexit, το σκληρό Brexit, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφυγεί την ε, ζημιά στην οικονομία της. Ε, αυτό νομίζω πρέπει να ε, ακούσουμε. Ακούσαμε πολλές απόψεις σήμερα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω αν υπάρχουν κάποιες πηγές για τα σχόλια. Ειδικά κύριε Λό, όταν μιλάτε για τρίτες χώρες που λένε ότι θα κάνουν κάτι. Αναφέρατε την Νότια Κορέα. Ποιες είναι οι πηγές σας όταν λέτε ότι θα έλεγαν όχι στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τις ε, συμφωνίες αυτές. Ευχαριστώ και τον ε, Νικολάη που ε, παρουσίασε λεπτομερώς τις επιλογές μεταξύ των οποίων και η επιλογή του να μην κάνουμε τίποτα. Πρέπει να δούμε το τι σημαίνει αυτό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ζημιά όπως αναφέρεται. Πρέπει λοιπόν να δούμε ακριβώς, γνωρίζουμε ότι η αβεβαιότητα ε, δεν ωφελεί της, ε, την οικονομία. Ε, επανέρχεται λοιπόν ως στρατηγική ή απλά βλάπτη της επιχειρήσης γενικώ. όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και μήπως θα έπρεπε εμείς ως Επιτροπή Εμπορίου να αναζητούμε αυτές τις λύσεις και την εμπορική στρατηγική που θα μας βοηθήσει να βρούμε έναν τρόπο για να έχουμε μελλοντικέ εμπορικέ σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για τους πρασίνους. Έχω δύο ονόματα. Δεν είναι δυνατόν και ο Γιάννικ και ο Κλάους. Ποιος είναι ο Σκιώδης. Γιάννικ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούγοντά σας. φαντάζομαι ότι ο Ντέβιτ Κάμερον έχει κρυφτεί σε κάνα υπόγειο και θα κάνει πολύ καιρό να βγει. Τέλος πάντων, πολύ σοβαρά, πραγματικά το βρίσκω τελείως τρελό, θεότρελο όταν τα σκέφτομαι αυτά που συζητάμε από πολιτική σκοπιές, Επί της ουσίας, επί το θέμα μάλλον των εμπορικών ποσοστώσεων της γεωργίας. Το θέμα είναι ποιο μέρος των ποσοστώσεων θα αναλογούν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρηση και ποιες, ε, ποιο μερίδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως σκέφτομαι λόγω χάρη τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Νέα Ζαλανδία. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις για το αρνί ορίζονται για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η βασική πηγή εισαγωγών και εξαγωγών πλατφόρμα θα λέγαμε για το κρέας του αρνιού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα το χειριστούμε αυτό. Και μετά ε, βλέπουμε δημοσιεύματα στον τύπο, διαβάζουμε ότι το City του Λονδίνου που φοβάται πολύ ότι θα χάσει ένα μέρος του, της του θα μπορούσε να γίνει ένας χώρος όπου οι αναδυνόμενες χώρες θα επενδύσουν και ιδίω θα απελευθερωθούν από μια σειρά από κανόνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λόγω των ε, ευρωπαϊκών αγορών. Λόγω χάρη οι επενδύσεις από τη Σαουδική Αραβία, τη Ρωσία ή και αλλού στην μεταβατική περίοδο θα μπορούσε η Μεγάλη Βρετανία να ε, μετατρέψει το ΣΥΤΙ σε μια ε, αγορά ε, τεράστια χρηματοοικονομική, η οποία θα την κάνει να μοιάζει περισσότερο με φορολογική παράδοση παράδεισο από ό,τι και σήμερα. Ευχαριστούμε για την ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση προς την κυρία Μπάρσμα που γνωρίζει τις Ολλανδο-Βρετανικές εμπορικές σχέσεις. Και ε, μιλήσατε για το τελωνιακό καθεστώς. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν μίλησε για τελωνιακή ένωση. Βεβαίως υπάρχει το θέμα των συνόρων στην Ιρλανδία και το τι θα γίνει με το εμπόριο. Οι Βρετανικές επιχειρήσεις και τα συνδικάτα αντέδρασαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Θα ήθελα όμως να ακούσω εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα βασικό στατιστικό στοιχείο για τη συζήτηση που δεν τα ακούμε ποτέ. Ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πέρσι είχε 96 δι στερλίνε έλλειμμα στα αγαθά, στο εμπορικό του σωζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο μιλάει για 300 δις στερλίνες, δηλαδή το σύνολο όλων των εξαγωγών το Ηνωμένου Βασιλείου σε αγαθά. Επειδή λοιπόν είναι τελείως ε, τρομακτικές αυτές οι προβλέψεις ότι μπορεί να πάψει το εμπόριο θα ήταν προ όφελο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχιστεί το εμπόριο, διότι έχουν ένα τεράστιο πλεόνασμα. Και εάν ε, συνεχίσουμε, καλό θα ήταν να κρατήσουμε ζωντανό το εμπόριο. Επίση, να πω το εξή, ότι είμαστε σε μια επιτροπή εξαίρετη, με εξαίρετο πρόεδρο και συναδέλφου. Και συζητάμε διαρκώ εμπορικέ συμφωνίε. Είναι πολύ, πολύ εύκολο όμω να ξεχνάμε ότι δεν χρειάζεται εμπορική συμφωνία για να γίνει εμπόριο, για να υπάρξει εμπόριο. Είναι σαφές ότι οι τρεις μεγαλύτεροι εξαγωγείς των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών κρατών ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κίνα, η ΕΠΑ η Ρωσία δεν έχουν εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κοιτάζω και του συναδέλφους μου προς τα αριστερά, που είναι και πολύ καλή πολιτική, δεν θα χρειαστούν κιόλα από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει εμποδιστεί το εμπόριο. Νομίζω η πιο ενδιαφέρουσα συνεισφορά Δεν ήταν αυτή η πολύ υποκειμενική και συγκινητική προσωπική τοποθέτηση της κυρίας Αντισκοτία για τα πολιτικά της του Ηνωμένου Βασιλείου. Νομίζω ότι υποτιμάται το γεγονός ότι αν θέλει κανείς να αγοράσει και να εξάγει θα το κάνει. Εάν θέλει κανείς σκοτσέζικο ίσκι θα τα αγοράσει ούτως ή άλλως. Ασχέτως ε, ποιες είναι οι νομικές ε, συμφωνίες. Αλλά ίσως να σχολιάσετε πάνω σε αυτό. Ναι, το ίσκι είναι και αυτό καλό και παλού. Ναι, να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για αυτήν την εντατική συζήτηση γιατί υπάρχει βεβαίως και το θέμα της συνεργασίας μεταξύ της ε, Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμένα θα με ενδιαφέρε περισσότερο η εσωτερική πολιτική κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία γιατί βεβαίως ε, η σύμβαση την οποία αναζητούμε εδώ πέρα θα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Παράδειγμα του χάνει. Αν δούμε την Ιρλανδία, όπου είναι πιθανό να προκύψει ένα νέο πρόβλημα και να γίνει εκεί άλλο δημοψήφισμα Ιρλανδικό. Γιατί μπορεί να θέλουν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σκοτία έχει το δικαίωμα ε, να έχει αντίρρηση σε αλλαγές ε, στο Σύνταγμα. Ε, και βεβαίως βλέποντας ότι και το Γιβραλτάρ είχε ψηφίσει κατά μεγάλη πλειοψηφία να παραμείνει και εκμεταλλεύεται το καθεστώς της Ένωσης. Ποιε πιθανότητε θα υπήρχαν ε, να παραμείνει η Ιρλανδία στην Ένωση ή παραδείγματος χάρη να ασκήσει κάποιο βέτο η παραδείγματο χαρη να ασκησει καποιο βετο η σκοτια στην ε, συνθήκη. Τι βεβαίω ε, και για εμάς το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα σκληρό Brexit. Γιατί αν δεν υπάρξει συμφωνία στην Μεγάλη Βρετανία, είναι ακόμη πιο απίθανο να υπάρξει συμφωνία εντός ε, της ε, Μεγάλης Βρετανίας και αν ακολουθηθούν διαφορετικοί δρόμοι, ποια απάντηση θα μπορούσαμε να δώσουμε για μια λογική οικονομική σχέση στο εσωτερικό της Βρετανίας. Αυτό με ενδιαφέρει. Σας ευχαριστώ. Και τέλος είμαι. Είμαι Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι που καθυστέρησα αλλά ήταν αδύνατο να έρχω γέρος. Θα ήθελα να κάνω δύο συγκεκριμένε ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το πώς ε, τίθεται ε, το θέμα των διαφόρων διαφορών που μπορεί να προκύψουν μεταξύ Ευρωπαίων και Βρετανών επιχειρηματιών στη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου, διότι είναι μια περίοδος αβεβαιότητας και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ ε, αυτών σε αυτή την περίοδο. Δεύτερον, συνεργασία σε θέματα εναέριων μεταφορών και ασφάλειας των αερομεταφορών. Υπάρχουν αεροπορικέ εταιρείε που τώρα είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, πετούν στον Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο. Ε, πώς σκοπεύει να γίνει η μετάβαση αυτών των επιχειρήσεων, των εταιριών. Πάρα πολλέ ενδιαφέρουσε ερωτήσει και ανυπομονώ να ακούσω τι απαντήσει των εμπειρογνωμόνων. Θα τους δώσω δύο λεπτά για να μας πούνε τα βασικά. Παρακαλώ. Η Μπάρμπαρα Πάσμα πρώτα. Δεν ε, είπαμε ποιος θα απαντήσει τι, επομένως θα απαντήσω εγώ σε κάποιους και θα αφήσω και περιθώριο για τους υπόλοιπους να δώσουν απαντήσεις. Τι πιστεύετε, ρώτησε κάποιο, ποιο είναι το καλύτερο σενάριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, όχι για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Και νομίζω ότι αυτή η μεταβατική περίοδο ε, είναι πάρα πολύ σημαντική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί ουσιαστικά κερδίζουν όλοι χρόνο για να ξέρουν τι ακριβώς χρειάζονται ε, και τι θέλουν να αποκομίσουν από αυτό. Διότι κάθε πλευρά έχει διαφορετική άποψη, διαφορετική τακτική και στρατηγική. Ε, το να εξαγοράσουν όλοι λοιπόν λίγο χρόνο, ε, ναι μεν αυξάνει την αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, που πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα κατά την άποψή μου, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτός ο επιπλέον χρόνος ε, να βοηθήσει να σταθεροποιηθεί λίγο ε, καλύτερη πολιτική κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνεται διαπραγμάτευση με έναν εταίρο ο οποίος ε, που είναι τόσο αβέβαιος για το ίδιο του το μέλλον. Και Εν τέλει αυτό θα βοηθήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω λοιπόν η μεταβατική περίοδος ε, να βοηθήσει να ε, διασφαλίσουμε ότι είναι πιο σταθερό εταίρο το Ηνωμένο Βασίλειο για τη διαπραγμάτευση. Όπω σα είπα εν τέλει το καλύτερο σενάριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι το πιο ήπιο Brexit διότι ούτως ή άλλο η αλλω η Ένωση βασίζεται στο ελεύθερο εμπόριο και νομίζω ότι θα πρέπει όταν κάποιος αποχωρεί θα πρέπει να τηρούνται αυτά τα πράγματα. Επόμενη ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληγεί τόσο πολύ από το Brexit, ε, ακόμα και 2% στο 2024, διότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες λόγω του Brexit για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύντομη απάντηση είναι ότι αν πάρουμε το παράδειγμα των κάτω χωρών, για παράδειγμα, ε, διότι δεν υπάρχει ίσως εξάρτηση από το Ηνωμένο Βασίλειο στις εξαγωγές ε, συνολικά, αλλά υπάρχουν κάποιες χώρες, όχι μόνο οι κατοχώρες, αλλά και η Ισπανία, οι άλλες χώρες που εξαρτώνται πάρα πολύ από τις εξαγωγές ε, ε, προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι χώρες λοιπόν θα επηρεαστούν σίγουρα και για τις κάτω χώρες υπολογίζουμε ότι σε ένα σενάριο ε, σκληρού Brexit οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές για τις κάτω χώρες και αυτό δεν είναι μόνο ε, συνέπεια των λιγότερων άμεσων εμπορικών σχέσεων αλλά και η πολύ ψηλού πληθωρισμού εισαγωγών και αυτό φυσικά θα επηρεάσει και την κατανάλωση και αυτό ισχύει και για άλλες χώρες Γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε μεν μόνιμη ζημία, αλλά τουλάχιστον μεταβατική ζημία ε, του 20% μέχρι το 2024 για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες χώρες όπως οι κατοχώρε, θα επηρεαστούν πολύ περισσότερο. Μπορεί να φτάσουμε και το 25% στην περίπτωση του σκληρού Brexit. Μετά. Να βρω και πού το έχω σημειώσει στα χαρτιά μου. η αλλαγή της στήριξης της Τελωνιακής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι λογικό. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικό εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου και πιστεύω ότι μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να βοηθήσει να μην έχουμε σκληρά σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αλλά το ερώτημα δεν είναι αν είναι λογικό. Ε, αλλά κατά πόσον υπάρχει πολιτικό περιθώριο στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια τέτοια λύση. Και τώρα να αφήσω το λόγο στους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Να περάσουμε απευθεία στην Κέρστη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι για το τι θα γίνει, ποιο θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί, φαίνεται ότι πηγαίνουμε προς κάποιο είδους συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα πάει αυτό και τι θα γίνει με τις δεσμεύσεις να παραμείνει ανοιχτό το σύνορο της Ιρλανδίας. Δυσκολεύομαι να σκεφτώ πώς θα τραγωνιστεί αυτός ο κύκλος. Για την λύση του ΠΟΕ για το αν θα υπάρξει συμφωνία τύπου Καναδά και τα δύο θα είναι οικονομικά επιζήμια και λέω ότι το καλύτερο είναι ένα ήπιο Brexit. Αλλά κατά τα άλλα το ήπιο Brexit δεν έχει κανένα νόημα από το, σε σύγκριση με το να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διατηρηθεί το status quo. Για κάποιες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν για τις επιδείς, επιδόσεις, για τις υπηρεσίες του εμπόριου από την Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι σημαντικό είναι να θυμόμαστε τις εκτιμήσεις από το Εθνικό Ινστιτούτο για τις Στατιστικές Έρευνες του Ηνωμένου Βασιλείου για την επιλογή του ΠΟΕ και τις... τη μείωση 69% στις συναλλαγές που μπορούν να υπάρξουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι τεράστια ζημιά για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ενδεχομένως ε, μπορεί να ωφεληθεί πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πολύ δύσκολο τα μοντέλα αυτά να φωτογραφίσουν το τι θα συμβεί. Δεν έχουμε ξαναδεί να εκτελήσεται άλλου είδου ε, διαπραγμάτευση τέτοιου τύπου η απομάκρυνση στο παρελθόν. Και το τι θα γίνει με την παραγωγή, τα αγαθά. Την... Υπάρχει και μια μελέτη από το CDP που λέει για 60% μείωση και 6% μείωση με τα μοντέλα τα στατικά. Ως προς τα θεσμικά ζητήματα εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι έχει αποκεντρώσει τις εξουσίες ε, το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκοτία, δεν έχει δοθεί αρκετή πολιτική προσοχή στο ότι δύο από αυτέ τι περιοχέ, η Βόρεια Ιρλανδία και η Σκοτία, ψήφισαν υπέρ τη παραμονή τώρα. Εάν ε, η Σκοτσέζικη Βουλή περάσει το νόμο για την συνέχεια των ε, συμφωνιών ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί το Westminster να παρέμβει και να πει ότι υπερέχει δική του νομοθεσία ή να πάμε δικαστήριο. Μοιάζει με εμφύλιο πόλεμο αυτό που συμβαίνει, έστω και φιλιρινικό. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να μην δούμε τι θα κάνουν οι πολιτικοί. Έχουν ζωτικό ρόλο εδώ και για την ερώτησή σας, μια σχήμα από τη Σκωτία και μου είπατε για το ουίσκι. Όταν μελετάει κανείς ε, οικονομία δεν ξεχνάει ότι οι φραγμοί, οι δασμολογικοί φραγμοί ανεβάζουν τις τιμές. Αυτό είναι το πιο απλό που μπορώ να πω. Ευχαριστώ με μια ανάσα. για το ερώτημα του David Martin για τους ε, κανόνες προέλευσης εάν ανταγωνιστής ε, παραπονιόταν επειδή ξέρω εγώ η Κορέα συνέχιζε να παρέχει προτιμησιακό καθεστώς ε, στον Ηνωμένο Βασίλειο παρά το ότι δεν είναι πια μέλος του Ηνωμένου δεν ξέρω αν θα δημιουργούσε προβλήματα. Το αλλά δεν νομίζω να γίνει ζήτημα στον ε, ΠΟΕ, γιατί ο χρόνος που θα χρειαζόταν για να επιληθεί αυτή η διαμάχη ε, θα ξεπερνούσε την μεταβατική περίοδο, οπότε δεν συμφέρει κανέναν. Ε, μιλήσατε για το μίνι, το αυτοκίνητο. Εγώ θα έδινα ένα άλλο παράδειγμα ένας κατασκευαστής που παράγει τη μηχανή στο Ηνωμένο Βασίλειο και την στέλνει στην Νότια Αφρική για να μπει στο ΣΑΣΥ και επανέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει της συμφωνίας με την Νότια Αφρική. Αυτό γίνεται μόνο γιατί υπάρχει το καθεστώς που, της όρευσης που θεωρεί κοινοτικό το προϊόν του Ηνωμένου Βασιλείου. Μου είπατε να αποκαλύψω τις πηγές μου. Ε, το πρώτο το οποίο θα έλεγα είναι ότι είμαι πεπισμένο πως πολλές χώρες θα προσπαθήσουν να κάνουν λίγη υπαγορά, γιατί θα ήταν αμέλεια να μην το κάνουν, εάν είναι προς το εθνικό τους συμφέρον να λάβουν κάποιε παραχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο την στιγμή που μπορούν, θα προσπαθήσουν να το κάνουν. Ε, υπάρχουν άλλε χώρε που έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα δυσκολεύσουν τα πράγματα Γνωρίζουμε για την Κορέα γιατί έχει αναφερθεί πολλές φορές στον Telegraph και γνωρίζω επίσης πως ε, παραπονιούνται γιατί έχω κάποιες πηγές στην κυβέρνηση που δεν θα τις ε, ε, αποκαλύψω για την Νότια Αφρική. Επίσης το έχουν γράψει και οι Times. Ένας πρέσβης είπε στους Times ότι θα αναζητήσουν υψηλότερους δασμούς από το Ινωμένο Βασίλειο και άλλες παραχωρήσεις τι θα κάνουν τώρα, γιατί η νέα προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου τέθη ενισχύ μόνο ε, την Δευτέρα. Οπότε θα δούμε το τι θα γίνει. Αλλά όπως είπε και ο Νικολάη υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με το ζήτημα ότι οι ειδοποιήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταλούν αργά τελευταία στιγμή, οπότε μέχρι τότε θα υπάρχει βεβαιότητα. για τις ε, σχέσεις με τη Νέα Ζηλανδία. Ε, κοιτάξτε, επειδή θα δεσμεύεται ακόμα το Ηνωμένο Βασίλειο, η συμφωνία αυτή με την ε, Νέα Ζηλανδία για τις ποσοστώσεις για τα πρόβια θα εξακολουθήσει να ισχύει. Λοιπόν, για το θέμα με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες που εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το ότι δεν έχουν εμπορική συμφωνία. Δεν ισχύει ακριβώς. Έχουμε τέτοιες συμφωνίες με την Κίνα, έχουμε συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης ε, για τις εταιρείε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 7 συμφωνίες με τις ΗΠΑ για το εμπόριο, για βιολογικά τρόφιμα και 6 άλλους κλάδους. Οπότε, ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται μια γενική εμπορική συμφωνία, αλλά ε, δεν ε, ισχύει το ότι δεν υπάρχουν συμφωνίες αυτή τη στιγμή. Κάτι τελευταίο. Σκοτσέζικο ισχύει. αγοράζουμε ε, ακόμα και αν υπάρχουν δασμοί. Αλλά υπάρχει λόγος που θέλουν να καταργήσουν τον δασμό 150% στην Ινδία. Γιατί θεωρούν ότι θα πουλήσουν περισσότερο ή όταν πέφτουν οι δασμοί, εντάξει μπορεί να μην επωφελείται 100% ο αλλά οπωσδήποτε δεν ανεβαίνει η τιμή. Ναι, πράγματι. Ο Νικολάη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Σκωτία, δεν θα σας πω τίποτα για το σκοτσέζικο whisky λοιπόν και θα σταθώ σε κάποιες ερωτήσεις ε, στην παρέμβασή μου. Καταρχάς, για τα διάφορα σενάρια, θέσατε δύο διαφορετικές ερωτήσεις, πολύ διαφορετικές. Ποιο πιστεύουμε ότι είναι πιο πιθανό και είναι πιο επιθυμητό να συμβεί. Ε, να πω ότι το πιο πιθανό, η πιο πιθανή πορεία που θα ακολουθήσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο ε, Βασίλειο είναι μια συμφωνία εταιρική σχέση ε, με μια συνιστό ελευθέρου εμπορίου και ε, κάποια άλλα θέματα συνεργασία, άμυνα κλπ. Αλλά κυρίω ε, θα έχουμε συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Προσωπικά, Όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, ε, εάν υπάρχει λόγος να υπάρχει τελωνιακή ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό θα το επιθυμούσαν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αυτό φυσικά ε, εξαρτάται και από τις εσωτερικές συζητήσεις του Ηνωμένο Βασίλειου. Τώρα, όσον αφορά τους κανόνες προέλευσης και τι πρόβλημα μπορεί να υπάρξει, ε, όταν ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν την εντοπιότητα του προϊόντος τελικά ε, αυτό θα εξαρτάται από τι αποφάσει που θα λαμβάνει κάθε επιχείρηση ατομικά. Ε, ποιο θα είναι το κόστο τη γραφειοκρατίας και των πιθανών δασμών ναι, και κατά πόσον αυτό ε, αξίζει να γίνει με την κατάσταση τη αλυσίδα προμηθειών ή αν θεωρούν να, ότι μπορούν να επιστρέψουν το κόστο στον πελάτη και να προσπαθήσουν να εξοικονομήσουν απαλού. Έγινε μια μελέτη για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. δεν έχω τα ακριβά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι είχαμε περίπου 15 με 20% επιχειρήσεων που ήδη κάνουν αλλαγή και ε, πιστεύω ότι ο καθένας θα λαμβάνει απόφαση ανεπιχείρηση. Δεν θα υπάρξει μια μεγάλη κίνηση κατάσταση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σιγά σιγά οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, ε, η αβεβαιότητα και το πώς χρησιμοποιείται κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για να πιέσει για τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι και από τις δύο πλευρές είδαμε ότι οι διαπραγματεύσεις ε, ε, εξαρτώνται από τα πολιτικά και όχι από τα οικονομικά συμφέροντα και ο τρόπος με τον οποίο θα διαρθρωθούν θα φανεί ε, μόνο στο τέλος και σημαίνει ότι η αβεβαιότητα θα είναι πολύ υψηλή σίγουρα μέχρι να υπάρξει υπογραφή και κύρωση της συμφωνίας αποχώρησης και νομίζω ότι η αβεβαιότητα έρχεται και από τις δύο πλευράς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί συνδέει τα δύο θέματα αλλά και από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου διότι υπάρχει μια πολιτική αβεβαιότητα για το κατά πόσο θα κυρωθεί και θα γίνει πλήρω αποδεκτή η συμφωνία αποχώρησης από το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέταρτον και τελευταίον. Όσον αφορά τι αεροπορικέ εταιρείε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση, γιατί σχετίζεται και με μια συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι απαραίτητο μόνο σε θέματα εμπορίου. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της μετάβασης ε, η αεροπορία εντός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νέας Αγοράς δεν πλήττεται γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει, επομένως θα συμμετέχει και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, πολιτικής αεροπορίας, θα αλλάξει όμως η σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και τρίτων χωρών. Και από τα τύπο διαβάζουμε ήδη ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν τονίσει το θέμα και έχουν απειλήσει να ε, προσφέρουν χειρότερη ε, πρόσβαση οι επιχειρήσεις αεροπορικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου από ό,τι έχουν οι ε, αεροπορικέ εταιρείε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να τονίσουν οι αεροπορικέ εταιρείε και πολύ δύσκολο το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρήσει την πρόσβαση που έχει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μια γενική λοιπόν εικόνα. Καταλάβαμε ποιες θα είναι οι βασικές δυσκολίες στην περίοδο μετάβασης και τώρα το ερώτημα είναι πώς θα διαμορφωθεί η σχέση μετά τη μεταβατική περίοδο. Ε, εμπορικές συμφωνίες ή τα μετρία συν, τρεις φορές καλύτερη. Πώς θα διαμορφωθεί αυτή η σχέση και με το τελωνιακό καθεστώς. Τι θα ισχύει. Έχουμε και άλλους πολύ έμπειρους ε, εμπειρογνώμονες για να μας πούν κάποια σχόλια για τις μελλοντικές σχέσεις και τη μορφή θα πάρουν. Πρώτα απ' όλα ο Στέφανο Ινάμα από την Jungtad που είναι ε, εμπειρογνώμων για τον ΟΗΕ στο τμήμα εμπορίου και ανάπτυξης. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να σας αναφέρω κάποια από τα πράγματα που ξέρουμε από το τι κάνουν οι χώρες με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Για το Brexit μου ζητήθηκε να σας δώσω κάποιες ε, σκέψεις μου για το τι πιστεύουμε θα είναι το μέλλον των εμπορικών σχέσεων. Μεταβατική περίοδος. Το Ηνωμένο Βασίλειο λογικά θα φύγει από την ενιαία αγορά και την Πολωνιακή Ένωση. Άρα θα αλλάξουν και σχέσεις του με τι τρίτε χώρες. Δεν θα έχει άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώ θα διαμορφώνονται αυτές. Το ερώτημα είναι λοιπόν το ερώτημα τι οικονομικούς χώρους μπορεί να διαμορφώσουν το Ηνωμένο Βασίλειο με τρίτες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες μετά την μεταβατική περίοδο εντόπισα τα απλούστερα θέματα, ακόμη και αν φαίνονται πάρα πολύ ε, δύσκολα. Ε, η εξάλληψη των δασμών και οι κανόνες για την προέλευση των προϊόντων. Οι προηγούμενοι ομιλητές ήδη έδωσαν κάποιες ε, ιδέες για το πώς θα διαμορφωθούν αυτοί οι εμπορικοί χώροι. Υπάρχει το ήπιο μοντέλο υπάρχει η συμφωνία τύπου ΠΟΕ ή με συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών όπως με την Ελβετία ή αυτές του οικονομικού, ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ή η Ευρωπαϊκή Περιοχή Ελεύθερων Συναλλαγών. Όλες αυτές θα μπορούσαν να ισχύσουν διευθετώντας και ρυθμίζοντας την σχέση ελεύθερων συναλλαγών Ηνωμένου Βασιλείου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι ποιο θα είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής και πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με τις τρίτες χώρες. Θα επαναλάβει απλώς, θα αντιγράψει φωτοτυπικά τις συμφωνίες που είχε όταν ήταν μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες αυτές, με τους εμπορικού τετέρους ή θα δώσει διαφορετικό περιεχόμενο, διαφορετικό νόημα στις μελλοντικέ ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Γνωρίζουμε περί λίγο πολύ τι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Ηνωμένο Βασίλειο ως προς τους κανόνες προέλευσης. κανόνες προέλευσης, αλλά με προστασία για τη γεωργία και την αλία και πιο ελεύθερα στη μηχανική και τα ηλεκτρονικά. Και βεβαίως και στην αυτοκινητοβιομηχανία ρωτιούνται όλοι πώς θα δημορφωθούν οι σχέσεις, επειδή είναι εντατικότατες οι σχέσεις εμπορικές ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Βασιλείου. Το θέμα είναι ότι θα υπάρχει σώρευση των κανόνων προέλευσης η ισόρρευση μπορεί να λύσει κάποια από τα προβλήματα, όμως υπάρχουν και όροι που πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα. Πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες περί προέλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν θα διαπραγματευτεί με τρίτες χώρες και τις εταίρους από εκεί μετά τη λήξη της μεταβατικής περίοδου θα διαπραγματευτεί τις συμφωνίες ελεύθερου συναλλαγών με τους ακριβώς ίδιους πανομοιωτικού κανόνε κανόνες προέλευσης όπως όταν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα ισχύσει η σώρευση των κανόνων προέλευσης βάσει των όσων ισχύουν και στην Γενική Διεύθυνση Trade. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Επίσης μια άλλη πτυχή πρέπει να σκεφτεί κανείς είναι οι συνέπειες στις εμπορικές ροές. Εδώ, για περάστε στο επόμενο. Εδώ πήραν το πιο φιλόδοξο, το πιο αισιόδοξο σενάριο, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ε, διαπραγματεύεται συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες ταυτόχρονα. Αυτό θα ισχύει τηρουμένο των αναλογιών και για τις άλλες 50 συμφωνίες που έχουμε με τους τωρινούς εταίρους. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο ε, με τους Αμερικανούς εταίρους τους κανόνες προέλευσης, μπορεί να είναι πιο φιλελεύθεροι, πιο ε, διαλεκτική εκεί μπορεί να υπάρξει μία Εκεί μπορεί όπως με το αλουμίνιο λόγω χάρη να υπάρχουν δασμοί 3%. Αλλά για ένα αυτοκίνητο ας πούμε, το οποίο κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά μετά επανεξάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί δεν θα υπάρχουν δασμοί, θα είναι duty free. Εδώ λοιπόν οι κανόνε προέλευση ισχύουν διαφορετικά. Σε το είδο τη συμφωνία, πόσο θα κοστίσει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο διοικητικό σύστημα ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση στα εμπορικά. Έπειτα το θέμα της σόρευσης. Το θέμα της σόρευσης μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα υπό τον όρο όμω, ιδίω στι σχέσει με του Αμερικανού, ότι ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση διπλωματεύεται έναν τέτοιο χώρο ελεύθερων συναλλαγών με, το Ενωμένο, με τι ΗΠΑ. Με του ίδιου κανόνε προέλευση όπω και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτή την περίπτωση η ισόρρευση θα μπορεί να γίνει. Όμως Το θέμα είναι ποιε προποθέσει θα ισχύουν ταυτόχρονα. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει ότι το Μένο Βασίλειο διαπραγματεύεται με τι ΗΠΑ. Ένα σύνολο κανόνων προέλευση που είναι πανομοιότυπο με αυτό το σύνολο κανόνων προέλευση που είχε διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τι ΗΠΑ. Αυτά για να σας δώσω μιας, κάποιες πρώτες ιδέες για το πόσο περίπλοκος είναι ο κατάλογος των προτεραιοτήτων που θα πρέπει να συζητήσετε. Μόνο και μόνο για τους δασμούς και τους κανόνες προέλευσης και όχι όλα τα υπόλοιπα. Όπως έλεγα, η σώρευση θα ισχύσει αν υπάρχουν πανομοιότυποι κανόνες προέλευσης. Για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά τους υπάρχει μια πολύ φορτωμένη ατζέντα. Είναι πανομοιότυποι κανόνες προέλευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες προέλευσης, η σώρευση πώς θα ισχύει, ανατομέα. Θα του έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα σύνολο κανόνων προέλευση και σώρευση για την αυτοκινητοβιομηχανία μόνο και να ισχύει μόνο για αυτό το κλάδο. Και όλοι οι ευάλωτοι τομεί να έχουν την ίδια μεταχείριση. Η αλληλεία, τα κλωστεφοντουργικά. Και επειδή έχουν κοινά εμπορικά συμφέροντα εκεί, μπορεί να είναι άλλοι τομεί που να διευθετηθούν διαφορετικά. Άλλο θέμα είναι να επιτραπεί ισόρευση στις νέες συμφωνίες, ακόμη και αν δεν είναι πανομοιότυποι κανόνες προέλευσης. Αυτή είναι μια νέα ε, αντίληψη, την οποία δεν έχουμε εφαρμόσει ποτέ ως τώρα, αλλά θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε όπως και στα πλαίσια της οικονομικής συνεργασίας με τις χώρες ΑΖΕΑΝ, του Νότιου Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος ε, εφόσον ασχολούμαστε με την ανάπτυξη και το εμπόριο σε τι σχέση θα έχει το Ηνωμένο Βασίλειο με τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε και τι αναπτυσσόμενε. και πώς θα ισχύει το πρωτομησιακό σύστημα, το σύστημα πρωτομησιακών δασμών. Πριν από ένα χρόνο, ένας ε, ηθήνων από το Ηνωμένο Βασίλειο με ρώτησε ποιοι είναι οι βέλτιστοι κανόνε για την περίπτωση αυτή και μια ένα παράδειγμα που το, το έδωσε ήταν οι κανόνες προέλευση στη, σχέση, στη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά ε, μετά την ε, σύναψη τη συμφωνία. Μου είπε, εμεί θέλουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Ωραία να, κάτι, να κάνετε κάτι καλύτερα, εφόσον όμω αυτό θα μπορεί να γίνει μόνο εφόσον οι ίδιοι κανόνε προέλευση ισχύουν στη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλιώ η σώρευση δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, πόσο σημαντική είναι η σχέση αυτή είναι ένα άλλο θέμα που προκύπτει, αλλά είναι πιο εύκολο ενδεχομένω να έχουμε μηδενική σώρευση αλλά περισσότερο φιλελεύθερου εμπορικού κανόνε. Θα φανεί αυτό. Θα φανεί γιατί δεν μπορεί κανεί να λάβει τεκμηρωμένη απόφαση τώρα. Ολοκληρώνοντα, θα μπορούσα να διατυπώσω ερωτήσει περισσότερο. Γιατί εγώ κυρίω δίνω συμβουλευτικέ υπηρεσίε σε χώρε στι εμπορικέ του διαπραγματεύσει και κάποια από τα ερωτήματα μπορεί να ανακύψουν εδώ είναι ερωτήματα μπορούμε απλώς να θέσουμε και να σκεφτούμε μελέτες που έχουν ήδη γίνει για τον οικονομικό αντίκτυπο του Brexit λόγου χάρη, αλλά ακόμα λείπουν μελέτες που να, να προτείνουν λύσεις. Λύσεις για να εφαρμοστούν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ή να λυθεί το πρόβλημα τη σώρευσης των κανόνων πρόέλευση είναι να έχουμε του καλύτερου κανόνε προέλευση, ώστε η αλυσίδα, η εμπορική να προφυλαχθεί, να μην υπάρξουν διακοπές και αναταραχές για τις εταιρείε. Ένας τρόπος να γίνει αυτό είναι να δημιουργήσουμε ένα μητρό ε, εισρώων και εκροών, να δούμε τι εισάγει και τι εξάγει δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο να πάρουμε τα επεξεργασμένα και μη προϊόντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιστρόφως, αλλά υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εδώ. Θα έλεγα ότι χρειάζεται ένας υψηλός βαθμός ακρίβειας για να καθορίσουμε τους καλύτερους κανόνες προέλευσης που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να χρησιμοποιηθούν στις νέες εμπορικές συμφωνίες. Και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον Ηνωμένο Βασίλειο. και μάλιστα το νωρίτερο Όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε αυτές τις μελέτες, τόσο πιο εύκολο θα είναι να λάβει κανείς μια απόφαση, η οποία να βασίζεται σε στοιχεία τεκμηριωμένα. Και ιδίω σε αυτό το στάδιο εξέλιξης των εμπορικών σχέσεων διεθνώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η επιλογή μιας, ε, ενός χώρου ελευθεροπορίου με τις είπα δεν ξέρω, με κάνει λίγο επιφυλακτικό. Έχω περάσει πολύ καιρό στις διαπραγματεύσεις με το TTIP, ας μείνουμε στο σημερινό μας θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Ρόμπερτσον τώρα είναι εκπρόσωπος ε, του ομίλου BMW στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μεγάλη παρουσία στο Ενωμένο Βασίλειο, όπως αναφέρθηκε. Κατασκευάζουμε το μήνυ. Εκατοντάδες χιλιάδες κινητήρες που εξάγονται στα εργοστάσια μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εκεί πέρα βεβαίως έχουμε δύο εταιρείες μας, η Μίνη και την Rolls Royce. Συνολικά έχουμε 8.000 ε, άμεσους ε, υπαλλήλου ε, και στηρίζουμε 5.000 θέσει εργασία στη δουλειά. Το βασικότερο κομμάτι είναι ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιομηχανίας. Δηλαδή είτε οι κινητήρες πηγαίνουν από το ένα εργοστάσιο στο άλλο ή πηγαίνουν εξαρτήματα στον Αμενό Βασίλειο και συναρμολογούνται ή πάνε από την Οξφόρδη στην Ολλανδία, τα Μίνι ή αλλού στον κόσμο, έχουμε μια ολοκληρωμένη αλυσίδα που έχει αναπτυχθεί εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε χαρακτηριστική περίπτωση και οι άλλες εταιρείε έτσι κάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατασκευάζονται γύρω στο 1,6 εκατομμύρια αυτοκίνητα το έτος και μεγάλο ποσοστό εξάγεται στην Ευρώπη και ε, μικρότερο ποσοστό στον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε από την σκοπιά του ότι συνεισφέρουμε στην Βρετανική οικονομία αλλά και στις Βρετανικές εξαγωγές έχουμε πολλές ροές ε, που αφορούν ε, τα πάντα να σας πω κάποια πρακτικά πράγματα. Κάθε μέρα έχουμε γύρω στα 260 φορτηγά που έρχονται και βγαίνουν από την χώρα για λογαριασμό μας και έχουν βεβαίως μια ανεμπόδιστη ροή, ακολουθούμε μια μεθοδολογία just in time με την έννοια ότι δεν έχουμε μεγάλα αποθέματα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ή αποθέματα αυτοκινήτων επίσης. Επίσης βλέπετε εκεί κάποια από τα δεδομένα Βεβαίω. Έχουμε αυτοκίνητα που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, πέρα από το ότι εξάγουμε μήνυ σε μεγάλους αριθμούς. Βλέπετε από τα 3 εκατομμύρια που έχουμε φτιάξει τα τελευταία 15 χρόνια, γύρω στα 2 εκατομμύρια έχουν εξαχθεί. Και κάθε μέρα δύο τρένα φεύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο γεμάτα για την ε, Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, όπως και πολλά άλλα ε, εξαρτήματα των αυτοκινήτων. Οπότε έχουμε μια ολοκληρωμένη αλυσίδα παραγωγής και είμαστε αντιπροσωπευτικοί θα έλεγα της αυτοκινητοβιομηχανίας του Ηρωμένου Βασιλείου. Επόμενη διαφάνεια. Και άλλη μια, να, μια ωραία εικόνα. Αυτή την διαφάνεια την έκανα γιατί την τελευταία ώρα ακούσαμε αρκετά για τα κράτη-μέλη και τον ΠΟΕ. Ε, σαφώς βεβαίως εδώ πέρα έχουμε ε, μόνο διαβαθμίσεις ε, της ζημίας. Δηλαδή ξεκινάμε από την καταπράσινη σειρά που είναι κράτος μέλος και όσο πάμε κάτω κοκκινίζει. Λοιπόν, υπάρχουν διαφορές προτάσεις για το τι είναι καλύτερο, γίνεται λόγος για ενιαία αγορά, συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, τελωνιακή ένωση. Ε, Ένα ειλικρινά σας λέω δεν με ενδιαφέρει πώς τα λέγεται. Εμείς έχουμε κάποιες απαιτήσει για να λειτουργεί η κατασκευή και οι πωλήσει και να λειτουργούν ομαλά και τα στοιχεία βεβαίως που βλέπετε στο πάνω μέρος της διαφάνειας είναι αυτά τα οποία χρειάζονται για επιτυχημένες επιχειρήσεις. Το άλλο θέμα που ετέθη είναι γιατί θα πρέπει να ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπα, υπάρχουν πολλά κομμάτια που διασχίζουν ε, σύνορα, ολοκληρωμένα αγαθά. Υπάρχουν εργοστάσια στην Ευρώπη που εξαρτώνται από εργοστάσια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε αυτά τα εξαρτήματα, αν ε, έχουν δυσκολία στο να μπουν ε, στην ε, Βρετανία, ακριβώ την ίδια δυσκολία θα έχουν για να μπουν μετά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα έχουμε προβλήματα και στις δύο όχθες της μάχη, εάν έχουμε μια πιο δύσκολη συμφωνία, όσο πιο κάτω πάμε δηλαδή εδώ πέρα στον κατάλογο. Και ανησυχώ ιδιαίτερος ότι υπάρχει αίσθηση ότι μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου είναι η απάντηση σε πολλά από τα προβλήματα ε, στην πραγματικότητα δεν είναι πολύ καλύτερη από μια συμφωνία τύπου γιατί θα υπάρχουν τελωνιακοί έλεγχοι, διοικητικά ζητήματα, καθυστερήσει στα σύνορα, ε, ζητήματα τοπικής ε, παραγωγής και πρέλευσης και ζητήματα βεβαίως ρύθμισης. Οπότε, όσο περισσότερο αντιλαμβάνεστε τις λεπτομέρειες και ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και εδώ πέρα στα δεξιά μου είναι η ειδική στις λεπτομέρειες εγώ απλά είμαι από το χώρο των επιχειρήσεων και από αυτήν την ε, σκοπιά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από πολιτική σκοπιά για ε, το τι θεωρούμε καλό αποτέλεσμα γιατί μπορεί να έχουμε έτσι, κάποιες ε, συνέπειες τις οποίες δεν επιθυμούσαμε στα σενάρια που ακούστηκαν την τελευταία ώρα. Οπότε Οι κίνδυνοι είναι σαφής, ε, συζητήθηκαν ήδη, είτε μιλάμε για δασμούς, ε, για το περιεχόμενο, καθυστερήσει στα σύνορα. Οι ρυθμιστικές αποκλήσεις ε, για τις οποίες δεν μιλήσαμε, εμείς θεωρούμε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να έχει ένα ενιαίο ρυθμιστικό καθεστώς, όπως μίλησε η Βρετανίδα Πρωθυπουργός για τη φαρμακοβιομηχανία και την αεροπορία και η βιομηχανία επειδή είναι παγκόσμια βιομηχανία, χρειάζεται ε, τουλάχιστον πανευρωπαϊκές προδιαγραφές όπως υπάρχουν ασιατικές και αμερικανικές. Δηλαδή το να έχουμε και άλλες προδιαγραφές ε, δεν φτάνει. Μετά έχουμε προβλήματα με την έγκριση τύπου που δεν ε, έχουν κάποια αξία για τους πελάτες μας τελικά. Οπότε το να υπάρχει μια αριθμιστική σύγκληση είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Συμπερασματικά λοιπόν. Επόμενη διαφάνεια. Οι απαιτήσει, όπως είπα, Έχουμε ορισμούς ε, και υπάρχουν ειδικοί εδώ πέρα για την διαφορά μεταξύ μιας συμφωνίας ελευθέρου και τελωνιακής ένωσης. Ε, δεν θα πω ότι τα ξέρω όλα, αλλά οι στόχοι για την αυτοκινητοβιομηχανία και την BMW προσωπώ συγκεκριμένα είναι μια αριθμιστική ευθυγράμμιση, απουσία δασμών, σύνορα χωρίς καθυστερήσεις, γιατί ε, αν έχουμε 260 φορτηγά για την BMW, έχουμε στα 2.000 φορτηγά για την αυτοκινητοβιομηχανία και 10.000 φορτηγά κάθε μέρα συνολικά από τα κύρια λιμάνια και οποιαδήποτε αναταραχή θα κοστίσει και στις δύο πλευρές. Ε, επίσης, ε, να μην Υπάρχει κάποιο αποκλεισμό λόγω του τοπικού ποσοστού παραγωγή και τα πολυτεχνικά ζητήματα που ανέφερε ο συνάδελφο εδώ στα δεξιά μου, η σώρευση των κανόνων προέλευση, ειδικά για τις ε, τρίτες ε, χώρες, είναι σημαντικό θέμα για εμάς. Και βεβαίως ε, μαζί με όλα αυτά η πρόσβαση σε εργαζόμενους και η κινητικότητα των εργαζομένων. Λοιπόν, υπάρχουν απαντήσεις για όλα αυτά, αλλά απαιτείται ένα βαθμό εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές της διαπραγμάτευσης να δούμε τις απαιτήσει ε, και να βρούμε τις πολιτικές και οικονομικές λύσεις που, όπως είπα, υπάρχουν, ε, αλλά πρέπει ακριβώ να ξεκαθαρίσουν οι λεπτομέρειε γιατί, όπως είπε και κάποιο άλλο ε, καλοδεχούμενα τα δύο χρόνια εφαρμογής, ή 21 μήνε αλλά για το υπόλοιπο του έτους ε, πρέπει να ξεκαθαρίσει το τι μορφή θα έχει η συμφωνία. Αλλιώς θα έχουμε άλλα δύο χρόνια αβεβαιότητας, ε, κάτι το οποίο δεν είναι προς το συμφέρον κανένας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας... Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω όλοι οι προβλεφτέ θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βρεθεί μια σύντομη λύση, αλλά θα θυμάστε ότι με τον Καναδά οι διαπραγματεύσει διήρχησαν 7 χρόνια. Ε, μάθαμε λίγο και εμείς ε, ελπίζω να τα κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε εδώ και τον πρόεδρο του Eurochambre, τον Κρίστοφ Λάιτελ και θα του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ήταν ε, εντυπωσιακό αυτό το παράδειγμα της ε, BMW. Η BMW ε, έχει παγκόσμια εμβέλεια και όχι μόνο στην Ευρώπη ε, και στη χώρα μου και στην ίδια μου την περιοχή ε, έχουμε κατασκευή ενός εκατομμυρίου κινητήρων για το εργοστάσιο της BMW, όχι μόνο της BMW αλλά και της BMW. Και καταλαβαίνετε λοιπόν πώς επηρεαζόμαστε όλοι. Μια κυρία στη συζήτηση ρώτησε ποιο είναι το πιο λογικό, το ποιο είναι το πιο πιθανό και ποιο είναι το πιο επιθυμητό σενάριο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εγώ. Το πιο λογικό θα ήταν να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιο πιθανό είναι μία έξοδος που δεν γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί. Και το πλέον επιθυμητό είναι να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος και να είμαστε και φίλοι ο, καθώς και εταίροι. Speaking also as Και όταν αναφέρομαι στον Ταβός, ε, αν μιλάω και ως πεπισμένος Ευρωπαίος. Είναι συναισθηματικό το ερώτημα όταν φεύγει ένα μέρος ε, της οικογένειας. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πάντα ενδιαφερόταν μόνο για την οικονομική συνεργασία. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια πολιτική, κοινωνική ή περιβαλλοντική ε, συνεργασία. Και επομένως θα πρέπει να πούμε ότι αν όντω είναι αυτή η ανάλυση, θα πρέπει να πουμε οτι αν οντως ειναι αυτη η αναλυση θα πρεπει να ε, πράξουμε και αναλόγως της ανάλυσης. βρέθηκα στο Λονδίνο και μάλιστα ε, έπεσα και πάνω σε μια διαδήλωση κατά του Brexit ενώπιον του Βρετανικού Κοινοβουλίου και κούνησα και μια ευρωπαϊκή σημαία. Ε, ήταν θέμα ε, καρδιάς για μένα, αλλά δεν αλλάζει τίποτα, είμαστε και ρεαλιστές συζήτησα με τον Υπουργό Εμπορίου και τον Υπουργό ε, Βιομηχανίας. Και πραγματικά δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν, διότι η κυβέρνηση είναι διαιρεμένη και υπάρχουν διάφορες απόψεις και η αντιπολίτευση έχει άλλη άποψη και άλλη λύση για την υπόθεση λένε απλώ ότι θέλουν να συμμετέχουν στην ενιαία αγορά, αλλά από την άλλη πρέπει να αποχωρήσουμε. Δεν θέλουν τελωνιακή ένωση, μάλλον δεν θέλουν δασμού αλλά να φύγουν από την τελωνιακή ένωση. Ε, αυτό δεν γίνεται να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει τρόπος να λειτουργήσει τέτοιο σύστημα. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα στοιχεία το 50% των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 5% των συνολικών εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει μια διαφορά, αλλά το θέμα δεν είναι ποιος θα ζημιωθεί περισσότερο. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις ζημίες, πώς μπορούμε να τις περιορίσουμε, πώς μπορούμε να αποφύγουμε δασμούς και να ε, αναζητήσουμε μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε τους μη δασμολογικούς φραγμούς. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν χρειάστηκε να ασχοληθούν με μία ε, αγορά εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν χρειάστηκε να ε, συντάξουν ποτέ, να συμπληρώσουν ποτέ τελωνιακή διασάφηση. Και πρέπει λοιπόν και εμείς να τους βοηθήσουμε. Ακούσαμε προηγουμένως ε, τα προβλήματα των μεγάλων επιχειρήσεων από τον εκπρόσωπο της BMW και εγώ έρχομαι να σας μιλήσω για τα προβλήματα των μικρών επιχειρήσεων. Επομένως, χρειαζόμαστε οικονομικές σχέσεις οι οποίες θα είναι όσο το δυνατόν στενότερες και πρέπει να γνωρίζουμε και ότι αυτό ενέχει και κάποιο κόστος. Το κόστος το γνωρίζετε και αναφέρθηκε σήμερα και από τους υπόλοιπου εμπειρογνώμονες, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω αυτά, αλλά εκατό εκατομμύρια τελωνιακές διασαφήσεις θα προκύψουν. θα είναι ετησίω, δεν θα είναι σωρευτικά. Ετησίω θα έχουμε επιπλέον 100 εκατομμύρια τελωνιακέ ε, διασαφήσει. να μην μιλήσω για πιστοποιητικά προέλευση. Υπάρχει έκθεση Τσιτσίνη η οποία λέει ότι έχουμε πάντα 5 με 10 δισεκατομμύρια ε, σε ποσά, αλλά συνδυάζεται και με ένα πρόβλημα για να δημιουργήσουμε και κατάλληλο χρόνο. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 10.000 δημοσίους υπαλλήλους για να διεκπαιρεώσουν όλες αυτές τις διασαφήσεις. Ε, είναι πολυτέλεια αυτό το πρόβλημα για την Ευρώπη και ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε λίγο αυτά τα ποσά. Και αναφέρθηκε από όλε τι πλευρέ η αβεβαιότητα. Και επομένω, καλό είναι να υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία μεν, αλλά η αβεβαιότητα δεν προσφέρει και τίποτα. Το να έχουμε μια ημερομηνία και να πούμε ότι θα έχουμε μια μεταβατική περίοδο είναι μεν κάτι, αλλά τι θα ακολουθήσει ε, και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και για του εμπορικού μα εταίρου. Συζητήθηκε το θέμα αυτό σήμερα. Οι εμπορικοί εταίροι, οι οποίοι ε, συνδέονται μαζί μα με συμφωνίε ελευθέρου συναλλαγών. Τι θα γίνει με αυτού. Κανεί δεν ξέρει και κανεί δεν μπορεί να απαντήσει. Και η πολιτική με το λαϊκισμό δεν ε, θεωρούν ότι τους απασχολεί. Όχι, δεν είναι δικό τους, είναι δικό μας ε, θέμα, πρέπει εμείς να το διαχειριστούμε. Οι επιχειρήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επομένως θεωρώ ότι είναι κρίμα, μεν, αλλά πρέπει να το διαχειριστούμε, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι διατεθειμένη να μας συνοδεύσει και να μας βοηθήσει και να βοηθήσει ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στις συνθήκες που θα προκύψουν. Και πρέπει να το κάνουμε όλοι. Και το λέω και στους φίλους του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι εδώ παρόντες σήμερα. Ελπίζουμε πραγματικά να υπάρχουν καλές σχέσεις στις επιχειρήσεις και στο μέλλον και ε, στην ευρωπαϊκή πλευρά. Ε, και εμείς ε, έχουμε αντίστοιχη αφοσίωση με εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και από τις μικρομεσαίες. Έχουμε εδώ τον Μίστερ Μικρομεσαίο ο οποίος πάντοτε προσπαθεί να επηρεάσει όλες τις συζητήσει προ όφελο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάντω, Θέλουμε να δούμε τι γίνεται και με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό έχουμε εδώ τον Λουκ Τριάγκλ, διευθυντή της Industriol. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ που προσκαλέσατε και εμάς αυτή την τόσο κέρια ακρόαση. Στη μεθεπόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Κατά πρώτον, ποιοι είμαστε. Είμαστε η Industry All της Ευρώπης, ε, μια ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους εργαζομένους ε, τις εταιρείε και τις κατασκευαστικές. Ε, είμαστε 7 εκατομμύρια εργαζόμενοι, τόσους εκπροσωπούμε μάλλον, σε όλες τις εταιρείε αυτοκινητοβιομηχανίες, φαρμακευτικές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Υπόθηκε και από προηγούμενους ομιλητές πόσο Σημαντικό είναι να κατανοήσουμε την πραγματικότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή στο εμπόριο και τι εταιρείε και πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε του στενού δεσμού και τις σχέσεις που έχουμε μεταξύ εταιρεών ε, παρασκευαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Το παράδειγμα που δόθηκε για την BMW είναι μια ε, πραγματικότητα, ε, σαφής πραγματικότητα. Όχι μόνο για την αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μπορώ να φέρω και άλλα παραδείγματα. Ένα παράδειγμα ακόμα. Στην Ευρώπη φτιάχνουμε και πολύ καλά ελικόπτερα. όμως το κουτί ταχυτήτων ενό ελικοπτέρου περνάει από τη μάχη 8 φορέ πριν καταλήξει να τοποθετηθεί σε ένα ελικόπτερο. Στα χημικά έχουμε πολλά πολλές μετακινήσεις ε, από τη μάχη ένθεν και ένθεν μέχρι κάτι να φτάσει να βγει στην αγορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα των εταιριών. Ε, πρέπει λοιπόν να το ε, υπερπηδήσουμε αυτό το εμπόδιο είναι άλλο η ιδεολογική συζήτηση και άλλο η πραγματικότητα. Το θέμα είναι τι σημαίνει να, επιβά... να αρχίσουμε να επιβάλλουμε δασμού και φραγμού, διοικητικού φραγμού, σε μια τέτοια πραγματικότητα που τη ζουν ήδη εταιρείε και όσε παρασκευάζουν προϊόντα. Είναι καθοριστική σημασία για τι ευρωπαϊκέ λοιπόν εταιρείε που παρασκευάζουν προϊόντα να παραμείνει ενιαία η αλυσίδα παραγωγής. Αλλά και το εσωτερικό εμπόριο στην ενιαία χώρα πρέπει να διαφυλαχθεί. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια ρυθμιστικής σύγκληση των δύο αγορών τώρα και στο μέλλον. Πρέπει να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση των κανόνων προέλευσης ε, και διοικητικέ ε, ελαφριέ διαδικασίε ε, πρόσβαση χωρί δασμούς και εμπόδια και άλλου φραγμούς και η ελευθερία της μετακίνησης, της κυκλοφορίας. Καλό είναι να κατανοήσουμε ότι η Βρετανική οικονομία και η Ευρωπαϊκή βασίζονται στις ειδικέ γνώσεις και την εμπειρία εργαζομένων που κυκλοφορούν από την Ευρώπη. Εάν από αύριο το Ενωμένο Βασίλειο δεν έχει πια πρόσβαση στο ταλέντο και τις δεξιότητες των ε, μηχανικών, ε, των ε, εργαζομένων με τις δεξιότητες που ψάχνει το Ενωμένο Βασίλειο και που τους έχει στην εγχώρια αγορά του, εάν δεν μπορεί να αντλήσει από αυτά τα ταλέντα στην Ευρώπη, θα πληγεί η ίδια ε, η βιομηχανία, όλος ο κλάδος ε, παραγωγής ε, στον Ηνωμένο και τούμπαλιν. Εάν δεν έχουμε εμείς πρόσβαση στα ταλέντα και τους εργαζομένους που έχουν εκπαιδευτεί στον Ηνωμένο Βασίλειο, εμείς χάνουμε. Αυτά λοιπόν συζητάμε σήμερα και κινδυνεύουμε να κάνουμε λιγότερο ανταγωνιστικά σε διεθνέ επίπεδο και τα 28 κράτη-μέλη. Δεν είμαστε μόνοι μα εδώ. Έχουμε να κάνουμε με ε, όλο τον κόσμο. Την Κίνα που είναι πολύ επιθετική, τη Ρωσία, τη Βραζιλία, τι ΗΠΑ. Εάν κάνουμε τα πάντα πιο δύσκολα, αν σχεράνουμε τα πάντα όχι μόνο για τον ΕΒ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αρχίσουμε να επιβάλλουμε δασμού, τότε η ευρωπαϊκή παραγωγή πολύ απλά, πολύ θα ακριβίνει και θα είναι λιγότερο ανταγωνιστική σε διεθνέ επίπεδο. Επόμενη διαφάνεια. Για μα, λοιπόν, για τι συνδικαλιστικέ οργανώσει, δεν θα σα ευνηδιάσει, ακούστηκε στην τελευταία παρέμβαση. Για μα, το θέμα είναι η κοινωνική ατζέντα του όλου θέματο ε, τη όλη συζήτηση. Διότι οι μελλοντικέ σχέσει και το πώ θα διαμορφωθούν μπορεί να οδηγήσουν σε ανταγωνισμό στα κοινωνικά. Ε, μία ε, κούρσα προς τα κάτω, στα κοινωνικά, στην απασχόληση, στην προστασία των εργαζομένων και ούτω καθεξής. Για μας λοιπόν σημαντικό είναι να διατηρήσουμε στις μελλοντικέ σχέσεις με το μενό Βασίλειο υψηλά πρότυπα και προδιαγραφές στα κοινωνικά και, ένα, ε, και κανόνες παιχνιδιού. Είναι προφανές και δεν θα σας ξαφνιάσει, διότι εδώ δεν εκπροσωπώ μόνο τις 27 χώρες ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου. Εδώ θέλουμε το κοινωνικό κεκτημένο, η ευρωπαϊκή κοινωνική ατζέντα, να θεωρηθεί ως βάση για τις μελλοντικές σχέσεις και στις κοινωνικές υποθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα το εξηγήσω αργότερα. Κατά δεύτερον, το ανέφερα και προηγουμένως, οπότε πολύ γρήγορα. Η απομάκρυνση, η αποχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο θα οδηγήσει και σε, σε αύξηση των διοικητικών δασμών. Ε, εάν δεν διαθετηθεί το θέμα αυτό κάπως, όλοι θα πληγούμε. Ε, μόλις στην αρχή της εβδομάδας, τη Δευτέρα, εκδώσαμε μαζί με τις χημικές ε, επιχειρήσεις της Ευρώπης, που είναι πολύ σημαντικές και για την Ευρώπη και για το Ηνωμένο Βασίλειο, μια κοινή δήλωση, όπου λέμε ότι υπάρχει μια σειρά από δυσκολίες για τις εταιρείε χημικών, εξαιτία των διαπραγματεύσεων του Brexit. Και μία από αυτέ, πέραν των κοινωνικών προτεραιοτήτων, όπου συμφωνούν και οι εργοδότε παρεμπιπτόντω, είναι και το θέμα της απόλυτης ανάγκης να υπάρχει εύκολη διοικητική διαχείριση. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι από την ΠΕΜΒΕ το έκαναν πολύ πιο σαφές με το παράδειγμα που, έδωσαν για τα φορτηγά. Και τρίτον, μην ξεχνάμε την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την κοινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Η Ευρώπη έχει τη φιλοδοξία μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι πλέον κοινοτόμο περιοχή στον κόσμο. Το έχει πει επανειλημμένω ξανά και ξανά του τελευταίου μήνε και χρόνια. Αυτή είναι η φιλοδοξία της και την συμμερίζεται και το Ηνωμένο Βασίλειο, υποτίθεται. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι σε ακαδημαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων, σε επίπεδο συνεργασίας, σχέσεων συνεργασία, μεταξύ ερευνητών που προσπαθούν να είναι καινοτόμοι στην Ευρώπη. Υπάρχει στενός συσχετισμό με το τι μεταξύ του τι συμβαίνει στον Ηνωμένο και τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με τα προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα που πρέπει να οργανωθούν Πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν στο μέλλον οι σχέσεις μας και η χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προγράμματα αυτά και τα οποία τα θέλουμε και στο μέλλον και θέλουμε να είναι καινοτόμα. Επόμενη διαφάνεια. Η Τερέζα Μέη, ακούστηκε πολύ σήμερα το απογευματόνομα, έχει βάλει πέντε τεστ και είπε ότι η μελλοντική συμφωνία πρέπει να προστατεύει τις θέσεις εργασίας και να δίνει και ασφάλεια για την απασχόληση. Η ερώτησή μας είναι τι θα πει αυτό, πώς θα το κάνετε. Για μας είναι σαφές ότι η πρόσβαση χωρίς δασμούς και φραγμούς είναι απαραίτητη συνιστόσα για να υπάρχουν ανταγωνιστικές θέσει εργασία. Μεν, αλλά αυτή η φιλόδοξη δήλωση τη Πρωθυπουργού ε, δημιουργείται ε, εξή πρόβλημα. Ε, βάζει και ένα σωρό κόκκινε γραμμέ και απαγορευτικά όρια. Αυτέ οι απαγορευτικέ γραμμέ, η διαφάνεια του ΙΑΝ τη ΜπενΔΕ, το δείχνουν ξεκάθαρα. Όλε αυτέ οι απαγορευτικέ γραμμέ εν τέλει μα φέρνουν στο βασικό πρόβλημα τη διαπραγμάτευση μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Ε, εδώ έχω τον περιβόητη διαφάνεια του Μπαρνιέ, ε, το ε, stay away του Brexit. Εδώ είναι αδύνατο να έχουμε συμφωνία όπως αυτή που είχαμε με την Νορβηγία. Αυτές οι απεγορευτικές γραμμές το κάνουν αδύνατο να έχουμε συμφωνία όπως αυτή που είχαμε με το... Ε, αδύνατο να έχουμε συμφωνία όπως αυτή που είχαμε με την Ελβετία ή με την Τουρκία πρέπει να δούμε μια συμφωνία τύπου Κορέας ή τύπου Καναδά. Δεν αρκεί λοιπόν αυτό. Ω συνδικαλιστικέ οργανώσει, όλοι μαζί τι κάνουμε. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε. Ξέρετε, γενικώ όλοι, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε πραγματικά τι θα πούνε όλε αυτέ οι κόκκινε επαγγελματικέ γραμμέ για την πραγματικότητα των εταιριών, για την ε, καθημερινότητα των εργαζομένων. Επόμενη διαφάνεια. Και τελευταία. Για μας μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών παρόμοια με τη ΣΥΤΑ του Καναδά δεν πάει αρκετά μακριά απλώς. Πρέπει να κατανοήσετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που νομικός θα είναι τρίτη χώρα, δεν είναι απλώς μια οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Θα έχει ειδικό καθεστώς. Και ήδη το έθεσαν και προηγούμενοι μιλητέ για τις ε, διαπλεκόμενες και τετεπλεγμένες εμπορικές σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας. Δεν είναι λοιπόν το ίδιο αυτό που θα συμβεί με τον Brexit όπως αυτό που συμβαίνει με τη Συμφωνία του Καναδά. Εάν δούμε εκεί τα πρότυπα της συμφωνίας αυτής υπάρχει μια σειρά από εξαιρέσεις στις συμβάσεις του ΑΕΛΟ και προ, προφανώς αυτό δεν μας αρκεί για το Ηνωμένο Βασίλειο. Συμπέρασμα λοιπόν, τι θέλουμε, φιλόδοξη κοινωνική ατζέντα στις διαπραγματεύσεις. Τι θα πει αυτό, θα πει ότι πρέπει να αποφύγουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ, να αποφύγουμε τον κοινωνικό ανταγωνισμό και ότι χρειαζόμαστε μία ρήτρα μη επαναχώρηση στι συμφωνίε αυτέ, όπου το κοινωνικό κεκτημένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει δεκτό ω ε, η βάση ως η αφετηρία. Και αυτό θέλουμε να συνεχιστεί και όταν το Brexit γίνει πραγματικότητα και να συνεχίσει να ισχύει και η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι δεν θέλουμε να πληρώσουν την πανταχούσα ε, και τα δικαιώματα τους το ίδιο επειδή γίνεται ανταγωνισμό ω προ τι αμοιβέ του από τι δύο πλευρέ τη μάχη. Λοιπόν, τα δικαιώματα των εργαζομένων, ε, κάτι που το υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή ε, Νομοθεσία, θα πρέπει να προστατευθούν με όσα ορίζονται για τι εταιρείε και την προστασία των εργαζομένων, για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασία και ούτω καθεξής. Είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να υποβαθμίσει τα εργασιακά πρότυπα για να υπάρξει περισσότερη ε, ανταγωνιστικότητα. Το ίδιο και για τους φόρους και τις φορολογικές συμφωνίες στο μέλλον. Ε, εν είδη συμπεράσματος λοιπόν δεν θέλουμε να γίνει ε, ένα παιχνίδι στα χέρια του ανταγωνισμού κοινωνική ατζέντα και να υπάρχουν ίσχυοι κανόνες παιχνιδιού που να βασίζονται στο ε, ισχυρό ευρωπαϊκό μας κεκτημένο. Ευχαριστώ πολύ. So, now Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο τώρα έχουν οι για δύο λεπτά. Να είστε παρακαλώ προσεκτικοί και να σέβεστε το χρόνο. Χόντε λίβε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όταν τα ακούμε όλα αυτά, ε, πρέπει να πω το εξή. Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις ε, μεταξύ των όσων ακούσαμε. Πρώτον. Δεύτερον, έχω την αίσθηση πως υπάρχουν κάποιες ιδέες που δεν είναι ρεαλιστικές. Όλοι θέμε soft Brexit, αλλά ίσως η άλλη πλευρά να θέλει κάτι διαφορετικό. Και το σενάριο βεβαίως με τα σύνορα. Ναι, το καλύτερο θα ήταν να μην υπάρχουν σύνορα. Ναι, αυτό θα ήταν το ιδεώδες εάν παρέμενε το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν το θέλει. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τώρα, γιατί ευθύς εξ αρχής ε, δεν ε, μπορώ να καταλάβω όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις του Brexit. Συγκεκριμένα δηλαδή, πώς φαντάζεστε το σύνορο μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας που δεν θα είναι σύνορο, που δεν θα το βλέπουμε, αλλά παρόλα αυτά θα είναι εξωτερικό σύνορο της Ένωσης. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο. Συγκεκριμένα, πώς φαντάζεστε ένα κράτος που πριν από 20-25 χρόνια σχεδόν σε μια άλλη ζωή είχε πει ότι δεν θέλει να υπογράψει την κοινωνική χάρτα γιατί έχει την δική του πολιτική στο θέμα αυτό κάτι το είχαν δεχτεί τότε όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Πώς θα πούμε τώρα, αν δεν δεχτείτε ILO και το Χ και το Ψ, τότε δεν θέμα. Ε, δηλαδή, Από τη μία λέμε θέλουμε, από τη μία λέμε δεν θέλουμε. Αυτή είναι σαν την κόκκινη γραμμή της ε, Τερέζας Μέη. Ε, περιμένω να πει κάπου και μία πράσινη γραμμή για να ξέρουμε ε, τι μπορούμε να συζητήσουμε τελικά. Θα ήθελα κάποιε διευκρινήσει λοιπόν για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. David Μάρτιν. Μετά από αυτό, ε, συμφωνώ πλήρω με αυτό το οποίο είπε ο Λουκ για τα κοινωνικά και το ότι πρέπει να διατηρηθούν, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι για πολλού από αυτού που ψήφισαν Brexit, όλο το νόημα ακριβώ είναι να ξεφορτωθούν όλα αυτά τα πράγματα παραπονιούνται για τον χρόνο εργασίας οδηγία ε, και τι άλλε οδηγίε κτλ. Και αναρωτιέμαι πόσο σοβαρά νομίζετε ότι θα πάει να ανταγωνιστεί η Βρετανία ρίχνοντας ε, τις κοινωνικές προδιαγραφές. Και τι μπορεί να κάνει επίσης στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άλλη γρήγορη ερώτησή μου μιλήσατε για μια παγκόσμια Βρετανία μετά το Brexit. Αλλά δεν ακούμε από την Βρετανική κυβέρνηση πρώτον αν υπάρχει ένα εφικτό χρονοδιάγραμμα να γίνει κάτι τέτοιο και το άλλο είναι με ποιον θέλουμε να κάνουμε αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Αν δούμε τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε που αναφέρατε. Έχουμε τον κύριο Τραμπ με την America First. Ε, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Αν πάρουμε μια χώρα σαν την Ινδία που ανέφερε η Βρετανική κυβέρνηση, γιατί θα επιτύχει το Ηνωμένο Βασίλειο εκεί όπου δεν τα κατάφερε την τελευταία δεκαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά καθώς ε, τα προβλήματα ήταν ε, βρετανικά συμφέροντα. Οι δασμοί στο ουίσκι που αναφέρθηκε και άλλα ζητήματα ήταν τα εμπόδια με την Ινδία. Και τέλος, ποια είναι αυτά τα προϊόντα που θα πουλήσουμε περισσότερο με μια συμφωνία ελευθερεμπορίου. Ε, τι, τι θα ζητήσει το, το Ηνωμένο Βασίλειο. Ποια αγορά δηλαδή προσπαθούμε να ανοίξουμε που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή και σύντομος. Ε, ε, ακούσαμε τον κύριο της Μπεμπέ, συμφωνώ με την ανάλυση που κάνατε, αλλά σας άκουσε η κυβέρνηση. Δηλαδή ότι ακόμα και αν φτάσετε Συμφωνία Ελευθέρου μπορεί, είμαστε πολύ χειρότερα από ό,τι τώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να με ακούσουν οι πανελίστες μας, ε, θα ήθελα να σα πω ότι είμαι Βρετανός συντηρητικός, αλλά έρχομαι εν ειρήνη. Ε, αισθάνομαι μια μηχανία, καθώς είμαι ένας από αυτούς που εμέσως ε, είναι και υπεύθυνο για το χάλι αυτό. Πριν θέσω ένα ερώτημα, ε, τέθη ένα ερώτημα από τον Κριστόφ όταν είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ποτέ δεν είχε πραγματικά επενδύσει στις ε, πολιτικές εξελίξεις ε, και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και μας ενδιαφέρει μόνο η οικονομική πτυχή και τα ωφέλη. Είμαστε όμως μια χώρα που πάντα λέγαμε ότι ήμασταν στην πρώτη γραμμή της κοινή αγοράς. Λέγαμε ότι εμείς τη φτιάξαμε, την βοηθήσαμε να μεγαλώσει κτλ. Αλλά βεβαίω. μαζί με αυτό αναγνωρίζουμε το ότι οι επιχειρήσεις έκαναν, έλαβαν κάποιες αποφάσεις με βάση την εξέλιξη της κοινή αγοράς. Γι' αυτό ακριβώς σήμερα βρισκόμαστε στην ε, κατάσταση ε, όπου κάποιοι μου λένε για γερμανικά αυτοκίνητα «Ε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι τουλάχιστον ευρωπαϊκά ή και παγκόσμια προϊόντα. Και ως χώρα, όταν είσαι σε αυτήν την θέση, έχεις μια ευθύνη να αναγνωρίσεις πως αυτό το οποίο συνδημιούργησες σήμερα απαιτεί κάποιες λύσεις. Τώρα, συνάδελφοι, ε, κάποιοι ανέφεραν ε, κάποιες από τις ε, συγκρούσεις και τις αντιφάσεις ε, στα επιχειρήματα των Brexiteer, αλλά για το σκοτσέζικο ουίσκι, David, εγώ όσο περισσότερο πίνω, τόσο ε, περισσότερο αντιλαμβάνομαι τα επιχειρήματά τους. Αλλά, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, ως α, ε, πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τον Νότιο Κάφκασο, Πήγα στον έλεγχο που υπάρχουν οι πιο εξελιγμένοι συνοριακοί έλεγχοι στον κόσμο μεταξύ Γεωργίας και Αρμενίας. Ε, τα χρηματοδοτεί μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί πέρα μπορεί ένα φορτηγό να περάσει σε δύο λεπτά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς έχουμε ένα χρόνο διάσχεση των συνόρων μηδέν. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι κάτι διαφορετικό ή όχι εντελώς. Η κυβέρνηση είπε ότι θα βγούμε και από την ψηφιακή ενιαία αγορά. Τι σημαίνει αυτό ειδικά σε σχέση με την έρευνα και την ανάπτυξη, γιατί το θέμα δεν αφορά μόνο τα πνευματικά δικαιώματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά τα ευαίσθητα βιομηχανικά δεδομένα σε μια τελείως διαφορετική νομική σφαίρα. Τι συνέπειες έχει αυτό, Χέλμουντ Σόλτς. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει στην ουσία του προβλήματος. Μιλάμε για την μελλοντική σχέση. Και υπάρχουν και τα ερωτήματα που έθεσε ο συνάδελφος ε, και ο σρόβολ πώς οι κόκκινες ή οι πράσινες γραμμές ε, θα γίνουν σεβαστές. Και ε, θα είναι σαφής. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο συνολικά πάντα λέγαμε ότι τρία σημεία θα πρέπει να μείνουν στη διαπραγματεύση, τα δικαιώματα των πολιτών. Νομίζω υπάρχει εδώ πέρα μια κοινωνική πτυχή, το θέμα της Βορείου Ιρλανδίας, ένα ε, συνοριακό θέμα που αφορά και το εμπόριο και τη μελλοντική εμπορική σχέση και το τρίτο ζήτημα των οικονομικών, της χρηματοδότησης. Και θέλω να είμαι σαφής. Μία μελλοντική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και κάποιες αλλαγές ε, των ε, πρακτικών. Όπως είπαμε και στην TTIP, δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε υποχωρήσεις στα ζητήματα τα αριθμιστικά. Και Βεβαίω αυτό ισχύει και για τα κοινοβούλια στα κράτη-μέλη. Ποια είναι τα διάφορα μοντέλα επίλυσης διαφορών που θα έχουμε. Οπότε όλες αυτές οι πτυχές ε, που συζητάμε ε, για μια συμφορία ελευθερμπορίου πρέπει να μας απασχολήσουν για το μέλλον και νομίζω είναι σαφές ποιο πρέπει να είναι το μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην χαμηλώσουμε τις προδιαγραφές που έχουμε επιτύχει στην ενιαία αγορά και στη σχέση με τρίτες χώρες. Αυτή είναι μια πρόκληση. Ακριβώ το θέμα είναι πώ βλέπετε αυτέ τι προσδοκίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριο Φιέρνερ. Νομίζω ότι αυτέ είναι κανονικά οι πιο εύκολε διαπραγματεύσει στον κόσμο. Ξεκινάμε από του δασμού συνήθω. Έχετε δασμού, όχι. Δεν έχετε δασμού, όχι. Ε, θα πάμε στου μη δασμολογικού φραγμού. Τι κανόνε έχετε, του ίδιου με εσά. Κανονικά θα έπρεπε να είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Και ε, εδώ ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε φραγμούς και να δημιουργήσουμε νέα εμπόδια στο εμπόριο και δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Οι διαπραγματεύσεις ε, συνήθως ε, έχουν τους πάντες κερδισμένους, αλλά εδώ οι πάντες θα βγουν χαμένοι σε σχέση με το που, από πού ξεκινάμε και αυτό δυσχεραίνει τα πράγματα. Βέβαια θα πρέπει να τίνουμε δίκον ους και να ακούσουμε τι έχει να μας πει το Λονδίνο και δεν θέλουν ε, ε, ενιαία αγορά, θέλουν αμοιβαία αναγνώριση. Η αμοιβαία αναγνώριση, αν καταλαβαίνω καλά, μπορεί να γίνει είτε μέσω ρυθμιστική ευθυγράμμιση ή μέσω ρυθμιστική συνεργασία. Υπάρχει κάποιο παράδειγμα ρυθμιστική συνεργασία τόσο προηγμένη με την εξαίρεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσε να εγγυάται και αμοιβαία αναγνώριση και να μην υπάρχουν αποκλήσει συνεχώ. Είπαμε όμω ότι ακόμα και αν πάμε στην ευθυγράμμιση, αν κατάλαβα καλά το μήνυμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του κυρίου Μπαρνιέ, δεν μπορεί να είναι Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κάρτα, πρέπει να τα δεχτούμε όλα αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πιο αυστηροί με το Ηνωμένο Βασίλειο από ό,τι κάναμε με την Ουκρανία, τη Μολδαβία, το Ισραήλ και εκεί έχουν πρόσβαση μόνο όταν ευθυγραμμίζονται. Και ρωτώ, είναι σωστό αυτό ή όχι. Και το αυτό ισχύει και για το φίλο μας από τα συνδικάτα. Ε, δυσκολεύομαι να λέω ότι πρέπει να λέμε το ένα στην Ουκρανία και το άλλο στην Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί εκεί δεν έχουμε καμία ευθυγράμμιση στον κοινωνικό τομέα. Ε, έχουμε δεχτεί τις δικές τους συμβάσει. ελπίζουμε ότι θα ευθυγραμμιστούν βεβαίω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υποχρεούνται να το κάνουν. Και ταυτόχρονα ο φορολογικό ανταγωνισμό υπάρχει και εντό τη Ευρωπαϊκής Είτε μα αρέσει είτε όχι, είναι πολύ δύσκολο να πούμε κάτι και να το επιβάλλουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε στα ίδια μας τα μέλη. Υπάρχει κάποια συμφωνία ελευθέρου συναλλαγή, υπάρχει χώρα που δεν έχει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Ε, οι περισσότερες έχουν και τέλος, εγώ δεν είμαι του εμπορικού, αλλά ε, έχετε έλλειμμα ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά με τις Ηνωμένε Πολιτείες υπάρχει πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Ε, και θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται. Ο Τραμπ θα ήθελε να μην υπάρχει καμία συμφωνία, αλλά με το Ηνωμένο Βασίλειο τι γίνεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα επανέλθω στην ερώτησή μου ε, για τον ε, Τζέρεμι Κόρμπιν και την Τελωνιακή Ένωση και το θέμα βεβαίως της Ιρλανδίας και των συνόρων και αν θα μπορέσουν να έχουν μια δική τους ε, πολιτική. Ο Κόρμπιν ε, λέει πως έχει κάποιες καλές ιδέες που έχει συζητήσει με βρετανικές επιχειρήσεις, ε, με κάποιες ιδέες. Ακούσαμε την κυρία Βάλτσμα και τον κύριο Ρόμπερτσον της BMW και τον κύριο Τρίγκλ. Τι άποψη έχετε γι' αυτό λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ και με πολύ μεγάλη χαρά δίνω το λόγο στην κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ παίρνω το λόγο με πολύ μεγάλη χαρά. Φοράω πράσινα, είμαι μέλος από τη Δημοκρατία της Ολλανδίας και γιορτάζουμε την ημέρα του Αγίου Πατρικίου λίγο αργότερα, ευπρόσδεκτοι όλοι. Ειλικρινά άκουσα μόνο το δεύτερο τμήμα αυτών των πολύ σημαντικών παρεμβάσεων, γιατί είχαμε μια άλλη συνεδρίαση που αφορούσε το Brexit στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Αν σας πω λοιπόν ότι πάσχω από Brexitίτιδα, νομίζω ότι θα καταλάβετε τι εννοώ και για να μιλήσω και λίγο πιο σοβαρά, εγώ εκπροσωπώ την περιφέρεια που έχει σύνορα με τη Βόρεια Ιρλανδία. Εμείς λοιπόν που νιώθουμε στο πετσί μας το πολιτικό πρόβλημα έχουμε και περισσότερο ε, ένταση όταν βλέπουμε προτάσεις, διαφάνειες και προτείνονται λύσεις. Για μένα δεν μπορεί να υπάρχουν σύνορα στη, μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας και σέβομαι τη σταγματικά η θέση της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσετε να με βοηθήσετε να καταλάβω πώς θα το πετύχουμε αυτό, δεδομένου ότι υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές του Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί αυτό με δυσκολεύει εμένα. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι εγώ ποτέ δεν θα ξανακοιτάξω ελικόπτερο χωρίς να σκεφτώ ε, που, από πού ε, προκύπτει το κυβότιο ταχυτήτων που έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ε, και τον κόσμο που ζούμε. Δεν έχω BMW, πολύ θα ήθελα να έχω, αλλά αυτά που μας παρουσιάσατε ήταν απίστευτα. Και πραγματικά πρέπει να πω, χωρίς να είμαι δύσκολη, γιατί δεν τα είχαμε ακούσει αυτά με μεγαλύτερη σαφήνεια πριν την ψηφοφορία ψηφοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο στο δημοψήφισμα. Όταν ε, σκέφτομαι την ενέργεια, το πολιτικό κεφάλαιο που επενδύουμε προσπαθώντας να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για να ελαχιστοποιήσουμε τις ζημίες για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματικά κουνά το κεφάλι μου και σκέφτομαι ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει πολύ καλύτερα για το λαό μας, εάν οι πολιτικές δεν ήταν τόσο κακοί. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Και ο κύριος Dartmouth. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ την προλαλήσασα για την εύγλωτη παρέμβασή της. Συνήθως δεν έχουμε τέτοια εύγλωτη, ε, τέτοιες εύγλωτες παρεμβάσεις ε, στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και τουλάχιστον όχι εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Όσον αφορά τις θέσεις ε, της ε, ε, Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και την Βόρεια Ιρλανδία υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο 43 σελίδων που το έχει δημοσιεύσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από 1,5 χρόνο περίπου το οποίο αναφέρει πώς μπορούμε να αποφύγουμε σκληρά σύνορα. Και θα ήθελα να σας το συστήσω και εσάς τον, και τον άλλον. Η κυρία Μαγκίνες, ε, ήμουν παρούσα όταν το παρουσιάσατε, δεν λύνει το πρόβλημα με όλο το σεβασμό. Ευχαριστώ, το διάβασα το έγγραφό Εγώ απλώς σας το σύστησα. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας το εξής, μια παρατήρηση. Ο κύριος Λόου ήταν πάρα πολύ καλός στην παρέμβασή του και να πω ότι στο βιβλίο μου, το οποίο το διάβασαν ελάχιστοι, προτείνω 11 διαφορετικές ρυθμίσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με εμπορικούς εταίρους της. Πλήρη συμμετοχή μέχρι και απλώς τελωνιακή ένωση, ελευθερία συναλλο... Ε, συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών κλπ. Και εδώ ακούσαμε και μία κόμμα. μια ε, κρυπτογραφημένη συμφωνία εμπορίου που από ό,τι φαίνεται έχει η Κίνα. Στην επόμενη έκδοση του βιβλίου θα προσθέσω και αυτή τη νέα κατηγορία. Να κάνω λοιπόν την παρατήρηση που είναι ε, και μάλλον παράδοξο. Όλοι αυτοί που είναι υπέρ του Brexit, όπως ο υποφαινόμενος ε, και τα υπόλοιπα 17 και εκατομμύρια ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλεια, ζήτησαν φιλία και ελεύθερο εμπόριο. Αν αυτοί του Remain που παρουσιάζουν όλα αυτά τα εμπόδια και ορισμένε φορέ είναι και στι παρυφές των απειλών αυτό το πράγμα. Ε, μήπως θα μπορούσαμε απλώ να προσπαθήσουμε να έχουμε φιλία και ελεύθερο εμπόριο και να ξεχάσουμε, να ξεπεράσουμε τα εμπόρια. Όλοι είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά αναζητούμε την καλύτερη λύση. Αλλά βεβαίω υπάρχουν και κάποια ερωτήματα εδώ στην αίθουσα. Η Γκοτλίβε το ανέφερε, το ανέφεραν ε, και η κυρία Μαγκίνες προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί. Να δώσω το λόγο λοιπόν στου εμπειρογνώμονε για δύο λεπτά ο καθένα. Και ξεκινάμε με τον Ιαν, γιατί πρέπει να φύγει λίγο νωρίτερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να προσπαθήσω να απαντήσω στην κυρία από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ίσως πρώτα. Ήταν πολύ σαφές το δημοψηφισμά μας και στην ΜΒΕ ήταν πολύ σαφέ το τι θα συμβεί, όμω εγώ δεν πιστεύω στην πολιτική ακριβώ, πιστεύω στη δημοκρατία. Τώρα πρέπει να βρούμε λύσει για κάτι το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο ψήφου σε δημοψήφισμα. Το σχόλιο λοιπόν που έκανα είναι ότι για την κατασκευή κάποιων προϊόντων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτή τη στιγμή ε, αυτή είναι η πραγματικότητα για την αυτοκινητομηχανία και το δικό μας, για την αεροναυπηγική κάτι άλλο, για τα γεωργικά επίσης. Ως κόσμος λοιπόν που δουλεύει σε επιχειρήσεις πρέπει να βρούμε απαντήσεις και εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς ότι θα καταλάβουν και τις δύο πλευρές του ίδιου επιχειρήματος ώστε να εμποδίσουν τη ζημιά που μπορεί να γίνει ε, και από τις δύο ακριβώς πλευρές. Η άλλη ερώτηση που θέλω να σχολιάσω είναι το αν ακούει η κυβέρνηση. έχει πολλές ευκαιρίες ο χώρος των επιχειρήσεων να συζητήσει με εκπροσώπους της κυβέρνησης και με την ίδια την Πρωθυπουργό κάποιες φορές, αλλά εν τέλει γίνεται λίγο παρασκηνιακή η συζήτηση αυτή, λίγο και κλεισμένων των θυρών. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξέρουμε τι γίνεται στις πολιτικές συζητήσεις που ακολουθούν τις δικές μας συνομιλίες. Πάντως, ε, δεκτικότητα και καλή υποδοχή έχουμε. Το τι συμβαίνει μετά ε, είναι κάτι που θα πρέπει να το ρωτήσετε στους ε, μπλεκόμενους πολιτικούς. Και μετά για τα επιμέρους ζητήματα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει να κολλάμε σε ορισμούς που καταλαβαίνουμε ότι συζητιούνται αλλά είναι οπισθοδρομικοί. Πρέπει να δούμε και τις δύο πλευρές της εξίσωσης είτε από την πλευρά των επιχειρήσεων είτε της παραγωγής και να βρούμε ε, μια πρόταση που να λειτουργεί. Δεν ενδιαφέρει αν θα είναι τελωνιακή ένωση, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας επιχειρηματίας στην Ευρώπη που θα έλεγε όχι σε αυτό. Αυτό που χρειάζεται να βρούμε είναι πολιτική επένδυση και απάντηση για να δοθεί τέλος και καλή έκβαση σε αυτή την ατζέντα. Ευχαριστούμε Στέφανο. Ευχαριστώ. Απλώς ένα παράδειγμα ήταν είπα, για τα τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε διπλωματεύσει. Παρόμοια προβλήματα θα προκύψουν ακόμη και αν το Ηνωμένο Βασίλειο ε, τον ίδιο οικονομικό χώρο με την Κορέα, ας πούμε. Ανέφερα τη ΣΥΠΑ γιατί εκεί το επίπεδο φιλοδοξιών είναι μεγαλύτερο. Όμως, από αυτή την πλευρά, τέλο πάντων από αυτά που άκουσα σήμερα, άκουσα ότι υπάρχει περισσότερο η τάση να πούμε στον Ηνωμένο Βασίλειο μείνετε μαζί μα και κοιτάξτε να βρούμε με τι τρόπο θα γίνει αυτό. Το πρόβλημα όμω είναι ότι θέλει να κάνει και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι επιλογέ εδώ είναι δύο. Είτε επαναλαμβάνει ε, όλε τι συμφωνίε Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ελεύθερων συνελλαγών με τρίτε χώρε, είτε όχι. Ακούσαμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ε, μου είπανε μάλλον και ακούγονται ειδήσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο σκέφτεται να πάει προ τα εκεί. Εάν όμω αναπτύξει κανόνε που είναι ανεξάρτητα από τα όσα ίσχυαν ε, όταν ήταν μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να σκεφτούμε τι τεχνική λύση θα δοθεί και όσο το δυνατόν συντομότερο. Διότι οι εταιρείε μα λένε τώρα ότι αυτό που χρειάζονται περισσότερο είναι κάτι το ε, σίγουρο, το βέβαιο. Και αυτό μπορεί να γίνει πιο γρήγορα από ό,τι και δημοτεύσει. Αν δεν βρείτε λοιπόν λύση για τι επιχειρήσει, δεν μπορούν μόνοι του. Και όταν τη βρούμε, θα επιβιώσουν. Όταν τη βρούνε, μάλλον, θα αναγκαστούμε να επιβιώσουμε. Δεν είναι πολιτικοί οι εταιρείε. Κέρδο θέλουν. Ό,τι και αν γίνει. Η σύστασή μου, ο κ. Ρόμπισον, μόλι έφυγε. Τέλο πάντων, ε, να. Ε, είμαστε τα δυνατόν πιο συγκεκριμένοι να έχουμε μια λύση πολύ χειροπιαστή. Νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε. Ναι. Θα συνεχίσω αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής και απαντούσε σε ερώτηση. Πρώτα απ' όλα ήταν ιστορικό επίτευγμα του Ηνωμένου Βασιλείου να διαμορφώσει την ενιαία αγορά αναντήρητα και το ε- υπερευχαριστούμε μέχρι και σήμερα. Αλλά γι' αυτό ακριβώς σας χρειαζόμαστε και στο μέλλον, διότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της και χρειαζόμαστε όθηση, χρειαζόμαστε ε, κινητήριες δυνάμεις, το ελεύθερο εμπόριο, ελεύθερες συναλλαγές. Ξέρουμε ότι απειλείται η Ευρώπη. Ξέρουμε ότι το ελεύθερο εμπόριο ότι μάλλον ακόμα και τώρα χρειαζόμαστε συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου. Περνάει ο χρόνος, η Ασία μεγαλώνει. Εάν ε, δεν προχωρήσουμε, εμείς θα φταίμε. Και για του μη εμπορικού φραγμούς. Αυτό θέλαμε και πάντοτε ήταν δεσμευμένο εδώ το Ηνωμένο Βασίλειο και αγωνιζόταν. Δεν τους ενδιέφερε η πολιτική εμβάθυνση των σχέσεων, η ασφάλεια ίσως, ε, τα κοινωνικά εκεί εμπόδιζαν και δεν ε, ήταν, αποτελούσαν μέρος της λύσης. Κατά τα άλλα ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο ένας επικοδομητικότατος εταίρος για την Ένωση. Άρα η δική μου αντίληψη της ερώτησης είναι γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό και, το, και στο μέλλον. Ακούστηκε ε, και για πράσινε γραμμέ, όχι μόνο κόκκινε. Εσεί έχετε μπλοκάρισμα στη σκέψη σα. Εσεί μπλοκάρετε τη δημιουργικότητά σα. Γιατί δεν έχετε πράσινε γραμμέ, τι θέλετε. Θέλετε πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Οκ, αλλά τι σα εμποδίζει. Υπάρχουν κάποιοι κανόνε που πρέπει να γίνουν σεβαστοί, αλλά πάντοτε υπάρχουν και λύσει. Είμαι επιχειρηματία. Αν έχω πρόβλημα, βρίσκω λύση. Μαζί με την ομάδα μου, μαζί με του συνεργάτε μου. Σε αυτό το πρόβλημα τώρα ε, δεν έχουμε βρει ακόμα λύση. Πρέπει να γίνει και σε αυτή την περίπτωση κάτι τέτοιο, πρακτικό. Αυτό θέλω να πω λοιπόν. Να είμαστε λίγο πιο πραγματιστές, λίγο πιο ρεαλιστές και ε, πιο δημιουργικοί. Όχι εγώ τα στυλώνω εδώ και εσύ τα στυλώνεις απέναντι και δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Να βρούμε μία λύση κοινή. Αυτό ενδιαφέρει την οικονομία και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα στον βοηθό μου ήταν δεν θέλω προβλήματα, θέλω λύσεις. Λοιπόν, Λουκ, θα είμαι σύντομος, θα ήθελα να απαντήσω όμως σε δύο-τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ναι, αντιλαμβάνομαι τους λόγους ε, του Brexit και ε, πρόσεξα τι είχε γίνει τις ε, τελευταίες εβδομάδες ε, στην δημόσια συζήτηση και στον τύπο του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά αυτό το οποίο υπόθηκε αμέσως μετά ήταν ότι το τέλος του 2009 θα έχουμε τη χώρα μας πίσω. Ε, ήδη αυτό έχει πάει για το τέλος του 2020 και η αγορά μέχρι το τέλος του 2020 και ελευθερή μετακίνηση τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2020. Οπότε τα πράγματα αλλάζουν και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι πως όταν διαπραγματευόμαστε πρέπει να έχουμε κατά νου το κοινωνικό κομμάτι ως Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να πιέσουμε το θέμα της κοινωνικής ατζέντα. Να μην είναι δηλαδή ζήτημα ανταγωνισμού, γιατί αυτό θα βλάψει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί γνωρίζουμε ακριβώς το θέμα αυτό γιατί θα πρέπει και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνδεθούν με τα θέματα αυτά. Το ένα είναι αυτό. Και άρα πρέπει να ενημερώσουμε γι' αυτό το θέμα, να εξηγήσουμε γιατί είναι το σημαντικό. Δεύτερον, και εδώ πέρα ίσως διαφέρει λίγο ίσως η άποψη μου από τους προηγούμενους ομιλητές ότι ναι θέλουμε πρόσβαση στην ε, εσωτερική αγορά ή κάτι παρόμοιο, γιατί έχει μεγάλη σημασία για την βιομηχανία. Αλλά να είμαστε σαφείς, δεν μπορούμε να το αποσυνδέσουμε από τις άλλες πραγματικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις τέσσερις ελευθερίες, ε, την ελεύθερη μετακίνηση, η αποδοχή του και εκτιμένου, γιατί δεν διαπραγματευόμαστε μόνο τη μελλοντική σχέση με τον Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και το μέλλον τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του 27. Φανταστείτε δηλαδή ε, να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα λέμε εντάξει, τελωνιακή ένωση και πρόσβαση και θα είναι πολύ εύκολο να έχουμε εμπόριο και ανταλλαγέ, αλλά από την άλλη δεν χρειάζεται να σέβεστε πλέον τα άλλα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ε, ελευθερία μετακίνηση, το κοινωνικό και εκτιμένο. Ε, όχι, τότε ανοίγει πόρτα και για άλλες χώρες ε, η πόρτα της εξόδου, γιατί και άλλες χώρες θα ζητήσουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Οπότε το θέμα δεν αφορά μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και το μέλλον της ίδιας της Ένωσης. Τρίτο και τελευταίο, η διακήρυξη του Κόρμπιν, α, εντάξει, τελωνιακή ένωση. Ναι, εντάξει, αλλά τι εννοούμε με αυτό. Υπ' αυτήν ε, την έννοια νομίζω πρέπει ακριβώς ε, να φύγουν αυτές οι κόκκινες γραμμές, να αρχίσει η διαπραγμάτευση και ε, η Ουκρανία δεν είναι το ίδιο με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε ακούσει ήδη για τις στενές ε, βιομηχανικές σχέσεις. Πρέπει να έχουμε κάτι καινοτόμο και φιλόδοξο, αλλά να μην αφορά μόνο το εμπόριο, αλλά και την οικονομική πτυχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους ε, πανελίστες. Νομίζω πως τώρα η εικόνα είναι σαφέστερη. Ίσως όχι η λύση, αλλά εντάξει. Το παλεύουμε. Και δίνω τον λόγο στην εισηγήτριά μας. Σας ευχαριστώ. Ε, δεδομένου του χρόνου, ε, μία σκέψη μόνο θα ήθελα να αναφέρω. Γνωρίζουμε τώρα λοιπόν πώς μπορεί να χειραγωγήσει κανείς τις εκλογές, τα δημοψηφίσματα και προκύπτουν νέα πράγματα κάθε μέρα. Υπάρχει μια δυνατότητα πιθανώς να μεταβληθεί η γνώμη στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Ποιος ξέρει. Να δούμε. ελπίσουμε ότι το παρελθόν δεν θα κρίνει το μέλλον. Ας το τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ. Τελειώνουμε με αυτό το σημείο. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, η συμφωνία με το Μεξικό ε, και το σχετικό πρωτόκολλο υπό το φως της ένταξης της ε, Κροατίας. Δίνω τον λόγο αμέσως στον προϊστάμενο, τον κύριο Γιώργινσεν. Όποιος θέλει να φύγει παρακαλώ ήσυχα. Ματίας, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι σύντομος. Πρόκειται για Σας ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε. Είναι μια πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για να ληφθεί μια απόφαση στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχουμε με το Μεξικό για να προσθεθεί εκεί και η ένταξη της ε, Κροατίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται για το τρίτο πρωτόκολλο υπό αυτήν την συμφωνία για τον σκοπό Το πρώτο πρωτόκολλο βεβαίως ε, ήταν για τους 10, το άλλο ήταν για τους 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα έχουμε την ένταξη της Κροατίας. Είναι μια απόφαση λοιπόν. Έχουμε ακριβώ τα κείμενα. Περιλαμβάνουν ε, μια μικρή προσαρμογή στην ποσόστοση της μπανάνας που έχουμε με το Μεξικό, πολύ μικρή, 10 Και αυτό γιατί η απώλεια του Μεξικού όσον αφορά τις εξαγωγές μπανάνες στην Κροατία είναι πολύ περιορισμένες. Αυτό είναι ένα από τα πρωτόκολλα. Όπως ξέρετε έχουμε κινήσει και άλλες αναλογικές διαδικασίες με Περού και Κολομβία και Χιλή και αυτό είναι άλλο ένα πρωτόκολλο. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Η Κάρολιν θα πάρει τον λόγο εξ ονόματος της Ημακουλάδα, ε, της ε, εισηγητριάς μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το 1990 και το 1997 ήταν η πρώτη χώρα που υπέγραψε εταιρική σχέση ε, και σχέση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μεξικό. Η συμφωνία αυτή τέθηκε σε εφαρμογή το 2000 και λαμβάνει υπόψη του στις εμπορικές σχέσεις και τη συνεργασία. Η συνολική συμφωνία περιλαμβάνει και διατάξεις εμπορίου. Στο άρθρο 6.2 της προσχώρησης της Κροατίας, ε, η Κροατία ανέλαβε να προσχωρήσει στη τις κείμενες συμφωνίες ε, που έχουν συναυθεί από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Η Κροατία προσχωρά, ε, προσχωρεί μέσω των ε, συμφωνιών που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Το Σεπτέμβριο του 2012 το Συμβούλιο έδωσε έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες ε, για να ε, συναυθούν τα σχετικά πρωτόκολλα. Ε, η συμφωνία με το Μεξικό ολοκληρώθηκε επιτυχώς και αυτό το πρωτόκολλο είναι το επιπλέον πρωτόκολλο στη συνολική συμφωνία με το Μεξικό για να λάβουμε υπόψη και την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει την συνάψη αυτού του πρωτοκόλλου το οποίο ε, συμπεριλαμβάνει και την Κροατία ως ε, μέλος ε, στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού. Και μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα προς την κύρωση αυτού του επιπλέον πρωτοκόλου, Υπάρχουν και κάποιες συμφωνίες του Κοινού Συμβουλίου που καθορίζεται στην Συνολική Συμφωνία και πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές για να γίνουν προσαρμογές στις προβλέψεις για το εμπόριο. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα για το περιεχόμενο αυτών των αποφάσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φίσας απουσιάζει. Η Έμμα Μακλάρκινγκ. Να πω απλώς ότι το ECR υποστηρίζει αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικά. Ελευθέρους δεν έχουμε. Γκουε. Σχόλια όχι. Οι πράσινοι απουσιάζουν. Το EFTD. Ο κύριος Ρούμπιχ. Ήθελα να συγχαρώ την συνάδελφο. Νομίζω πως είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Όλοι γνωρίζουμε πως η Κροατία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά και η σχέση με το Μεξικό θα αποκτήσει μια νέα διάσταση και νομίζω ότι θα αυξηθεί η αγοραστική δύναμη και των δύο πλευρών και μπορούμε να το στηρίξουμε ως ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ωραία. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Απίστευτο. Μάλιστα. Ματίας. Έχετε την ευκαιρία να σχολιάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Τα έγγραφα βασίζονται σε αντίστοιχες ε, φωνές προσχώρησης όπως και στο παρελθόν. Είναι τα συνήθη. αποτελούνται από αποφάσεις που θα προσαρμόσουν ε, τις κοινέ ε, αποφάσεις Συμβουλίου του Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού 2000 και 2 κάθετος 2001 που είναι διατάξεις για το εμπόριο και τις υπηρεσίες ε, του πυλώνα εμπορίου της Συνολικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού. Όσον αφορά την ουσία, όπως είπα, θα γίνουν αλλαγές στους κανόνες προέλευσης, διότι θα υπάρχει ένα παράρτημα ε, πλέον και στα κροατικά. Θα υπάρχει προσαρμογή ε, στις δημόσιες προμήθειες για να λάβουμε υπόψη και ε, τους φορείς που θα συμπεριλάβει η Κροατία στη συμφωνία και φυσικά υπάρχει και μία πολύ μικρή, όπως σας είπα, και είναι η πραγματική ουσιαστική αλλαγή, μία αποζημίωση για απώλεια προτιμησιακής πρόσβασης ε, του Μεξικού ε, στην κροατική αγορά. Και αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένουμε και την επίσημη έγκριση του Συμβούλιο για να προχωρήσει το όλο θέμα. Σχέδιο έκθεσης εφόσον υπάρξει η έγκριση 16 και 17 Μαΐου για να ψηφίσουμε τον Ιούνιο ανάλογα με το τι θα κάνει και το Συμβούλιο. Μια και μάλλον μας ακούει εδώ το Συμβούλιο και κάποιος εκπροσωπό του, ε, ανασκουμποθείτε λίγο. Βλέπετε ότι στο Κοινοβούλιο όλοι είναι υπέρ του να δώσουν σύμφωνη γνώμη για τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε και το σημείο 11 και τώρα να περάσουμε καυτό το θέμα. Δασμοί χάλιβα και αλουμινίου από τη ΣΥΠΑ. Περιμένουμε τον κύριο Ντεμάρτη, Γενικό Διευθυντή για το Εμπόριο της Γενικής Διεύθυνσης Trade δηλαδή, και θα ξέρετε, θα θυμάστε ότι το θέμα αυτό το συζητήσαμε στην προηγούμενη Ολομέλεια με τον αρμόδιο επίτροπο. Πολλά έχουν ε, λεχθεί από τότε που έγινε αυτή η συζήτηση στην Ολομέλεια. Ήταν ε, ο Αμερικανός υπεύθυνο ε, εδώ στις Βρυξέλλες, ε, η κυρία Μάλστρομ πήγε στην Ουάσιγκτον και ο Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας πήγε μια βόλτα. συνάντησαν τον κύριο Ρος, κάποιους γερουσιαστές, μέλη του Κογκρέσου, είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί γρήγορα. Αλλιώς, εάν ε, ισχύσουν την Πέμπτη Παρασκευή οι δασμοί, αυτό μπορεί να ημειώσει την, ε, ευρωπαϊκή ευρωπαϊκές και θα πλήξει όχι απευθεία τι ε, εξαγωγέ μόνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ τη ΣΥΠΑ, καθώ δεν ξέρει κανεί ποιε τελωνιακέ γραμμέ είναι αυτέ που θα αφορούν οι δασμοί, αλλά θα επηρεαστεί και ο όγκος χάλιβα που φτάνει στην Αμερικανική αγορά και στην Ευρωπαϊκή. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας, κάποιους μηχανισμούς επίσης. Όλοι ζητούν από τις ΗΠΑ να μην υπονομεύει τις διευθυντήσεις του ΠΟΕ. Εγώ ο ίδιος απέστειλα επιστολή στην λεγόμενη Επιτροπή Μίνσκ και τις επαφές που έχουμε με τους ομολόγους μας στις ΗΠΑ τις εκμεταλλευτήκαμε για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάπως τα πράγματα, την θέση του Προέδρου της χώρας. Έχουν ακουστεί πολλές επικριτικές φωνές και στη ΗΠΑ, και γίνονται όλο ένα και πιο δυνατές παρόλο που ο πρόεδρος του Κογκρέσου, ο κύριος Γουάιν, διαφώνησε ανοιχτά με την επιβολή αυτών των δασμών και κάποιοι γερουσιαστές το ίδιο. Οι εταιρείε ακόμα δεν έχουν κανένα δείγμα από τον πρόεδρο της θα γνώμη. Η αναγγελία για τους δασμούς που θα βασιζόταν ε, στο νόμο, τον υπέροχο νόμο του 62 είναι κάτι που το έκανε ο πρόεδρος αποφασίζοντας να δράσει από μόνος του αν κάποια συμφέροντα της χώρας στο επίπεδο της ασφάλειας ε, βρίσκονται σε κίνδυνο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δύναται και επιτρέπεται ο πρόεδρος να, ε, λάβει, να αναλάβει δράση μόνος του. Δεν ξέρω κατά πόσο να αποτελεί θέμα δημόσια ασφάλεια, διότι μόνο το 3% τη παραγωγή χάλιβα στη ΣΥΠΑ ε, έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια. Η όλη η συζήτηση μεταξύ των νομικών και δικηγόρων στη ΣΥΠΑ έχει να κάνει με το κατά πόσον χρήση αυτού του νόμου που είναι από την εποχή του ψυχρού πολέμου είναι κάτι το λογικό και εφικτό. Και πολλές εταιρείε φαντάζομαι ότι και εντός είπα, θα έχουν πρόβλημα στο Κογκρέσο. Υπάρχει η άποψη ότι θα πρέπει να αλλάξει ο παλιός αυτός νόμος για να πάρει την εξουσία στα χέρια του ακριβώς ε, το Κογκρέσο με τους εκλεγμένους ερετούς αντιπροσώπους. Έκανα ό,τι μπορούσα να δώσω κάποιες πληροφορίες για την ε, σε εξέλιξη, διένεξη και ελπίζω ότι θα φτάσει ο Ζανλουκ. Soon until then I will give the floor to Jean-Luc immediately and we have... Όταν έρθει θα του δώσω αμέσως το λόγο. Έχουμε πυρογνώμονες και κάποιους από τους ενδιαφερομένους εκπροσώπους όσων πλήττονται από αυτή την προσέγγιση. από τη Eurofora, εκπρόσωπο της Χαλιβουργίας στην Ευρώπη και το Γενικό Γραμματέα της All καθώς και εκπρόσωπο των εργαζομένων στη Χαλιβουργία. Μετά το Ζανλούκ λοιπόν θα τους καλέσω να μας μιλήσουν. Save your voice. We might just... Κοίταξε, ίσως κάνουμε ένα διάλειμμα για να σταματήσετε να μιλάτε. Καλά, αυτό μπορώ και εγώ. Otherwise, I would say something about um, uh, or maybe being quiet. Ίσως να σοπάσετε, είναι ένα καλύτερη. Skills, I don't know. So, there's a wonderful proposal. Εξαιρετική πρόταση. Θα αρχίζαμε στις 5 και 20, αλλά ας κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Πολύ σύντομο το διάλειμμα. Λοιπόν, ήρθαν όλοι. Ζαν Λουκ, καλώς ήρθες. Κάνα μία εισαγωγή για τις εξελίξεις ε. και το πρόβλημα ήταν οι εξελίξεις, ε, η έρευνα και τα λοιπά. Το μόνο το οποίο δεν ξέρουμε είναι το αποτέλεσμα της επίσκεψης ε, της ε, Σεσίλια Μάλμστρομ στην Ουάσιγκτον. Οπότε αναμένουμε να ακούσουμε από εσάς το τι έγινε και τις δυνατότητες αντίδρασης. Λοιπόν, έχετε αμέσως τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα η επίσκεψη της ε, Σεσιλίας ε, συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν μπορώ λοιπόν ε, τώρα παρά να σας πω ότι συνεχίζονται οι επαφές. και βεβαίως ε, γίνονται κάποιες ε, δομητικές ε, συζητήσεις και συναντήθηκε η Σισίλια Μάνστρομ με τον κύριο Μπαρός χτες το απόγευμα και αποφάσισαν να ξεκινήσει μια διαδικασία ακριβώς για τις ανησυχίες που υπάρχουν στον τομέα του αλουμινίου και του χάλιβα. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια εξέλιξη για μια πιθανή εξαίρεση και ο πρέσβης, ο κ. Λάιτχάιζερ, αναφέρθηκε σε μια πιθανή εξαίρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Αυστραλία και την Αργεντινή και πιθανώς ε, και κάποιες άλλες χώρες ε, στην παρέμβασή του σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών της ε, Βραζιλίας. Οπότε τίποτα νεότερο σε αυτήν την φάση. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ επιφυλακτικοί. Οπότε θα ξεκινήσω με το πόσο έχει η κατάσταση αυτήν την στιγμή Αλλά η βεβαιότητα μπορεί να σημαίνει ότι το μεσημερί της Πέμπτης, ε, βράδυ δηλαδή, ε, η Παρασκευή πρωί, οι επιπλέον ε, αμερικανικοί δασμοί που βασίζονται στο 2.32 να εφαρμοστούν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια επιβεβαίωση ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αν και έχουν υπάρξει επικοδομητικές συζητήσεις. Όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή τα πράγματα στην Ουάσιγκτον, ε, η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 12.30, οπότε οι συζητήσεις συνεχίζονται. Οπότε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιτρέψατε μου να ξεκινήσω ε, ευχαριστώντας σας ε, για την στήριξή σας σε μια αναλογική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Αμερικανικά μέτρα. Δείχνουμε ένα ενωμένο μέτωπο. Σήμερα λοιπόν θα αναφερθώ σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα το τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής με την αβεβαιότητα στην των Δεύτερον το τι περιμένουμε να συμβεί και το τι ελπίζουμε. Ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε πρόσφατα την επιβολή δασμών 25% στο χάλιβα και 10% στο αλουμίνιο. Το έκανε ε, σύμφωνα με το άρθρο 232 του νόμου περί εμπορίου. Το συγκεκριμένο άρθρο ήταν έκπληξη. Αυτό είχε νομοθετηθεί στον ψυχρό πόλεμο για να χρησιμοποιηθεί κατά εχθρικών χωρών και βλέπουμε ότι σήμερα χρησιμοποιείται αλλιώ. Λείπομεθα για διάφορους λόγους ε, για το ότι είπα αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέτρα και το να το αιτιολογούν για με λόγους εθνικής ασφαλείας είναι ένας κίνδυνος. Υπονομεύει το πολυμερές εμπορικό σύστημα που είναι ο καλύτερος τρόπος να επιτύχουμε δίκαιο εμπόριο που θα βασίζεται σε κανόνες. Επιπλέον είναι ένα απογοητευτικό μήνυμα όσον αφορά την εμπιστοσύνη καθώς η Ευρώπη εδώ και καιρό είναι εταίρος στον τομέα της ασφαλείας και νομίζουμε ότι δεν απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΙΠΑ οι Είμαστε δε πεπισμένοι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξαιρεθεί από αυτά τα μέτρα. Η Επίτροπος Μάλστρομ κατέστησε αυτά τα πράγματα ξεκάθαρα στη συναντήση με τον πρέσβη και τον Υπουργό τον κύριο Ρος. Σε αυτήν την φάση δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν και πότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαιρεθεί, εάν εξαιρεθεί. Εάν δεν εξαιρεθούμε, θα υπάρξει μια στιβαρή και αναλογική απάντηση. Ε, προετοιμάζουμε αυτό το σενάριο. Ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα. Ακόμα και αν ε, δεν είναι σίγουρο, αλλά μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Είμαστε σε στενή επαφή με τους ε, ομολόγους μας ε, στις ΗΠΑ. Η Σεσίλια Μάστρο μεταφέρει το μήνυμα ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σαφήνεια και αν δεν εξαιρεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρξει μια άμεση απάντηση. Η απάντηση αυτή έχει ήδη εξηγηθεί από την Επίτροπο στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Θα έχει τρεις πτυχές. Προσφυγή στον ΠΟΕ, μια διασφάλιση για να προστατεύσουμε τις αγορές μας, και θα αντισταθμίσουμε τα ωφέλη των ΙΠΑ σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες γιατί θεωρούμε πως ε, τα μέτρα που λαμβάνουν οι ΙΠΑ δεν είναι θέματα εθνικής ασφαλείας, είναι κατ' ουσίαν μια καμουφλαρισμένη προσπάθεια προστατευτισμού. Σκοπεύουμε λοιπόν να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και το πολυμερές εμπορικό σύστημα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και όπως σας είπα, προσγειώθηκα πριν από λίγες ώρες από το Δελχείο που υπήρχε μια σημαντική υπουργική διάσκεψη που οργάνωσε ο ΠΟΕ και η Ινδία ε, εκπροσώπησα την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους προφανείς λόγους δεν μπορούσε η κυρία Μάλστρομ και οφείλω να σας πω πως οι περισσότεροι από τους 50 συμμετέχοντες εξήγησαν ε, την βαθύτατη ανησυχία τους για τα μέτρα του άρθρου 232 και την μονομέρεια και επίσης, ε, χωρίς να είναι το σημερινό μας θέμα, αλλά το αναφέρω γιατί πολιτικά έχει μεγάλη σημασία, ε, ότι και εκτός της εμπορικής πτυχής υπάρχει μια κρίση, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος ε, να παραλύσει ο μηχανισμός επίλυσης ε, διαφορών στον ΠΟΕ για πάνω από ένα χρόνο. Μέτρα αυτά λοιπόν τα επιλέξαμε προσεκτικά. Δεν θέλουμε να κλιμακώσουμε την κατάσταση. Θέλουμε να λειτουργήσουμε εντός του νομικού πλαισίου του ΠΟΕ να είμαστε αυστηροί αλλά αναλογικοί. Δεν πρέπει να αντιδράσουμε υπερβολικά, αλλά ούτε και να αντιδράσουμε λιγότερα από όσο θα πρέπει. Το πρώτο λοιπόν μέρος είναι η αντίδραση στο άρθρο 2.32 για να έχουμε κάποια δικαιοσύνη στο πολυμερές εμπορικό σύστημα. Αλλά θα χρειαστεί χρόνος ε, και είναι άμεσος ο κίνδυνος για τα οικονομικά μας συμφέροντα. Και βεβαίω λαμβάνουμε υπόψη το ότι χρειάζεται χρόνος στον ΠΟΕ και η πιθανή παράλυση που ανέφερα μπορεί να συμβεί, οπότε πρέπει να λάβουμε τώρα τα πιο αποτελεσματικά μέτρα. Γι' αυτό έχουμε κάποιες άμεσες ε, αντιδράσεις πέρα από τις μακροπρόθεσμες. Το δεύτερο τμήμα της αντιδρασής μας είναι να προστατεύσουμε τις αγορές μας από την ε, αλλαγή των εμπορικών ροών. Οι ΗΠΑ θέλουν να μειώσουν τις εισαγωγές χάλιβα κατά 30 εκατομμύρια τόνους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να θυσιάσουμε το ότι είμαστε ανοιχτοί στο εμπόριο, αλλά πρέπει να προστατευτούμε από αφύσικες στρεβλώσεις της αγοράς. Αυτό σημαίνει παρακολούθηση της αγοράς και το να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε γρήγορα όπου αυτό είναι δυνατόν. Δεν θέλουμε να κλείσουν περαιτέρω οι αγορές χάλιβα και αλουμινίου και ενθαρρύνουμε και τους εμπορικούς μας εταίρους να κάνουν το ίδιο. Εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, τότε υπάρχει η επιλογή ε, η τρίτη, δηλαδή να απαντήσουμε δίκαια και νομίμως ε, να υπάρξει μια αντιστάθμιση ε, στα πλαίσια της συμφωνίας του ΠΟΕ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Από την ε, Παρασκευή ήδη διαβουλευόμαστε για το ποια προϊόντα θα μπορούσαν να περιληφθούν σε έναν κατάλογο αντισταθμιστικών ενεργειών. Ε, είναι διαθέσιμος ο κατάλογος ε, και στην ιστοσελίδα μας και μετά την διαβούλευση θα οριστικοποιεί. Στην αρχή θα μιλήσουμε για αντιστάθμιση δύο 1,8 ε, δισεκατομμυρίων ευρώ, που είναι λιγότερο από την απώλεια των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, γιατί σεβόμαστε πλήρω τα κριτήρια τη συμφωνία διασφάλιση που έχουμε υπογράψει ε, στον ΟΠΟ, ειδικά το άρθρο 8. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αποφύγει μια σοβαρή εμπορική διαμάχη που δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όλοι γνωρίζουμε πως η ρίζα του προβλήματος ε, που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα αμερικάνικα μέτρα δεν είναι το εμπόριο, είναι οι υπερβολικές ε, δυνατότητες παραγωγής που υπάρχουν ε, στον Χάλιβα. Το έχουμε συζητήσει με τις ΗΠΑ στο παρελθόν. Κάποιες χώρες χρησιμοποιούν τεράστιες επιδοτήσεις, παράγουν σε συνθήκες μη αγοράς και συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για αυτό το ζήτημα και σκοπεύουμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον. Είναι δύσκολη η κατάσταση χρειάζεται σαφήνεια, αλλά δεν σημαίνει αυτό εμπορικό πόλεμο. Η ΕΠΑ είναι εταίρος πολύτιμος σε πολλούς τομείς, στην ασφάλεια, στην παγκόσμια πολιτική και στο εμπόριο. Η διατρατική σχέση έχει ζωτική σημασία και για εμάς και για τους Αμερικανούς. Δεν αναζητούμε σύγκρουση με τους Αμερικανούς εταίρους, αλλά μια λύση. Εν τω μεταξύ θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας με έναν τρόπο συμβατό με τον ΠΟΕ και αναμένω και τις ερωτήσεις σας γιατί αυτός ήταν ο στόχος αυτής της ε, συνάντησης και, αναμέν, και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, πολύ Ζαν Λόκ για την ε, παρουσίασή σου. Να δώσω τώρα το λόγο στο Γενικό Διευθυντή της Aerofair, τον Άξελ Έτναρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε και κύριοι, είναι τιμή για μένα να είμαι προσκεκλημένο εδώ για να συζητήσω ε, μαζί σας ε, τον, ε, την απειλή του 232 για τον τομέα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και για τον τομέα του χάλιβα και νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω και εκ μέρου των συναδέλφων του τομέα του αλουμινίου. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σαφήνεια των όσων μας είπε. Τα τελευταία χρόνια ο ευρωπαϊκός τομέας χάλιβα αντιμετωπίζει πολλές σοβαρές καταστάσεις που διακυβεύουν και τη βιωσιμότητα του τομέα. Η χρηματοοικονομική κρίση το 2009, η κράση της Ευρωζώνης το 2011, ε, κινέζικα προϊόντα χάλιβα τα οποία εισραίουν στις αγορές ε, το 2015 και 2016. 95.000 ε, εργαζόμενοι στον τομέα του χάλαβα έχασαν τις θέσεις εργασίας τους ε, από το 2009. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του δυναμικού της, του τομέα του χάλιβα. Ε, η σταδιακή ανάκαμψη στη ζήτηση του Χάλαβα το 2015 και το 2016 ήταν προ όφελο μόνο των εισαγωγεών και όχι των ε, κατασκευαστών Χάλιβα. Και παρόλα αυτά, χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αποφασιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου για να καταπολεμήσει το ντάμπινγκ στο χάλιβα και να αντιμετωπίσει και την υπερβολική δυνατότητα παραγωγή, σταμάτησε αυτή η τάση το 2017. Για πρώτη φορά σε πέντε χρόνια, οι επιχειρήσει μα μπορούν να έχουν βιώσιμο ε, περιθώριο κέρδου ε, τη τάξη του 6%. Ένα ποσοστό το οποίο καθορίστηκε από την ε, εξυγχρονισμό των μηχανισμάτων των συστημάτων εμπορίου άμυνα πέρσι, αλλά φυσικά ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη. Χρειαζόμαστε συστημική ανάκαμψη ε, στα επόμενα χρόνια για να μπορέσουν οι κατασκευαστές χάλιβα να επενδύσουν σε εγκαταστάσεις, σε προγράμματα έρευνας και ε, ανάπτυξης, ψηφιοποίηση και ανάπτυξη τεχνολογιών για την ε, μείωση της χρήσης άνθρακα και για τη μελλοντική βιομηχανία στην Ευρώπη. Και πάλι η ανάκαμψη λοιπόν διακυβεύεται με την, ε, ε, ε, ο χάλιβα που αναμένεται να εφαρμοστεί αυτή την Παρασκευή. Ε, από τα όσα έγιναν και ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, είπε ότι τα μέτρα θα ισχύσουν για πολύ καιρό. Οι εξαγωγέ χάλιβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις Ηνωμένε Πολιτείε ήταν κύκλου εργασιών 6,5 δις ευρώ. Εκτιμούμε ότι 25% δασμοί μπορεί να εξαιρέσουν τουλάχιστον το 50%, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια τόνους εξαγωγών προς την ε, ε, αμερικανική αγορά. Οι συνολικές εισαγωγές ήταν 25 εκατομμύρια τόνοι το 2017, 26 εκατομμύρια τόνους αν λάβουμε υπόψη και τις χώρες ναύτα, τον Καναδά και το Μεξικό, όπως πρότεινε ε, ο πρόεδρος Τραμπ. Ε, προτείνουμε ότι τουλάχιστον το μισό του του ογκού, 13 εκατομμύρια τόνοι, μπορούν να εξαιρεθούν από την Αμερικανική αγορά και να πάνε σε άλλες αγορές και κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια μεγάλη ανοιχτή αγορά οι μεγάλοι εξαγωγή προς τις Ηνωμένε Πολιτείε θα ανακατευθύνουν τι εξαγωγέ του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ήδη ιδιαίτερα δραστήριοι. Για παράδειγμα, η Νότια Κορία, Κορέα, η Τουρκία, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Βραζιλία, η Κίνα, η Ρωσία και η Ουκρανία η απώλεια των ε, εξαγωγών προς τις ΗΠΑ Πολιτείες ε, σε συνδυασμό με τις επιπλέον εισαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποχρεώσουν τους κατασκευαστές να μειώσουν την παραγωγή κατά 2 δισεκατομμύρια τόνους και να ε, τεθούν εν κινδύνο και οι ε, θέσεις εργασίας των εργαζομένων στον τομέα του Χάλιβα χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας, έκλεισαν εγκαταστάσεις μέχρι τα τελευταία δύο χρόνια και η Eurofair υποστηρίζει πλήρως ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ε, υποστηρίζει όλες τις νόμιμες μεθόδους για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή. Οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ήταν ιδιαίτερα ανοιχτέ και του τελευταίου μήνε συζήτησαν μαζί μα με τον τομέα του Χάλιβα όλε τι εναλλακτικέ λύσει και αντάλλαξαν στοιχεία για να μπορέσουμε να δράσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και μάλιστα και όσο το δυνατόν πιο δραστικά. Παρ' όλα αυτά κάνουμε έκκληση πρώτον προς τις Ηνωμένε Πολιτείες για να αποφύγουμε οποιαδήποτε κλιμάκωση. Δεν είναι προς το συμφέρον κανονής να ξεκινήσει εμπορικός πόλεμος. Αυτό που είναι ζωτική σημασία για το δικό μας τον κλάδο, αμέσως να ελέγξουμε όλες τα προϊόντα χάλιβα τα οποία καλύπτονται από τις ε, δασμούς για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον κλάδο και τους εργαζομένους μας. Χρειαζόμαστε προσωρινή να μέτρα διασφάλισης, τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, εντός τεσσάρων εβδομάδων ή δυνατόν. Αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε ποσοστάσεις, να καλύπτουν το ευρύτερο φάσμα προϊόντων για να αποφύγουμε επιπλέον προβλήματα σε εισαγωγέ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης θα πρέπει να συνεχίσουμε να ζητάμε πλήρη εξαίρεση Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους δασμούς. Και φυσικά ε, είναι ε, πολλά υποσχόμενο το γεγονός ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο της εξαίρεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πέλη αναμένουμε να εκτραπούν 11 εκατομμύρια τόνοι χάλιβα και κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε επίπεδο εισαγωγών τα τελευταία χρόνια θα μπορέσει να παραμείνει ανοιχτά η αγορά ε, για ε, εισαγωγές στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Για να είμαι σαφής, εμείς δεν θέλουμε να κλείσει η αγορά χάλιβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πέραν των συγκεκριμένων όγκων χρειαζόμαστε ένα δασμό το οποίο να έχει αναστηλτικό αποτέλεσμα. Ε, το 2016-2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μακράν η μεγαλύτερη αγορά εισαγωγών χάλιβα στον κόσμο. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν επιπλέον εισαγωγές και επιπλέον ε, εκτροπές. Ε, βλέπουμε τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης του Τραμπ ήδη τους πρώτους δύο μήνες του έτους. Ε, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 12% ακόμα πάνω από τα ιστορικά υψηλά του 2017. Η αύξηση είναι πάνω του 65% αύξησης που είχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Μισό λεπτάκι ακόμα κύριε Πρόεδρε. Για κάποια προϊόντα ε, έχει υπάρξει αύξηση των εισαγωγών μέχρι και 75% το πρώτο αυτό δίμηνο του έτους. Ζητάμε λοιπόν από του αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα συναντηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Παρασκευή και την Πέμπτη να θέσουν το θέμα υψηλά στην προτεραιότητά τους, ε, να υπάρξει μια στεναρή αποφασιστική απάντηση για να προστατεύσουμε τον τομέα χάλιβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που έχει πάρα πολλές ε, χιλιάδες θέσεις εργασίας και πάρα πολλές έμεσες θέσεις εργασίας. Και θέλουμε οι κυβερνήσεις να δράσουν αποφασιστικά για να ε, αντιμετωπίσουν τα αίτια της παγκόσμιας δυνατότητας παραγωγής και να ληφθούν μέτρα παγκοσμίω όπως προσπαθεί να κάνει το Παγκόσμιο Φόρουμ για το Χάλιβα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή Ευχαριστούμε και τώρα από την Industry All, ο κύριος Τριάγκλη. Ευχαριστώ, είμαι ο Λεπ Τριάγκλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τους εργαζομένους, τις περισσότερου τομείς που κατασκευάζουν προϊόντα, μεταξύ των οποίων χαλιβουργία και αλουμίνιο. Να δείτε τον ιστότοπό μα σας προσκαλώ, να δείτε τι έχουμε δημοσιεύσει ως τώρα για το θέμα. Για μένα ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό το μέτρο, η πρωτοβουλία και η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ που έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ έχει και ενέχει τον κίνδυνο να επηρεάσει θέσεις εργασίας και εργαζόμενων στην Ευρώπη. Στο παρελθόν δεν ήταν πάντοτε απλό για τη χαλιβουργία <clears throat> να διοργανώσει όλε τι συνδικαλιστικέ οργανώσει τη χαλιβουργία στο ίδιο μέτωπο. Όμω τώρα είμαστε συνασπισμένοι. Καταδικάζουμε λοιπόν όλοι μαζί οι συνδικαλιστικέ οργανώσει και χαλιβουργία, ε, χαλιβουργίες, εταιρείες χαλιβουργίας σε όλη την Ευρώπη τις αποφάσεις του κυρίου Τραμπ και των ΗΠΑ. Από την άλλη, είναι επίσης σαφές ότι και εμείς ως συνδικαλιστές συνειδητοποιούμε ότι το εμπόριο είναι σημαντικό για να υπάρξει ανάπτυξη και θέση εργασία. Το ελεύθερο όμω εμπόριο πρέπει να είναι και δίκαιο. Οι δασμοί αυτοί θα το επηρεάσουν, θα το ζημιώσουν και θα δημιουργήσουν αθέμητο ανταγωνισμό στο μέλλον. Επίση, εδώ έχουμε να κάνουμε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίο δεν ε, προχωρά στι πολιτικέ αποφάσει, στην πολιτική πορεία βάσει των όσων γνωρίζουμε από τη μέχρι τώρα εμπειρία μα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να επανασταθμίσουμε τις πρωτοβουλίες του, να τις αναχαιτήσουμε από την ευρωπαϊκή πλευρά. Και αυτό έχει σχέση και με την δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρέπει να αντιδράσουμε και όχι να είναι υποτονική αντίδρασή μας. Συμφωνώ λοιπόν με την προηγούμενη σας δήλωση. Και να θυμίσω ότι είμαστε σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς ε, ομολόγους και συναδελφούς, διότι θα δείτε ότι όταν υπέγραψε την αποφασή του ο κύριος Τραμπ, περιστοιχιζόταν από εργαζομένους της εταιρείας της Χαλιβουργίας ε, της Αμερικής, οι οποίοι σε μεγάλο μέρο ήταν και μέλο τη ε, Αμερικανική Ομοσπονδία Εργαζομένων τη Χαλιβουργία. Είμαστε σε επαφέ λοιπόν μαζί του και είναι νομίζω σαφέ σε όλου μα εδώ από την ευρωπαϊκή πλευρά ότι πρέπει να εξηγήσουμε στου Αμερικανού ομολόγου μα ότι ε, αποφάσισε ο πρόεδρο Τραμπ είναι επιζήμιο και για του εργαζομένου τη Χαλιβουργία, αλλά όχι μόνο στη Χαλιβουργία και γενικότερα σε εταιρείε παραγωγή προϊόντων. Θα γίνει ο Χάλιβα πιο ακριβώ δεν θα σα πω τώρα τι λεπτομέρειες ε, λόγω χρόνου, πίεσης χρόνου, αλλά πολλά προϊόντα στις ΗΠΑ κατασκευάζονται με ευρωπαϊκό χάλιβα. Αυτό λοιπόν θα είναι επιζήμιο. Εδώ έχουμε ένα ρόλο να αντιδραματίσουμε και το αντιδραματίζουμε ήδη προσπαθώντα να πείσουμε του Αμερικανούς ομολόγου μα για τι δυσκολίε, για τι αρνητικέ συνέπειες που θα υπάρξουν στο τέλο τη διαδικασία για τις θέσει εργασία και τι εταιρείε του. Συνοψίζοντα, λοιπόν, υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ε, βρεθούν μέτρα ε, απάντησης, αλλά δεν θέλουμε να υπάρξει κλιμάκωση κάποιου εμπορικού πολέμου. Αυτό δυστυχώς ε, μας κάνει να συνειδητοποιούμε ότι απέναντί μας στην Ουάσιγκτον έχουμε να κάνουμε με κάποιον ο οποίο καταλαβαίνει μόνο τη δράση, την αντίδραση και τα αντίπεινα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τα μέτρα επαναστάθμιση τη όλη ε, κατάσταση, αλλά να είναι αναλογικέ οι αντιδράσει μα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε να καταλάβουν ότι η Ευρώπη χρειάζονται εξαίρεση στου δασμού. Για πολλού λόγου που αναφέρθηκαν και προηγουμένω. Αλλά ακόμη και αν και υπ' αυτήν την έννοια θα συμφωνήσω με αυτό που είπε προηγουμένω ο Άξελ. Ακόμη και αν υπάρξει εξαίρεση, θα πρέπει να σκεφτούμε τα μέτρα διαφύλαξη μέτρα διασφαλιστικά, διότι θα υπάρξει πλεόνασμα και μάλιστα ακόμη μεγαλύτερο πλεόνασμα στην αγορά του χάλιβα. Αυτό θα δημιουργήσει dumping στην ευρωπαϊκή αγορά, διότι δεν θα μπορεί πλέον να πάει αυτό ο χάλιβα στην αμερικανική. Άρα χρειαζόμαστε μέτρα διασφαλιστικά. Όμω Πρέπει να είμαστε και σαφεί και ξεκάθαροι, να γνωρίζουμε τι εννοούμε με τα διασφαλιστικά μέτρα και τι συνέπειε μπορεί να υπάρχουν σε ορισμένε χώρε. Τέτοιου είδου μέτρα μπορεί να οδηγήσουν και σε πρόσμενε συνέπειε στι ε, πληγήσει χώρε. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι ε, η πρόθεσή μα. Ναι, λοιπόν, μέτρα διασφάλιση, αλλά να είναι πολύ καλά υπολογισμένα, να τα σκεφτούμε, να τα μελετήσουμε και να είμαστε και εδώ αναλογικοί ε, στο μέτρο δηλαδή του λογικού στις αντιδράσεις μας για να αποφύγουμε έναν διεθνή εμπορικό πόλεμο. Αυτή είναι η δική μας συνεισφορά από την πλευρά των εργαζομένων στις εταιρείες Χαλιμπουργίας. Ευχαριστούμε πολύ, Λουκ. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να καλωσορίσω τον Υφυπουργό Οικονομικών του Μεξικού. Καλώς ήρθατε. Emma, you are the first. Έμα, έχετε τον λόγο. Μάλιστα. Ωραιότατα. Α, συγγνώμη, για δύο λεπτά, ε. Για να το, το ξέρουν όλοι. Μη φοβάστε, μη φοβάστε. Καλώς ορίζω το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει το τι κάνει για να καταπολεμήσει την πλεονάζουσα παραγωγική δυνατότητα και βεβαίως υποφέρουμε και εμείς ε, όπως και η ΕΠΑ και αναλαμβάνουμε δράση από κοινού. Και χαίρομαι που η κυρία Μάνστρομ συζητάει με τον Γουλμπερ για να ζητήσει μια εξαίρεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Έχουμε, μια... Έχουμε μέτρα επιτήρησης των εισαγωγών χάλιβα. Ποια είναι τα σχέδιά σας ε, και πώς θα λυθεί η απόφαση για να ληφθούν ανάλογα μέτρα και για το αλουμίνιο και ποιες διευκρινήσεις έχετε λάβει για την διαδικασία για να ζητήσει μια ευρωπαϊκή εταιρεία εξαιρέσεις και επιπλέον η Κομισιόν έχει σκεφτεί πως οι εξαιρέσεις σε κάποια προϊόντα ίσως έχουν αρνητικές ε, συνέπειες ε, στο εμπόριο χάλιβα και αλουμινίου στην εσωτερική αγορά και το άλλο μου ερώτημα είναι ποιε αγορέ ε, θα επηρεαστούν από την αλλαγή των ονών του εμπορίου. Ευχαριστούμε Μαρία Αρενά. Μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση σε σχέση με τα διασφαλιστικά μέτρα και το τι έχει σχεδιαστεί ως τώρα. Ακούσαμε τους κοινωνικούς εταίρους μας και τους ενδιαφερομένους και είπαν ότι πρέπει να πάνε τα πράγματα γρήγορα, να δούμε εάν έχουν ξεκινήσει σε σχετικές ε, έρευνες για ασφαλιστικά μέτρα και εσείς ήθελα να μας πείτε τι χρόνο ότι θα χρειαστούν λίγο πολύ αυτές οι, ε, λήψη αυτών των μέτρων. Επίσης ένα συγκεκριμένο προϊόν, τα rebars, όπως ε, λέγονται, δυσκολεύτηκα να βρω την μετάφραση μέχρι και στα γαλλικά. Δεν αναφέρονται στον κατάλογο που ε, μας δώσατε εσείς Όμω, ε, επειδή τα είπατε και μιλήσατε για στρέβλωση του ανταγωνισμού, υπάρχουν χώρε όπω η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία που έχουν ήδη πληγεί από αυτή τη στρέβλωση. Πώ μπορούμε λοιπόν να ε, προσθέσουμε τέτοια προϊόντα στον κατάλογο εφόσον δεν έχουν ακόμη καλυφθεί και ποια είναι η διαδικασία για να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ακόμα και οι φίλοι που είναι υπέρ του ελευθερου μπορούν να κάνουν λάθη. Ε, η μόνη φορά που ξέρω ότι έχει γίνει ποτέ τέτοια εξαίρεση για λόγους εθνικής ασφαλείας ήταν η Σουηδία δεκαετία του 70 ε, για τα άρβιλα λέγοντας ότι δεν μπορούν να πάνε ξυπόλοιτοι οι στρατιώτες μας αλλά γελιοποιηθήκαμε και σε ένα χρόνο τα αποσύραμε ελπίζω το ίδιο να γίνει και τώρα και υποφέρω και ε, βεβαίως Συμπάσχω με τους ε, φίλους ε, του κλάδου, αλλά πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο μάλλον θέλουμε να αποφύγουμε και ελπίζω να συμφωνούμε εδώ. Πρώτον, κλιμάκωση και δεύτερον βεβαίως ε, έχουμε μια υπονόμευση των κανόνων του εμπορίου. Αλλά και πέρα δεν έχω πιστεί από την Κομισιόν. Όσον αφορά λοιπόν τα αντίπεινα και τις σχετικές διατάξεις για δασμούς. Ποιο λάθος κάναμε το 2002, γιατί τότε περιμέναμε την απόφαση του πάνελ. Τώρα ε, το ίδιο σκέφτεστε, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ ε, μάλλον θεωρεί ότι έχει να κάνει με παιδιά. Και εγώ ως πατέρας ξέρω ότι πάντα πρέπει να είσαι διατηρημένο να κλιμακώσεις. αν ε, κλιμακώσει και αυτός με τη σειρά του, τι κάνουμε. Θα έχουμε 2.000 ήδη ε, δασμών. Δεύτερον, ε, για, τις, ε, για την διασφάλιση της αγοράς δεν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε μια αύξηση των εισαγωγών. Το να το κάνουμε προληπτικά θα έχουμε άλλη σύγκρουση με τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, δεν θέλω να έχουμε είπα εναντίον Ευρωπαϊκή Ένωσης και Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον Βραζιλία, Κορέα κτλ. Τρίτον, δεν μου αρέσουν οι διαπραγματεύσει. Δεν έχω πρόβλημα με τη Σεσίλια, αλλά το πρόβλημα μου είναι ότι είμαστε τώρα στην Ουάσιγκτον γιατί αυτό θέλει θέλει να έρθουν όλοι στην Ουάσιγκτον και να ζητιανεύουν επί ποινή απόσυρσης από την λίστα αυτή. Και όταν το κάνει αυτό, θα το κάνει ε, παραβαίνοντας ε, τις συμβάσεις του ΠΟΕ. Γιατί τότε ξεχνάμε το μάλλον ευνόμενο κράτος και την ίση μεταχείριση. Και νομίζω ότι βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσουν αυτοί οι δασμοί, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μπορούμε να είμαστε λοιπόν λίγο ψύχρεμοι. Ευχαριστώ. Μα πάντα, πάντα. Καρολίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, αυτές οι εξαιρεσει που θέλει να διαπραγματευτεί η Σισίλια Μάνστρομ είναι θετικές, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοια και υπάρχει ένα πιο μακροπρόθεσμο πρόβλημα. Και ακούω τώρα ότι δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Αυστραλία και άλλες χώρες. Επικίνδυνο λοιπόν το παιχνίδι, οπότε Ποιο είναι το θέμα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την υπερβολική παραγωγική δυνατότητα και τα φθηνά προϊόντα. Το γνωρίζουμε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες και να έχουμε ένα εμπόριο που θα βασίζεται σε κανόνες και θα είναι δίκαιο. Το ερώτημά μου βεβαίως είναι εάν τώρα ε, κάνει αυτές τις διαπραγματεύσεις η Σεσίλια Μάνστρομ ε, μπορεί να κάνει και τις παραχωρήσεις που πιθανόν θα απαιτηθούν και τι μορφή θα έχουν αυτές και το ερώτημα είναι ξέρετε ε, το, το αν δώσουμε θάρρος ε, στον Τραμπ ε, τι θα ακολουθήσει είναι ένας αναξιόπιστος τέρος θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ποια είναι η καλύτερη λύση όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά συνολικά να βρούμε μια καλή ε, λύση για να λειτουργούμε όλοι με βάση κάποιους κανόνες. Μάλιστα, ωραιότατα. Κυρία Λοκοσιένσκα. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι βεβαίως ελπίζουμε η Σεσίλια Μανστρομ να τα καταφέρει να επιτύχει μια λύση με τις ΗΠΑ, αλλά μιλάει με τον Τραμπ, οπότε δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Η απόφαση των ΗΠΑ ε, γνωρίζουμε ότι εξετάζεται αυτήν την στιγμή από την Κομισιόν για να μειώσουμε ακριβώς τους δασμούς και όπως είπε ο Γενικός Διευθυντής στην περίπτωση αυτών των προϊόντων ε, θα πρέπει ίσως να υπάρχουν κάποια αντισταθμιστικά μέτρα και σε έναν από τους καταλόγους μιλάμε για καλλιντικά make-up ε, για το πρόσωπο ε, make-up γενικώ. Ε, προφανώς αυτό επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες. Μιλάμε και για άλλα προϊόντα καθημερινής χρήσης στην Ευρώπη και στη χώρα μου, στην Πολωνία. Οπότε θα ήθελα να γνωρίζω από τον Γενικό Διευθυντή πώς ε, θα επιβάλλετε αντίμετρα για τον χάλιβα τα οποία θα είναι καλλιτικά. Γιατί στον τομέα του χάλιβα και του αλουμινίου γνωρίζουμε ότι το κόστος θα είναι τεράστιο. Αλλά γιατί επιλέξατε αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα. Ε, στον κατάλογο που ίσως καλύπτονται από κάποιους περιορισμούς ε, ή αντισταθμιστικά μέτρα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω ότι ε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι για εξαίρεση για την βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι λύση και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχετε συγκαλέσει το φόρουμ Χάλιβα των G20 για να υπάρξει μια συνεννόηση και με τους άλλους εξαγωγείς ε, Χάλιβα από τις ε, χώρες αυτές ε, και βεβαίω, και σε σχέση και με τον ΠΟΕ για να υπάρξει μια γενική λύση. Συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι το θέμα είναι υπερβολικής ε, παραγωγικής ε, δυνατότητας, όχι μόνο τη συγκεκριμένη σύγκρουση ε, με την ανακοίνωση του Πρόεδρου. Και εδώ πέρα νομίζω πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και στην Κίνα υπάρχει μείωση της παραγωγής το τελευταίο 1,5 έτος και θα επηρεαστούν 5, 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ε, οπότε το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα εάν λάβετε κάποια μέτρα διασφάλισης θα περιλάβετε και προϊόντα τα οποία δεν προβλέπονται μέχρι στιγμής όπως ε, ο τους ε, του σκυροδέματος και ένας εκπρόσωπος της Eurofair ήδη μας είπε το τι σημαίνει αυτό για τους ε, παραγωγούς ε, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπεύετε να περιλάβετε όλα τα προϊόντα χάλιβα και αλουμινίου. Κύριε Σίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σκίκου. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι συνέπειες ε, σε οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο, άμεσες και έμεσες για την Ευρώπη, που μπορεί να προκύψουν από το κλείσιμο της αγοράς του χάλιβας της Αμερικής και κυρίως επειδή ε, θα αλλάξουν οι εξαγωγές ε, χάλιβα από χώρες όπως η Τουρκία, η Ινδία, η Νότια Κορέα ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω ότι αναφερόμαστε σε 40 εκατομμύρια τόνους που φτάνουν σήμερα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά αυτή την κατάσταση λοιπόν θα είμαι πάρα πολύ λακωνικός. νομίζω ότι όπως πολύ σωστά ε, μας είπε ο Γενικός Διευθυντής είναι σαφές ότι σε περίπτωση που υπάρξει κλείσιμο της αγοράς θα πρέπει αμέσως να ε, ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα προφύλαξης. Και το θέμα είναι τι περιλαμβάνει αυτό το μέτρο προφύλαξης. Εμείς θεωρούμε ότι ε, για να προφυλάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρξει και έρευνα από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου για τα διάφορα προϊόντα χάλιβα. Και επομένως θα πρέπει να καλύπτει όλα τα προϊόντα τα οποία ε, αφορούν την ε, διάταξη των ΗΠΑ 232 και όχι απλώς ε, να γίνει μια προεπιλογή. Δηλαδή, αν κάνουμε προεπιλογή και υποδείξουμε ποια προϊόντα ίσως θεωρούμε ότι θα πρέπει να προφυλάξουμε, κάνουμε, διαπράττουμε ένα στρατηγικό σφάλμα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε το σύνολο του συστήματος του χάλιβα της Ευρώπης, γιατί αλλιώς τα στοιχεία είναι πολύ απογοητευτικά. Μπορεί να φτάσουμε σε απώλεια τουλάχιστον 20.000 υπαλλήλων και 140 έμεσων θέσεων εργασίας. Είναι δηλαδή πλήγμα για το σύστημα της απασχόλησης του συγκεκριμένου κλάδου. Η Τιτσιάνα Μπεγκίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με τα όσα είπε μόλις τώρα ο συνάδελφος Τσίκου. Ε, προφανώς ε, η ανησυχία για μας ε, δεδομένων και των πρόσφατων υποθέσεων με την Κίνα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά θα ήθελα να ζητήσω και κάτι ακόμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα είναι σωστή η παρατήρηση για την υπερβολική δυνατότητα παραγωγή και όλα αυτά. Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια οι Ηνωμένε Πολιτείε κάλυπταν μόνο κατά 80% και πολύ συχνά και νωρίτερα τι ανάγκε του με την προσωπική του παραγωγή. Ε, Μήπω λοιπόν ελοχεύει και κάτι άλλο πίσω από όλα αυτά τα μέτρα ε, του Τραμπ. Και τι θα μπορούσε να αποκομίσει, τι θέλει να αποκομίσει από την Ευρώπη. Ε, ακούγονται διάφορες υποθέσεις, μεγαλύτερες θεσμεύσεις των κρατών ε, για ε, χρηματική συμβολή στο ΝΑΤΟ. Βέβαια δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, αλλά και ένα από τα αιτήματα των Αμερικανών μπορεί να είναι και επιβράδυνση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων και πολύ άλλο. Γνωρίζουμε όλη την ιστορία για τις ορμόνες, η οποία είναι ευρέω γνωστή. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχετε κάποια περισσότερα νέα που να θεμελιώνουν όλες αυτές τις υποθέσεις επίσης ε, ποιες δεσμεύσεις ή μπορεί να μας ζητήσουν ε, ε, και αν θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί να αναλάβει επίσημη δέσμευση να μην υπαναχωρήσει για τις προτεγραφές μας και να μην υπάρξει τουλάχιστον μια εμπορική ρήξη την οποία δεν επιθυμεί κανείς από εμά. Η κυρία Μινέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Ντεματή. Ακούμε ότι οι επιχειρήσεις ε, δεν έχουν ανάγκη αυτά τα αντισταθμιστικά μέτρα και δε ότι δεν ε, χρησιμεύουν σε τίποτα. Και μας λέτε τώρα ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσετε αν υπάρξουν σοβαρά παράπονα. Και μετά ακούμε ότι ε, προσπαθείτε να εξασφαλίσετε μια εξαίρεση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει επιλογή να αφήσετε τι χώρε να κάνουν διμερεί ε, συμφωνίε. Παραδείγματο χάρη η Ολλανδία έχει πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα και μιλάμε για πάρα πολλέ θέσει εργασία. Γιατί είστε κατά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως την Επίτροπο Μάλστρομ για τη δέσμευσή της ε, για την όλη αυτή υπόθεση. Είναι απόλυτα σαφέ και από τη σημερινή συζήτηση ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να ε, καθυστερήσει να αναλάβει δράση. Νομίζω ότι ακούσαμε σαφέστατα από τον κλάδο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει την αναζήτηση για νέες εισαγωγές από τρίτες χώρες που δεν θα μπορούν πλέον να εξάγουν προς την ε, στι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε αυτή την πρόσβαση και θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα προφύλαξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να καλύπτει όλη το φάσμα των προϊόντων που καλύπτονται από του Ευρωπα... Αμερικανικού δασμού και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι εισαγωγέ ε, τα τελευταία χρόνια και να βασίζονται σε ποσοστώσει. Αυτό θα επιτρέψει να παραμείνει ανοιχτή η ευρωπαϊκή αγορά, αλλά να μειώσει αποτελεσματικά τι εισαγωγέ. Και έτσι θα πρέπει να αποφύγουμε και κερδοσκοπίε και να μην υπερβούν τι ποσοστώσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα πρέπει να λάβει αντισταθμιτικά μέτρα για όλα τα προϊόντα ένα προς ένα, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί υπερβολική ποσότητα κάποιου προϊόντος στις ευρωπαϊκές αγορές. Και συμφωνώ και με κάποιους από τους προλαλήσαντες ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει τα αίτια του προβλήματος. Χώρες όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ιράν, η Ινδία συνεχίζουν να αυξάνουν τους όγκους παραγωγής τους και στρεβλώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την παγκόσμια αγορά. Οι παραγωγοί τους ε, δεν έχουν συνθήκες αγορές ε, για πρόσβαση σε κεφάλαια ε, ή θέματα όπως η απασχόληση και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος λοιπόν να επιτύχουμε αυτά τα στόχους είναι να συνεργαστούν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Πολιτείε αντί να ξεκινήσει ένας ε, δαπανηρός πρόλεμος ο οποίο δεν θα οδηγήσει πουθενά. Ευχαριστώ πολύ η Μακουλάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη από το Γενικό Διευθυντή διότι δεν μπόρεσα να είμαι εδώ από την αρχή της ε, συζήτησης. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Εγώ ξέρω ότι οι στρατηγικές δεν περιγράφονται, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δρά με ευφυΐα, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπάθησε να διαβιβάσει την πιθανότητα ε, κυρώσεων. Προσπάθησε όμως να επηρεάσει λίγο τα πράγματα για να αποφύγει εμπορικό πόλεμο. Και νομίζω ότι ο κατάλογος των προϊόντων που παρουσιάστηκε δεν είναι τυχαίο που περιλαμβάνει ευαίσθητα προϊόντα για τις Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής ε, και υπάρχει πρωταγωνιστικός ρόλος ε, στο Κογκρέσο και στη Γερουσία και νομίζω ότι είναι στρατηγική επιλογή και τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω αποκομίσει. Αυτό που φοβάμαι όμως εγώ από τον Τραμπ είναι ότι ε, δεν υφέρουν οικονομικοί λόγοι, υπάρχουν πολιτικοί λόγοι για τους οποίους γίνεται όλο αυτό, διότι δεν είναι τυχαίο ότι μόλις έγιναν εκλογές στο Πίτσπουργκ που είναι η πρωτεύουσα του Χάλιβα των Ηνωμένων Πολιτειών όπου κέρδισε ο Τραμπ ε, το 2016 με 10 μονάδες διαφορά και τώρα κέρδισαν οι δημοκρατικοί με μικρό περιθώριο αλλά κέρδισαν οι δημοκρατικοί και ε, ανέστρεψαν φυσικά ε, το ποσοστό στην πρωτεύουσα του Χάλιβα. Και ο Τραμπ φυσικά ε, θέλει να αντιμετωπίσει αυτό λαμβάνοντα υπόψη και τι εκλογές του Νοεμβρίου και προσπαθεί να βρει ένα στοιχείο το οποίο να είναι προ όφελό του και φυσικά ε, θέλει να βοηθήσουμε να ε, καταπολεμήσουμε το πρόβλημα της υπερβολικής παραγωγής. Θα ήθελα να συμφωνήσω, να δω αν συμφωνείτε εσείς και να μου πείτε αν θεωρείτε εσείς ε, ότι υπάρχει κάποιο όριο στον Τραμπ, διότι δεν θα τελειώσουν οι εκλογές τον Νοέμβριο το 2018, μετά θα υπάρχουν οι προεδρικές εκλογές ε, και ε, πάντα θα υπάρχει κάποιος στρατηγικός στόχος εκλογικός, στον οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον προστατευτισμό ως στοιχείο για να κερδίσει εκεί όπου απειλείται από τα εκλογικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν ε, θα μπορούσε να ενταχθεί όλο αυτό στο σκεπτικό σα και σε αυτή την περίπτωση πώς μπορούμε να έχουμε μια πολιτική στρατηγική που να πηγαίνει εντελώ αντίθετα προς τους κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Από πλευρά μου και τρεις διευκρινιστικές ερωτήσει. Δεν είναι πολύ σαφέ ποιε γραμμέ και ποια προϊόντα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο για τα μέτρα προστασία. Περιλαμβάνονται οι σωλήνες, οι ρόδες. Ποια πράγματα θα καλύπτονται από τα μέτρα αντιστάθμισης. Επίσης, ο Λάιτχάουζερ υποσχέθηκε να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις για τις εξαιρέσεις. Ξέρουμε ότι το Μεξικό και ο Καναδάς και η Αυστραλία περιμένουν μπα και του δοθεί καμιά εξαίρεση από, από αυτού του δασμού. Ποια είναι τα κριτήρια, Υπάρχουν κριτήρια για τι εξαιρέσει που θα δοθούν. Και τρίτον, δεν μπορώ καν να φανταστώ τι μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη στις, ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις. Διότι δεν έχουμε επιδοτήσεις, δεν έχουμε dumping στη χαλιβουργία μας σε αυτό το μέτωπο. Τι να τους προσφέρουμε για να πείσουμε τον κύριο Τραμπ να προβλέψει εξαίρεση. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις και πολύ εύστοχες. Για το μηχανισμό παρακολούθησης στο Χάλιβα. Ναι, Λογικό θα ήταν να καλύπτει τώρα και το αλουμίνιο. Ποια θα είναι η διαδικασία για πιθανές εξαιρέσεις. Είναι εντελώς ε, και μόνον θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών, εγχώριο και εσωτερικό. Οι χρήστες στις είπα μπορούν να υποκινήσουν τη διαδικασία που δεν θα έχει όμως καμία σχέση με τους εξαγωγείς των τρίτων χωρών. Μπορεί να συνδεθεί, να συσχετιστεί, αλλά εκείνοι οι χρήστες θα πρέπει να προβάλλουν τα επιχειρήματά τους και γι' αυτό υπάρχουν τα σχετικά κριτήρια, αλλά εμείς δεν μπορούμε να εμπλακούμε απευθείας παραγωγή προϊόντων χάλιβα και αλουμινίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες τους. Είναι μια κλασική διαδικασία. Ως προς την ε, ερώτηση της κυρίας Αρενά για τα διασφαλιστικά μέτρα και το χρόνο που θα πάρει όλο αυτό, η διαδικασία για τα μέτρα διασφάλισης εντάσσεται και διέπεται από πολύ αυστηρά κριτήρια. Αυτά τα αυστηρά κριτήρια προβλέπουν για την έναρξη έρευνας. Εξεταστική διαδικασία για την κάλυψη των προϊόντων. Είναι δύο οι φάσεις της διαδικασίας. Πρώτα απ' όλα έρευνα με τη δυνατότητα λήψης προσωρινών μέτρων δεδομένου του, συνόλου, του αριθμού των συνόλου των διαδικασιών περίπου μέσα σε ένα δίμηνο και για τα οριστικά μέτρα, τα τελικά μέτρα, χρειάζεται πιο πολύς χρόνος. Πάνω από 6 μήνες θα έλεγα. Για τα προσωρινά λοιπόν μέτρα. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για αρμοδιότητα της Επιτροπής με επιτροπολογία για τα προσωρινά η Επιτροπή αποφασίζει υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ενισχυμένη πλειοψηφία που να διαφωνεί με τα προσωρινά μέτρα. Για τα ε, οριστικά, τα τελικά μέτρα πρόκειται για εξαίρεση στη διαδικασία της επιτροπολογίας ε, σε σχέση με τη λειτουργία της όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Εκεί χρειάζεται ενισχυμένη πλειοψηφία υπέρ όλων των κρατών μελών για τα τελικά μέτρα. Ως προς την κάλυψη. Το πιο απλό, εφόσον ξεκινήσει έρευνα, και το πιθανότερο ότι θα γίνει αυτό, εντός ολίγων ημερών θα είναι μεγάλη ομάδα των προϊόντων που θα καλύπτονται για να είμαστε βέβαιοι ότι διαφυλάσσουμε το σύνολο των προϊόντων, ενώ το δυνατό μεγαλύτερο σύνολο στην περίπτωση του χάλιβα και του αλουμινίου. Αυτό δεν προδικάζει την τελική μας επιλογή. Αυτή θα γίνει βάσει της κατάστασης που θα έχει διαμορφωθεί στην αγορά. Και μπορούμε να δράσουμε πολύ γρήγορα, ώστε μέσα σε ένα διάστημα σύντομο σχετικά, χάρη στα μέτρα ε, παρακολούθησης, τα μέτρα με τα οποία παρακολουθούμε, να ξέρουμε ποια είναι τα, πιο, τα προϊόντα που απειλούνται περισσότερο. Τώρα, η ίδια ερώτηση με τα καλλιντικά. Παραδόξως. Για τα μέτρα επαναστάθμισης. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την προστασία της δικής μας βιομηχανίας χάλιβα και αλουμινίου. Είναι ένας τρόπος να προστατευθούμε από τη σκοπιά του ΠΟΕ και της επίλυσης διαφορών εκεί με προϊόντα που να επανασταθμίσουν τα μέτρα που έχουν ε, λάβει οι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν είναι αντίπεινα, είναι αντίμετρα. Θα πρέπει όμως η επιλογή των προϊόντων να είναι ανάλογη με τα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει επιτακτική ανάγκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν δηλαδή να υποκατασταθούν μεταξύ τους και υπάρχει και άλλη δυνατότητα κάλυψης της προσφοράς. Στα καλλιτικά δεν είναι επιτακτική ανάγκη αμερικανικής παραγωγής ας πούμε και για τα διασφαλιστικά μέτρα βεβαίως ο πλεισμός κυροδέματος θα καλύπτεται. Αυτό που λέτε λοιπόν κυρία Αρενά είναι ο κατάλογος επαναστάθμισης. Δεν έχει καμία σχέση. Ένα τρίτο των γραμμών ε, για, το, για τους δασμούς αφορούν το χάλιβα, ένα τρίτο τους άλλους δημοκρατικού κλάδους και ένα τρίτο τα λοιπά. Τον κατάλογο λοιπόν αυτό τον καθορίσαμε βασιζόμενοι σε οικονομικά κριτήρια αλλά και πολιτικά γιατί ξέρουμε καλά την πολιτική γεωγραφία παντού στον κόσμο. Όταν υπάρχουν εκλογές σε κάποιες τρίτες χώρες δεν έχει και πολύ σημασία. Το ερώτημα του κυρίου Φιέλνερ. Πρώτον, δεν είμαστε σε φάση και δεν έχουμε πρόθεση κλιμάκωσης. Το θέμα της επαναστάθμισης. Αυτό που κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από τη σκοπιά της επίλυσης διαφορά του ΠΟΕ. Στο άρθρο 8 προβλέπονται 60 μέρες για να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό δεν καθορίζει το αν μετά από το, τη λήξη αυτού του διαστήματος θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Αν όμω τώρα δεν λάβουμε μέτρα, μετά δεν θα έχουμε κάνει τη δυνατότητα να προβλέψουμε αντίμετρα ε, και να συμμορφωνόμαστε και με τους κανόνες του ΠΟΕ. Αυτό έγινε και το 2002. Υπήρχαν διασφαλιστικά μέτρα. Δεν ήμουν τότε στην Γενική Διεύθυνση Trade, ήμουν στην Άγκρη. Δεν τα είχα παρακολουθήσει τόσο στενά, όμως αυτό που ξέρω είναι ότι τελικώς επανασταθμίσαμε το θέμα της ε, κατάργησης των παραχωρήσεων, αλλά δεν πήραμε αντίμετρα μέσα στα πλαίσια, στα πλαίσια της επαναστάθμισης, διότι η εξαίρεση που είχαμε πάρει τότε μας έφτανε. Και γρήγορα ενεργοποιήθηκαν και οι κανόνες του ΠΟΕ, οπότε ε, θα χάναμε αν είχαμε αντισταθμιστικά μέτρα διαφορετικά. Είχαν θεωρηθεί άκυρα. Τώρα, στην περίπτωση αυτή, τα διασφαλιστικά μέτρα, κατά τη δική μας την ανάλυση, είναι ότι η αγορά του χάλιβα στη ΣΥΠΑ πάνε καλά, έχουν αυξηθεί τιμές περισσότερο από κάθε άλλη αγορά. Στο παρελθόν έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια, όπως και εμείς. Και έχουν λάβει μέτρα αντι-dumping και πολύ αυστηρά αλλά η καλύτερη της εταιρεία έχει αυξήσει το κέρδος της κατά 35% το 2017 σε σχέση με το 2016. Και οι περισσότερες εξαγωγές την περίοδο μετά το 2014 ε, μειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2017 υπήρξε συνολικός μείωση, όχι για όλα τα προϊόντα, παρά την αναγγελία τον Απρίλιο του 2017. Άρα οι προϋποθέσεις για να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα δεν πληρούνται. Να επιβεβαιώσω ότι είμαστε πολύ ψύχρεμοι. Φροντίζουμε να είναι το κεφάλι μας στη θέση του και να παραμένει και στη σωστή θερμοκρασία, ώστε να μην χάνουμε τη λογική μας. Ε, για τις διαπραγματεύσεις. Συζητήσεις γίνονται για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία μηδέου ενδιαφέροντος. Ποτέ δεν διαπραγματεύομαστε η Ποτέ. Και ακόμη κι αν στο τέλος της διαδικασίας φανεί ότι υπάρχει εξαρτή, θα φανούμε πάρα πολύ συνετοί. Διότι δεν ξέρουμε εν τέλει ποια θα είναι η ε, απόφαση του ίδιου του πρόεδρου του Τραμπ. Και νομίζω ότι ό,τι λύση και αν βρεθεί, ακόμη και αν δοθεί εξαίρεση, πρέπει να υπάρξει απομάκρυνση εξάλληψη των παραχωρήσεων. Διότι αν ε, ε, εξαλειφθεί και η εξαίρεση, η παπειλή, κράτος απειλής ξαφνικά θα μπορούμε να πάρουμε αντίμετρα. Την περασμένη εβδομάδα μπορώ να σας πω ότι υπήρξε και στήριξη από τα κρατημέλη για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαστε πολύ αποφασισμένοι, θα επιδείξουμε πυγμή, θα φτάσουμε τη διαδικασία στο τέλος και αν η εξαίρεση ε, δοθεί, κάτι που δεν είναι καθόλου σίγουρο, Αυτό θα έχει σχέση με την αποφασιστική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σας το είπα, ε, δεν ε, σταμάτησα να εργάζομαι για το θέμα. Συνάντησα πολλούς ε, και βουλευτές και άλλους ενδιαφερομένους και από παντού υπάρχει διάθεση να βρεθεί μια λύση με τη διαδικασία αντιστάθμισης και να βρούμε μία ε, λογική λύση μακροπρόθεσμα για το ε, εργατικό δυναμικό. για τον κύριο Σόλτ. Ναι, μιλάμε για υπερβολική παραγωγή, αλλά δεν χρειάζεται να ψάξουμε τη λύση της εξαίρεσης χωρίς νομιμοποίηση των μέτρων των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ. Το εξήγησα νομίζω και λεπτομεριακώς. Ναι, θέλουμε ένα σύστημα που να βασίζεται σε κανόνες. Ναι, στο G20 είμαστε πιο δραστήριοι στο φόρουμ για το Χάλιβα. Πραγματικά με τα χαράς να δεχτούμε κι άλλους εκεί. Όμως φανταστείτε ότι δεν θα λύσει τα πάντα, δεν θα λυθούν τα πάντα στο φόρουμ του Χάλιβα. Ναι, η Κίνα άρχισε και αυτή να προβλέπει μέτρα, αλλά συνεχίζεται η επιδότηση και στον τομέα του Χάλιβα και του αλουμινίου. Δεν είμαι βέβαιος ότι οι αριθμοί που αναφέρθηκαν είναι εντελώ ακριβείς. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή δεν είναι περίεργο η Κίνα, η Ινδία και άλλες, ε, κάποιες άλλες χώρες να επιδοτούν την ε, παραγωγή του χάλιβα. Το πρόβλημα με την Κίνα είναι ότι μεταξύ του 2012 και του 2016 είχαν αύξηση στην παραγωγή του χάλιβα ενώ μειωνόταν η ζήτηση. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί αυτή η αύξηση δυνατοτήτων δεν βασίστηκε μάλλον γιατί βασίστηκε σε επιδοτήσεις και δεν ακολούθησε την ε, τάση της αγοράς. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή είναι πολύ μεγαλύτερη από την εγχώρια ζήτηση και την ε, ζήτηση της εξωτερικής αγοράς. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και οπωσδήποτε θα το κάνουμε. Για την ερώτηση του κ. Σίκου, νομίζω μου σαφής ότι τα μέτρα διασφάλισης δεν θα αποκλείσουν κανένα προϊόν από την έρευνα και θα δούμε τελικά τι πρέπει να γίνει και αν υπάρξουν τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην προστασία της βιομηχανίας, αλλά με έναν τρόπο που θα ελαχιστοποιεί την ε, στρέβλωση του εμπορίου. Δεν θέλω τώρα να το πω δημοσίως, αλλά δεν αποκλείεται τίποτα. Υπάρχουν τρόποι πάντως για να μειωθεί η στρέβλωση του εμπορίου, γιατί πρέπει να αποφύγουμε ε, να, να διαδοθούν αυτά τα μέτρα σε ολόκληρο τον κόσμο και να έχουμε μια δραματική κατάσταση. Πρέπει να σκεφτούμε και το τι θα κάνουν οι άλλοι. Για την ερώτηση του κ. Μπεγκίν. Ε, για την υπερβολική παραγωγή νομίζω ότι απάντησα οπωσδήποτε δεν μπαίνουμε σε συζητήσεις και οπωσδήποτε συζητήσεις για τις προδιαγραφές των τροφίμων. Δεν θα δώσουμε ανταλλάγματα ε, στην διαπραγμάτευση και δεν υπάρχει τέτοια διαπραγμάτευση, τις προδιαγραφές ε, των τροφίμων, ε, την προστασία του καταναλωτή. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Όλα τα προϊόντα λοιπόν που μπαίνουν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα σέβονται τις προδιαγραφές των τροφίμων. Δεν τίθεται ζήτημα. Δεν, δεν είναι θέμα προσυζήτηση. Το ερώτημα της κυρίας Μελέα που μίλησε για αντίπεινα. Δεν κάνουμε αντίπεινα. Ε, έχει σημασία και η ορολογία. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί και για την δυνατότητα των κρατών μελών να προσπαθήσουν για μια μεμονωμένη εξαίρεση. Δεν ξέρω, εγώ, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι και το πιο αποτελεσματικό. Αυτοί που προσπαθούν να διχάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κερδίσουν και νομίζω όπως ξέρετε ισχύσαν τη ενώση και αυτό θα συμβεί και τώρα. Οπότε. Ναι, ναι. Και τις αγορές των ΙΠΑ πρέπει να διατηρήσουμε. Να μην γίνει εμπορικός πόλεμος. Απάντησα ήδη. Νομίζω τώρα της κυρίας Πινέιρο. Μπέντ, οι ερωτήσεις σας για τις ε, γραμμές ε, της τελωνιακής των ΙΠΑ. Θα δούμε όταν ε, θα ληφθούν τα μέτρα. Πιθανώς θα καλύπτει όλες τις γραμμές. Λαμβάνοντας υπόψη το τι θα συμβεί. Για τις κατευθυντήριες γραμμές δεν νομίζω ότι θα δούμε κατευθυντήριες γραμμές σε τελική ανάλυση. Νομίζω πως υπήρχαν κάποια στοιχεία που ανέφερε ο πρέσβης ο κύριος Σλάιτχάιζερ όταν είχαμε την τριμερή και την διμερή συζήτηση πριν από 15 μέρες ε, και νομίζω ότι ήταν ακριβώς δύσκολο να γίνουν αυτές οι συζητήσεις, δεν ήταν τόσο απλό και είχαμε ακριβώς ε, την πολύ επιτυχή τριμερή δήλωση με είπα και Ιαπωνία για συμπεριφορά που δεν συνάδει με την αγορά και για τις επιδοτήσεις, αλλά το σημαντικό ήταν η αποτελεσματικότητα των μέτρων υπεράσπισης του εμπορίου. Και βεβαίως δεν ε, υπάρχει νομίζω καμία αμφισημία στο φόρουμ του Χάλιβα, το είδατε, είναι πάρα πολύ καλό το έγγραφο, δεν ε, καλύπτει βεβαίως τα πάντα, αλλά το ξέρετε εσείς και οι συντονιστές ε, των ομάδων και ε, νομίζω μπορείτε να διαβουλευτείτε. Είναι ένα πολύ καλό έγγραφο θα έλεγα. και δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτή που ξεκίνησε αυτήν την κρίση. Και αν δούμε τα νούμερα, η ΕΠΑ τα τελευταία 10 χρόνια έχουν κόψει την παραγωγή χάλιβα κατά 10% και το μισό από αυτό τα τελευταία χρόνια οι ΕΠΑ λοιπόν έχουν μικρότερη παραγωγή αλλά έχει διατηρηθεί λίγο πολύ τα ίδια τα τελευταία χρόνια. Ε, υπήρχε βεβαίω η δραματική αύξηση της παραγωγής στην Κίνα και στο αλουμίνιο, όπω είπαμε. Και η τελευταία σας ερώτηση, αν προσφέρουμε διαπραγματεύσεις. Όχι. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε. Ποτέ δεν διαπραγματευόμαστε υπό καθεστώς απειλής. Γιατί έτσι νομοποιούμε αυτό το οποίο θεωρούμε μέτρα που δεν συμφωνούν με τους κανόνες του ΠΟΕ. Εμείς παραμένουμε πολυμερείς ε, και σεβόμαστε τις διαδικασίες του ΠΟΕ και επιπλέον έτσι, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο πλαίσιο του ΠΟΕ ε, για να έχουμε κανόνες οι κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν να υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα επίλυσης διαφορών που θα λειτουργήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Ζανλουκ για τα ξεκάθαρα λόγια σας ε, και το μήνυμά σας, ε, το οποίο το χρειαζόμασταν σήμερα. Ολοκληρώνεται λοιπόν η σημερινή μας ε, συνεδρίαση και βεβαίως το θέμα αυτό θα το δούμε και στην έκθεσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.